Καλημέρα σε όλους σας και καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής Αναφορών. Δυόμιση είχαμε προβλέψει να αρχίσουμε, αλλά δεν βλέπω εδώ αρκετό κόσμο, ούτε καν απαρτία δεν έχουμε. Ας αρχίσουμε όμως παρόλα αυτά. Πίτερ, εσύ και οι υπόλοιποι, καθίστε παρακαλώ και θα μπορέσουμε έτσι σιγά σιγά να προχωρήσουμε και να περάσουμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Προσπαθώ να κοιτάξω γύρω εδώ και να δω αν είναι εδώ στην αίθουσα αυτοί που πρέπει να πάρουν το λόγο σε λίγο. Δεν είναι όμως. Τέλος πάντων όσοι είσαστε, καθίστε. Και επιτρέψτε μου σιγά σιγά να αρχίσω να σας ενημερώνω για το σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη τα αποτελέσματα που είχαμε στη ψηφοφορία γραπτής ε, διαδικασίας για την ε, ένσταση ε, από την ημερήσια διάταξη το συντονιστών του 25 η Μαρτίου. Λοιπόν, εγκρίθηκαν αναφορές, έτσι όπως εγώ πρότεινα ως ο πρόεδρος, εκτός από τις εξής. Αναφορά 10-13 η οποία θα παραμείνει ανοιχτή. Θα σταλεί στην ΕΝΒΗ προς ενημέρωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας στείλει παραπάνω πληροφορίες. Αναφορά 10-20 και 11-15 θα παραμείνουν ανοιχτές και θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει και να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. 11-25 τώρα. Ε, δηλώθηκε ως παραδεκτή και ο αναφέρον θα πάρει τις κατάλληλες πληροφορίες και μετά θα στείλουμε την αναφορά αυτή στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για γνωμοδότηση. Και θα ζητήσουμε επίσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερες πληροφορίες. Όσον αφορά τώρα τα θέματα Β, τα αποτελέσματα από την προηγούμενη φορά είναι τα εξή. Αναφορά 60 θα παραμείνει ανοιχτή και προβλέπεται συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις αρχές της επόμενης κοινοβουλευτικής θητείας και αναφορά 224 θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να έχουν εγκριθεί τα νέα κείμενα. Επίσης κλείσαμε τις αναφορές 853, 316, 373, 1227 και 1304. Αυτά είναι τα αποτελέσματα από τη συνεδρίαση των συντονιστών. Αυτά συμφωνήθηκαν. Σημείο 4. Διάφορα. Εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι φτάνουμε στο τέλος της θητείας μας, είτε το πιστεύετε είτε όχι, και θα έχουμε όμως ε, την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε μεταξύ μας. Δικιά μου αρμοδιότητα είναι το κοκτέιλ της Επιτροπής μας, το οποίο θα λάβει η χώρα την Τετάρτη 10 του μηνός, την επόμενη Τετάρτη δηλαδή, στις 6.30 το απόγευμα. Οπότε, να είσαστε έτοιμοι για μια πολύ όμορφη συνάντηση μεταξύ μας για να ευχηθούμε ένα τον άλλον ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Πού, πού, ρωτάει κάποιος από την το πού θα σας το ανακοινώσουμε αργότερα. Ε, ψάχνω να βρω έναν όμορφο χώρο. Γι' αυτό δεν ξέρουμε ακόμα, περιμένουμε τον πρόεδρο να μας πει πού. Αλλά να ξέρετε ότι ο στόχος μου είναι το καλύτερο, ο καλύτερος χώρος για αυτό το κοκτέιλ. Πάντα το καλύτερο. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε το καλύτερο και το υψηλότερο. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πού θα γίνει τελικά αυτό το κοκτέιλ. Τώρα ήθελα να είναι εδώ η Μπεντρίς Μπεσέρα. Γιατί έχουμε την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Και δεν είναι εδώ. Ωραία. Η Μπέτρις Μπεθέρα δεν είναι εδώ, αυτό είναι ένα γεγονός. Οπότε στρέφομαι προς ε, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το θέμα. Η Ελένη Μπουλανζέρη έχει το λόγο. Ε, είσαστε εδώ. Ναι. Ωραία. Καλώς ήρθετε και σας δίνουμε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αν συμφωνείτε, Έχουμε εδώ τις επιπτώσεις της έκθεσης και την ενημέρωση όσον αφορά την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, όσον αφορά τα τελευταία δύο χρόνια, μετά το ψήφισμα δηλαδή. Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για την έκθεση επίσης της κυρίας Μπεσέρα, που είναι η συγγήτρια και να ξέρετε ότι ήταν αρκετά πλήρης. Δεν έχω βέβαια πολύ χρόνο ούτε κι εσείς για να σταθούμε επιμακρό σε αυτό. Πάντως όσον αφορά την έκθεση ηθαγένειας από το 2017 θα θυμόσαστε ότι και το Συμβούλιο είχε καταλήξει σε συμπεράσματα για την έκθεση αυτή βάσει του έργου λέει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Θα ξέρετε σίγουρα επίσης ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκπονήσει διάφορες εκθέσεις σε επίπεδο της Επιτροπής Δεγματικών Υποθέσεων για τις διατάξεις όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Θαγένεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν βασίστηκε στις εκθέσεις αυτές και ε, συμφωνεί φυσικά με το στόχο αυτό για να υπάρχει Ευρωπαϊκή Θαγένεια. Τώρα μετά τις συστάσεις της έκθεσης μετά το 2017 ε, θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία. Πρώτον, για τα δημοκρατικά δικαιώματα. Φέτος, όχι, πέρυσι, πέρυσι, το 2018, ετοιμάσαμε μια έκθεση για τις τοπικές εκλογές, για τα δικαιώματα δηλαδή ε, εκλογής σε τοπικό επίπεδο των Ευρωπαίων που μετακινούνται. Τι ισχύει για τα δικαιώματά τους, το δικαίωμα στην ενημέρωση, ποιοι περιλαμβάνονται σε αυτό το δικαίωμα, πώς θα γίνει η ψηφοφορία πιο εύκολη και πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Η δημοκρατία ήταν κάτι πολύ σημαντικό ε, πέρυσι. Είχαμε το κολόκιουμ, το συνέδριο για τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να ετοιμαστεί αυτό το συνέδριο κάναμε και μια έρευνα ε, για να συγκεντρώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες ποια είναι η άποψη των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά τα δημοκρατικά δικαιώματα, αν πιστεύουν ότι χρειάζεται βελτίωση και πού πιστεύουν ότι πρέπει να αναλυφθεί δράση. Επίσης, μετά την υπόθεση Cambridge Analytica, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέδωσε ένα πακέτο μέτρων το Σεπτέμβριο του 2018 για να διασφαλίσει ελεύθερες εκλογές ήταν ένα πακέτο που είχε να κάνει και με τα δικαιώματα αυτά, αλλά και με συστάσεις προς τις χώρες μέλη και τα πολιτικά κόμματα. Τώρα συνεργαζόμαστε με τις χώρες μέλη και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τις εκλογές, για να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, βέλτιστες πρακτικές, εν της προετοιμασία των ευρωεκλογών. Είχαμε ήδη δύο συναντήσεις στο δίκτυο αυτό και θα έχουμε μια τρίτη αυτή τη βδομάδα. Ένα από τα σημαντικά ζητήματα της έκθεσής μας ήταν η ενημέρωση των πολιτών. Έχουμε πολλές εκστρατείες ενημέρωσης και γενικές και ειδικές τέτοιες εκστρατείες σε σχέση με δικαιώματα των πολιτών. Ε, πρόσφατα είχαμε κάτι για την προστασία των καταναλωτών, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τα δικαιώματα που έχουν ε, για να προστατευθούν. Επίσης συζητάμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς θα ενημερώσουμε καλύτερα τους πολίτες για το δικαίωμά τους στην ε, άσκηση αυτή, άσκηση δηλαδή του δικαιώματος τους να συμμετέχουν στις εκλογές. Στην ίδια λογική, δημοκρατία και ενημέρωση δηλαδή, κάναμε πολλά και πέρυσι. Ένα άλλο θέμα ήταν η ισότητα και τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΕΔΟ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει οπωσδήποτε να εφαρμόσει διάφορες δράσεις για την ε, ενίσχυση της ισότητας ε, των ατόμων ΛΟΕΔ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ετοιμάσει έκθεση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί βάσει όλων αυτών των εκστρατιών ε, ενημέρωσης και πληροφόρησης. Τι άλλη εξέλιξη θα μπορούσα να σας αναφέρω. Α, ναι, την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολύ πρόσφατα, τον Ιανουάριο φέτος δηλαδή ήτανε, για την επένδυση στην ηθαγένεια. Ένα πρώτο βήμα είναι να εντοπίσουμε πώς μπορούμε να επενδύσουμε σε προγράμματα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και πώς θα πείσουμε τις χώρες μέλη να διασφαλίσουν ένα νέο πλαίσιο για την ασφάλεια, την προστασία των πολιτών. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει αυτή τη βδομάδα. Και όλα όσα κάνουμε δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας. Έχουμε τους ίδιους κανόνες διαφάνειας, δηλαδή που έχουμε πάντα. Ε, υπάρχει ημερήσια διάταξη των συναντήσεων αυτών, το, τα θέματα, το περιεχόμενο, όλα. Και κάτι ακόμα, πολύ ενδιαφέρον πρακτικά, είναι η πρόταση που εκδώσαμε για τα έγγραφα των ε, κατοίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρχει ένα έγγραφο πιο ασφαλές. Οι Ευρωπαίοι που κυκλοφορούν θα μπορούν πιο εύκολα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία και συμπεριλαμβάνεται σε αυτό και ένα έγγραφο που θα έχουν στη διάθεσή τους που θα είναι περισσότερο ασφαλές. Επίσης, μια άλλη πρόταση για ταξιδιωτικό έγγραφο. Όταν δηλαδή κάποιος χάσει το έγγραφό του, το, είτε διαβατήριο είτε ταυτότητα σε μια τρίτη χώρα να μπορεί να έχει ένα τέτοιο ταξιδιωτικό έγγραφο για να μπορεί να επιστρέψει στη χώρα του. Υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος θεμάτων πάντως. Σημαντικό είναι και το ε, Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δίνουμε πολύ σημασία στις αποφάσεις του δικαστηρίου αυτού. Υπάρχει η υπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία διεφυλικών ζευγαριών. Υπάρχει το θέμα της απώλειας της θαγένης μιας χώρας μέλους. Όταν πρόκειται για Ευρωπαίους πολίτες, το θέμα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας, όπως καταλαβαίνετε, έχει μεγάλη σημασία. Έπειτα υπάρχουν και διατάξεις της συνθήκης που λαμβάνουμε υπόψη μας. Κάθε τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει τις εξελίξεις όσον αφορά το δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Θαγένεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτή η Επιτροπή, η Επιτροπή Αναφορών, από την αρχή της κοινοβουλευτικής θητείας προσπάθησε με διάφορους τρόπους να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές, στις ευρωεκλογές με διαφορετικούς τρόπους. Η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου θα είναι μια ευκαιρία για να καταστεί η Ένωση πιο δημοκρατική και η Κομισιόν τη ζητήσαμε να μας ετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψήφου στις ευρωεκλογές και αυτό το σύστημα να διατεθεί σε όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητάμε από την Κομισιόν επίσης να δώσει συνέχεια σε παράπονα που έχουν ακουστεί για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις ε, τοπικές και αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Είναι σημαντικό να δούμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε οι οποίοι μετακινούνται για διάφορου λόγου, από ένα κρατό μέλο, σε ένα άλλο κρατό μέλο, για να παραμείνουν είτε για σπουδέ, είτε για επαγγελματικού λόγου, είτε για οικογενειακούς λόγου, θα πρέπει να διατηρήσουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα στι εθνικέ ε, εκλογέ τη χώρα προέλευσή του, που δεν είναι ε, που δεν συμβαίνει τώρα α πούμε για του Βρετανού χάνουν αυτό το δικαίωμα μετά από 15 χρόνια παραμονή στο εξωτερικό. Και αυτή η επιτροπή, η δική μας επιτροπή, έπαιξε σημαντικό ρόλο και τόνισε ε, στις ε, τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τον Brexit το πρόβλημα αυτό. Είπαμε το θέμα αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά. Η Επιτροπή μας, λοιπόν, πρέπει να αισθάνεται περήφανη τώρα στο τέλος της θητείας που τόνισε τόσο σημαντικά θέματα, τόσο ε, ενδιαφέροντα για τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στα δρόμενα, στα δημόσια δρόμενα. Λοιπόν, θέλει κάποιος να πει τίποτα? Όχι. Άρα, μπορούμε να πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, το οποίο είναι η ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαία Μεσολαβήτρια, την κυρία Έμιλι Οράιλι, ε, για τα προτινόμενα νέα προνόμια της, η οποία όμως δεν είναι εδώ. Νομίζω ότι θα έρθει όπου να είναι. Ας την περιμένουμε λιγάκι μέχρι να φτάσει. Αν κάποιο άλλο στο μεταξύ θέλει να πάρει το λόγο για να θέσει κάτι άλλο, ε, περιμένω στην κυρία Ράιλι, α του δώσουμε το λόγο. Ο Πίτερ πάντα έχει κάτι να πει, πάντα, κατα... πάντα, κατα... πάντα κάτι σκέφτεται, αλλά όχι σήμερα. Μήπω κάποιος άλλος. Πίτερ, εμπρό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ δεν θα αναφερθώ στην τελευταία έκθεση που αφορά μόνο την υπηκότητα αλλά και το θέμα των διαπραγματεύσεων του Brexit. Νομίζω ότι με πολύ αυθόρμητο τρόπο προτείναμε να γίνει αυτή η συγκεκριμένη έκθεση που αφορά και τα δικαιώματα των νέων και χαίρομαι ιδιότερα που βλέπω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δείχνουν ενδιαφέρον και δέχονται αυτές τις προτάσεις μας. Το θέμα του δικαιώματος ψήφου είναι κάτι που πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη και βεβαίως πρόκειται και για ένα σύνολο υπηρεσιών και δικαιωμάτων που δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε όπως παραδείγματο χάρη περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων, χρόνιες ασθένειες, οι λεγόμενες σοβαρές ασθένειες και νομίζω ότι το θέμα αυτό των ασθενειών, το θέμα που αφορούν, τα θέματα αυτά που αφορούν κάποιον που παραδείγματος χάνει έχει πάει σε μια άλλη χώρα, από τη Γαλλία έχει πάει στη Γερμανία και του συμβαίνει κάτι το σοβαρό, ένα σοβαρό ατύχημα. Όλη αυτή η διευθέτηση είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει και δεν είναι μόνο οι επιμέρους αναφορές αλλά γενικότερα τα δικαιώματα των νέων και το θέμα της υπηκότητας και το θέμα των νέων είναι κάτι που δεν μπορεί να αποτελέσει πρόγραμμα ή σχέδιο εθνικό μίας της μίας ή της άλλης κυβέρνησης. Είναι κάτι που αφορά όλη την Ευρώπη και θα πρέπει να υπάρξει από μας ε, συνείδηση ότι είναι θέμα ύψης της προτεραιότητας. Τώρα να καλωσορίσουμε τη φίλη και συνάδελφο, την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, κυρία Εμιλή Ράιλι, που την προσκαλέσαμε για να αντιδράσει για, πάνω στην έκθεση που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία ένα ψήφισμα για σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίζει τι τις γενικές προϋποθέσεις ε, για τις, την διεξαγωγή των ε, καθηκόντων της, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή γενικά. Έχετε το λόγο για να αντιδράσετε ε, στα όσα θέτει και όσα επιτάσσει αυτό το ψήφισμα. Καλησπέρα, Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε τον τρόπο που θα προχωρήσουμε και το γραφείο ε, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή τι θα κάνει μετά από το θέμα για το οποίο μίλησε η κυρία Βίξτρομ. Θα ήθελα πριν περάσω στην ουσία, να κάνω μια μικρή ε, αναδρομή στο παρελθόν. Τα τελευταία πέντε χρόνια το Κοινοβούλιο υποστήριξε το γραφείο μου. Ε, αντιμετωπίσαμε άριθμα παράπονα ε, και τη δουλειά που κάναμε για το Frontex, για τη διαφάνεια του Συμβουλίου, για τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων Brexit, για τις πρακτικές των ε, θεσμικών οργάνων για τον κώδικα διοντολογίας κομισιών και για την ε, επίλυση σύγκρουσης συμφερόντων. Στην ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων του Ombudsman ε, πάντα λάβαμε πλατιά στήριξη από την Ολομέλεια και στη δουλειά που κάναμε τη διαφάνεια στο Συμβούλιο υπήρχε μεγάλη συνένεση σε όλες τις πολιτικές ομάδες, σε όλο το πολιτικό φάσμα. Σας ευχαριστώ για αυτά τα μηνύματα έτσι, εμπιστοσύνης του Κοινοβουλίου και ειδικά τη Επιτροπή σα προ το πρόσωπό μου και το γραφείο μου. Είπα κατά επανάληψη ότι το γραφείο τη Διαμεσολαβήτρια είναι ισχυρό μόνο εφόσον έχει ισχυρή στήριξη. Το Φεβρουάριο το Κοινοβούλιο υιοθέτησε μία έκθεση για τον αθεωρημένο καθεστώ του Διαμεσολαβητή με στήριξη από όλε τι πλευρά. Θέλω να ευχαριστήσω ιδίω τον κύριο Ραγκέλ από το ε, ΑΦΚΟ και το ΕΛΚ και την άλλη μία εισηγήτρια για την έκθεση. Ε, εγώ δεν ήθελα αναθεώρηση του καθεστώτος μου. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, ευχαριστώ για την υποστήριξη αυτή και θεωρώ ότι το καθεστώς αυτό θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, το κείμενο θα σταλεί στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο επίσημα αυτό το μήνα και θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει το Συμβούλιο, πρέπει να συνενέσει και πώς θα αντιδράσει την πρόταση του Κοινοβουλίου. Επίσης, είπα πολλές φορές στο παρελθόν ότι το γραφείο μου είναι μικρό αλλά έχει μεγάλα, μεγάλα καθήκοντα και εντολή και για να μπορέσει η ομάδα μου να εκπληρώσει αυτά τα καθήκοντα προς το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων υπάρχουν τέσσερις προϋποθέσεις ε, που πρέπει να λάβουμε υπόψη και στο μέλλον. Πρώτον, φυσικά, η ανεξαρτησία που είναι το κλειδί οποιοδήποτε διαμεσολαβητή. Να υπάρχει ένα ανεξάρτητο φορέα ε, προ τον οποίο θα προσφεύγουν οι πολίτε εάν δεν του εξυπηρετεί καλά η δημόσια διοίκηση. Δεύτερο στοιχείο, το οποίο αφορά ε, τις δύο ερευνητικές αρμοδιότητες που έχει το γραφείο μου, ισχυρές αρμοδιότητες, δηλαδή ο αναφέροντας είναι στο ίδιο επίπεδο με το θεσμικό όργανο, αναφέ, έχει δυνατότητα να φέρει όλες τα στοιχεία της υπόθεσης. Ε, μπορούμε να ερευνήσουμε τα, τα έγγραφα της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καλέσουμε υπαλλήλους να καταθέσουν. Έχουμε αυτέ τι δύο ε, αρμοδιότητες που είναι πολύ ουσιαστικέ για να ενισχύσουν την ήπια δύναμη και τις που έχει το γραφείο μου. Ε, χαίρομαι που τι κρατήσαμε αυτέ τι σημαντικέ αρμοδιότητε. Τρίτο στοιχείο είναι η πόρη. Αυτή τη στιγμή το γραφείο μου έχει 65 ε, θέσεις ε, σε δύο ε, τόπους ε, και ασχολείται με 2.000 παράπονα με στον χρόνο σε 24 γλώσσες. το 2018 είχαμε αύξηση κατά 17% των παραπώνων. Ε, τμήμα τη στρατηγική μα, τη στρατηγική μου, είναι να ξεκινήσουμε κάποιε έρευνε με δική μα πρωτοβουλία τα πρόσφατα χρόνια, ε, χάρη ε, και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο του Διαμεσολαβητών και αυτό αύξησε και την ορατότητά μα ε, και φτάνουμε και σε πιο πολλού πολίτε. Ε, η πρόταση του Κοινοβουλίου ζητάει μεγαλύτερη εμπλοκή του διαμεσολαβητή στου τομεί ε, των καταγγελώντων, whistleblowing, και ε, στι υποθέσει κατά τη παρενόχληση για να κάνουμε οτιδήποτε θα πρέπει να υπάρξει αύξηση του σπόρου στο γραφείο μου για να κρατήσουμε το, τα πρότυπα ψηλά και να εξυπηρετήσουμε του πολίτε καθώ θα χειριζόμαστε τα παραπονά του. Επίση, διαπαραταξική υποστήριξη είναι ε, εκ των όνου κάνευ για το γραφείο μου αυτό. Και όπω και η προκάτοχή μου θα προσπαθήσω να έχω την υποστήριξη όλου του Κοινοβουλίου για τη δουλειά που κάνω. Η ψηφοφορία το Φεβρουάριο έδειξε το γραφείο του διαμεσολαβητή απολαμβάνει διαπαραταξίακή. Ε, υποστήριξης και θέλω να είμαι στο ύψο των περιστάσεων και στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Ε, όταν υιοθετηθεί το Μάιο το νέο, εκλεγεί το νέο ε, κοινοβούλιο και υπάρξει και νέο πρόεδρος, θα δούμε τι θα γίνει με το μέλλον του γραφείου και ενημερωτικά σας λέω ότι η πρόθεσή μου είναι να ξανακατεύω υποψήφια και να πάρω και ανανέωση της ε, εντολής, της θητείας μου τότε θα βασιστώ ε, στη δουλειά που έχουμε κάνει από το 2013 και μετά και ε, πιστεύω ότι η χρησιμότητά μας, ε, χάρη στην στήριξη του Κοινοβουλίου, θα εδραιωθεί ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σας σήμερα και είμαι έτοιμη να απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ. Υπάρχει σαφώς ευρεία υποστήριξη. Είδατε ότι υποστηρίχθηκε στην Ολομέλεια με μεγάλη πλειοψηφία. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και ευχαριστούμε και εμείς για την εξαιρετική συνεργασία η οποία ελπίζουμε να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Μπορούμε τότε να περάσουμε κατευθείαν στην Επιτροπή. Ο κύριος Λεφεύρ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Ορέλη για την παρουσία της και δεν είναι η πρώτη φορά εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Μας ζητήσατε να σας ενημερώσουμε όσον αφορά το χρονοδιάγραμμά μας, όπως σήμερα έχει προγραμματιστεί σε σχέση με τη γνωμοδότηση. Καταλαβαίνετε ότι η επιστολή του Κοινοβουλίου έφτασε στις 25 Μαρτίου. Είναι ίσως λίγο νωρίς για να μπορέσουμε να σας υποβάλουμε ένα σοβαρό χρονοδιάγραμμα καθότι δεν υπάρχει απολύτως καμία προθεσμία ε, στην επιστολή του Κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ξεκινήσει την ανάλυση της προτινόμενης αναθεώρησης ήδη από την υιοθέτηση του ψηφίσματος και του σχεδίου κανονισμού, πριν από λίγες εβδομάδες δηλαδή, και η αναθεώρηση αυτή η οποία συμπεριλαμβάνει πολλές τροποποιήσεις και τροπολογίες που υιοθετήθηκαν στην Ολομέλεια θα πρέπει να κάνουμε μια εις βάθος ανάλυση και κατόπιν αφού τηρηθούν όλες οι εσωτερικές διαδικασίες σύνταξης διαβούλευσης με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και γενικές διευθύνσεις θα πρέπει στο τέλος να τηρήσουμε και την συνήθη ε, διαδικασία που ισχύει στην Επιτροπή. Βεβαίως δεν μπορώ να σας πω ποια θα είναι η ημερομηνία για την υποβολή της γνωμοδότησης, αλλά το συντομότερο δυνατόν και τηρώντας ε, την ε, διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί θα σας ε, ενημερώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λεφεύρ, λέει πρόεδρος. Κύριε Ορέλη, θέλετε να απαντήσετε. Α, ο Πίτερ. Όπως πάντα ο Πίτερ. Καταρχήν θα ήθελα να χαμογελάσω Νομίζω ότι την επόμενη φορά δεν θα ξαναστείλουμε επιστολή στην Επιτροπή χωρίς προθεσμία, χωρίς ημερομηνία. Τέλος πάντων, ναι. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή για τη συνεργασία της. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στη λέξη διαφάνεια και να απαντήσω εδώ στην κυρία Ορέλη. Για μένα διαφάνεια στην τριμερή συμμετοχή στο διάλογο που έχουμε μεταξύ ημών της Επιτροπής και του Συμβουλίου, νομίζω θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τους ε, πολίτες και τις προσδοκίες τους, οι οποίοι μας παρακολουθούν αν υπάρχει διαφάνεια στις ανταλλαγές απόψεων που έχουμε μεταξύ μας, στις διαδικασίες. Και νομίζω ότι κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών, παραδείγματο χάρη, όταν μιλάμε για διαφάνεια, μιλάμε για μια ξεκάθαρη διαδικασία. Πολλές φορές είναι ονομαστική η ψηφοφορία μας. Διαφάνεια επίσης σημαίνει και αυτό ελπίζω στην επόμενη θητεία να αυξηθεί αυτή η διαφάνεια και αυτό μπορεί να γίνει και μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών αλλά νομίζω και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή βρίσκεται σε καλή κατεύθυνση αλλά για μένα η δυσκολία συνεχίζει να εμφανίζεται στο Συμβούλιο. Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Δεν θέλω τώρα να μπω στις λεπτομέρειες ε, της διοικητικής διαδικασίας ε, στο Συμβούλιο, αλλά αποφασίζει κάτι το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη ακολουθούν, υλοποιούν και ουσιαστικά συνεχίζει να υπάρχει αυτή η συνειδητοποίηση ότι κάπου αλλού στις Βρυξέλλες, κάπου μακριά, κάποιες μυστικές διαδικασίες αποφασίζουν και επιβάλλουν. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το ξαναδούμε. Το Συμβούλιο θα πρέπει να αντιμετωπίζει με περισσότερη διαφάνεια και τις δικές του διαδικασίες αλλά και αυτά που συμβαίνουν εδώ στο Κοινοβούλιο γιατί νομίζω ότι τα κράτη-μέλη και για το καλό και για το κακό βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες από κάποιον λαμβάνονται και βεβαίως ο ρόλος του διαμεσολαβητή σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε αυτή η διαφάνεια να αυξηθεί και αυτό να γίνει με ένα πιο ευανάγνωστο τρόπο, να σταματήσει αυτό το μαύρο κουτί με το οποίο πολλές φορές παρομοιάζουμε το Συμβούλιο και από το οποίο βγαίνουν κάποιες αυθαίρετες αποφάσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ, Πίτερ. Θα ήθελα και εγώ να υπενθυμίσω σε όλους το άρθρο 228 της Συνθήκης ε, για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά κάνει μία έκκληση προς όλα τα κρατημέλη να υιοθετήσουν και πως όλα τα θεσμικά όργανα να υιοθετήσουν διατάξεις για να διευκολύνουν την λειτουργία και την εφαρμογή των αποφάσεων του Ombudsman, του διαμεσολαβητή. Και βεβαίως μέχρι το τέλος Μαρτίου, αλλά και ουσιαστικά μέχρι το τέλος της θητείας μας Έχουμε ακόμα κάποια βήματα να κάνουμε. Εννοείται ότι αυτό θα συνεχιστεί και στην επόμενη θητεία και πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν. Κυρία Ορέλη, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως, πάρα πολύ ενδιαφέρον θα είναι να μπορέσουμε να δούμε και εμείς τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τη διαφάνεια, συμφωνώ πολύ με αυτά που είπε ο κύριος Γιάρ. Και κυρίως ε, το θέμα που αφορά τη διαφάνεια στο Συμβούλιο, που ευθύθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Υπάρχουν κάποιες συστάσεις από μέρους μας. Πρώτον, όσον αφορά τα κράτη-μέλη, δεν ζητάμε δημοσίευση, αλλά ζητάμε να εγγράφονται κάπου οι λήψεις αποφάσεων. Όντως, Πολλές φορές οι διαδικασίες δεν βασίζονται σε έγγραφα. Τα έγγραφα είναι πολύ λίγα, οι δημοσιεύσεις είναι πολύ λίγες. Αλλά σίγουρα και βάσει του κανονισμού 1049 θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που τηρούνται. Τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, Κάποιες από τις αποφάσεις δεν είναι εύκολο να περάσουν και να στηριχθούν από πλειοψηφία. Και εδώ στο Κοινοβούλιο βεβαίως υπάρχει ευρεία υποστήριξη αυτών. Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στο Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κρατημέλη όπως η Δανία, η Σουηδία, η Ολλανδία που έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους. Νομίζω και η Προεδρία της Φιλανδίας που έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους η διαφάνεια να γίνει μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας τους. Απ' την άλλη βεβαίως έχουμε και τις εκλογές και παρόλο που οι κρίσεις όπως αυτή του Brexit έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες υπάρχουν και κάποια θετικά που απορρέουν από αυτές τις κρίσεις. Οι Ευρωπαίοι πολίτες σήμερα έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα, περισσότερο. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό εδώ να δείξουμε το ρόλο των θεσμικών οργάνων, ότι υπάρχει λογοδοσία και να σταματήσει αυτή η θεωρία ότι κάπου αποφασίζονται όλα αυτά στις Βρυξέλλες και ότι παίζουν ρόλο και οι θεσμοί αλλά και τα άτομα. Ωραία. Έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο, στο εργαστήριό μας για τη σύγκρουση συμφερόντων, ακεραιότητα, λογοδοσία και διαφάνεια στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Είναι από το τμήμα ΓΑΜΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό προετοίμασε το εργαστήριο αυτό. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους εδώ και θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Τέρι Κάμπρας πρώτα απ' όλα. Τον παρακαλώ να έρθει εδώ και να συμπροεδρεύσει μαζί μου αυτό το κομμάτι της συνεδρίασής μας. Λοιπόν, αγαπητοί ευρωβουλευτές, ομιλητές, συμμετέχοντες, ε, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σε αυτό το εργαστήριο και επιτρέψτε μου να αρχίσω με κάποιες τεχνικές πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι η συμμετοχή είναι για όλους, έτσι, σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες. Η διερμηνία θα υπάρχει σε όλες τις γλώσσες σήμερα, εκτός από τα πορτοκαλικά, τα φιλανδικά, τα τσεχικά, τα ελεθουανικά και τα κροατικά. Να ξέρετε επίσης ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο το εργαστήριο αυτό, οι παρεμβάσεις δηλαδή των ομιλητών θα μαγνητοσκοπούνται επίσης. Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες, ό,τι έχουμε ηλεκτρονικά δηλαδή υπάρχει διαθέσιμο και σε χαρτί και βέβαια ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας. Οπότε και πάλι καλώς ήρθατε. Το εργαστήριο αυτό επικεντρώνεται στην σύγκρουση συμφερόντων στο ευρύτερο πλαίσιο ακαιρεότητας, λογοδοσίας και διαφάνειας μέσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς τους ευρωπαϊκούς. Όπως όλοι γνωρίζουμε τα θέματα αυτά αλληλοσυνδέονται. και υπάρχει βέβαια κράτος δικαίου που διασφαλίζει τη δημοκρατία σε μια οικονομία που λειτουργεί. Θέλουμε λοιπόν έτσι να προωθήσουμε την καλή διακυβέρνηση και να ενισχύσουμε επίσης την νομιμότητα και την αξιοπιστία όλων των ε, δημοσίων ε, οργάνων. Υπάρχουν πολύ σημαντικά εργαλεία για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και τις πρακτικές κακής διακυβέρνησης. Πρέπει να αποφεύγουμε, να προλαμβάνουμε, να εντοπίζουμε και να λύνουμε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Και γι' αυτό εμείς στην Επιτροπή μας αυτή σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με στόχο σιγά σιγά να ξεκαθαρίζουμε και να ενισχύουμε το ηθικό πλαίσιο μέσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς. Είναι μια διαδικασία που εννοείται ότι δεν τελειώνει ποτέ. Δεν είναι ότι λέμε μπράβο τσεκ αυτό το έκανα και τελείωσε. Επανακτιμάται η κατάσταση συνεχώς. Όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν ε, τα δυνατά του σημεία και τις αδυναμίες τους. Και πρέπει λοιπόν όλοι να φροντίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλύψουμε τα κενά, όπως ε, υπογραμμίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14 η Σεπτεμβρίου του 2017 για την διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όπως επίσης και σε ένα άλλο ψήφισμα της 13 Δεκεμβρίου του 2018 στην ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητε του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017. Την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα εγκρίναμε την απαλλαγή για το 2017 όπου εκφράστηκε εκεί ε, ξεκάθαρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις συγκρούσεις συμφερόντων, κυρίως όταν πρόκειται για τον ορισμό υψηλά ειστάμενων αξιωματούχων, ε, όπως επίσης σε σχέση με τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ζητήσεων μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. Εδώ πέρα θα ακούσουμε την κυρία Ορέλη που την ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή της εδώ. Ε, θα μας παρουσιάσει τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως χάρη στο έργο της και θα μας μιλήσει και για τις προκλήσεις που έχουμε στο μέλλον. Μετά θα ακούσουμε τον Κριστιαν Ρόκ, που είναι διευθυντής για υγεία και ευημερία και συνθήκες εργασίας στην Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια, θα ακούσουμε για την σύγκρουση συμφερόντων στις ε, διάφορες ευρωπαϊκές υπηρεσίες από την κυρία Αναστασιάδη, η οποία αντικαθιστά την Έλεν Φως, που είναι καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ και η οποία ρώστησε ξαφνικά. Θα μας παρουσιάσει λοιπόν τα προκαταρτικά ευρήματα μελέτης που ανέθεσε η, το τμήμα ε, πολιτικής για τα δικαιώματα των πολιτών και σταγματικές υποθέσεις και στο τέλος θα ακούσουμε τον κύριο Ντέρκ Ντέτκεν που είναι επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας και ασφάλισης της ΕΦΣΑ. Θα μας μιλήσει για το δίκτυο ε, οργανισμών, για τη σύγκρουση συμφερόντων στην διαχείριση των ευρωπαϊκών ε, οργανισμών επίσης. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο και πάλι στην Έμιλη Ορέλη για την αρχική της παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα. Θέλω να κάνω την εξή παρατήρηση. Γενικά, τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σημειώσει πρόοδο, είναι πιο ανοιχτά, λογοδοτούν περισσότερο τα τελευταία πέντε χρόνια. Με τη στήριξη και την πίεση του Κοινοβουλίου. Το γραφείο μου, η κοινωνία των πολιτών και χιλιάδε ε, δημόσιοι που δουλεύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετούν τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνεια, λογοδοσία ε, και θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό. Φυσικά, ε, οι επιδόσεις διαφέρουν από φορέα και θεσμικό όργανο σε θεσμικό όργανο. Και γενικά έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κακοδιοίκηση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν λήψεις μετά από έρευνες που έχουμε κάνει και όπως έχω πει ε, και στο παρελθόν, η Κομισιόν του Γιούνκερ έχει κάνει προσπάθειες ούτως ώστε να γίνουν τα θεσμικά όργανα πιο ανοιχτά και να λογοδούν περισσότερο. Αυτός είναι ο σκοπός εξάλλου της διαφάνειας. Η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της Κομισιόν και του Γραφείου μου είναι γενικά καλή και δημοσιεύει τώρα ε, τα πρακτικά της Κομισιόν με τους λομπίστες και προσπαθούμε να βελτιώσουμε το αρχείο διαφάνειας. Έχουν αναθεωρηθεί ε, οι κανόνες για τους ειδικούς συμβούλους και ο κώδικας διοντολογίας της Κομισιόν. Έχει ε, βελτιωθεί η διαφάνεια των εμπορικών συνομιλιών και υπάρχει ψηλό επίπεδο διαφάνειας στις συνομιλίες για τον Brexit. Η Κομισιόν επίσης ήταν το προθεσμικό όργανο το οποίο μετά τις συστάσεις μου δημοσίευσε τα ονόματα ε, των ανωτάτων υπαλλήλων τα οποία φεύγουν και πάνε στον ιδιωτικό τομέα μαζί με τις συνθήκες ε, που τους βάζει η Κομισιόν για να διαχειριστεί τη σύγκρουση συμφερόντων. Ε, και άλλα θεσμικά όργανα ακολουθούν το ίδιο παράδειγμα και εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις τι υποχρεώσει του με βάση το άρθρο 64 του κανονισμού υπηρεσιακή κατάσταση και αυτά είναι καλά, αλλά μπορούν να γίνουν περισσότερα σε αυτόν τον τομέα. Έκλεισα μια έρευνα πρόσφατα για το πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται την ε, κατάσταση των κυλιόμενων θυρών, α πούμε, των ε, ε, υπαλλήλων τη που φεύγουν από την Κομισιόν και πάνε ας πούμε, στο ιδιωτικό τομέα. Ε, δεν γίνονται αυτά εν μία νυχτή. Και ω διαμεσολαβήτρια προσπαθώ να επιφέρω μία πιο μακροπρόθεσμη αλλαγή νοοτροπία. Χρειάζεται λοιπόν επιμονή. Ε, όταν ένας δημόσιο υπάλληλο πάει στον ιδιωτικό τομέα ή αντίστροφα, γίνεται μια υγιή ανταλλαγή δεξιοτήτων και προσόντων. Όμω αυτές οι κυριόμενες ε, θύρες ε, συνοδεύεται από πιθανού σοβαρού κινδύνου και πρέπει να του διαχειριστούμε αυτού του κινδύνου. Ε, Αυτέ οι κυλιόμενε στήρε μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο σύγκρουση συμφερόντων με τι υποχρεώσει ενό δημοσίου υπαλλήλου, παραδείγματο χάρη να αποκαλυφθούν εμπιστευτικέ πληροφορίε ή να χρησιμοποιηθούν κακώ και μπορούν ε, να χρησιμοποιήσουν πρώην υπάλληλοι ε, τι επαφέ του ε, και να τι χρησιμοποιήσουν ε, προ το συμφέρον του στα λόμπι. Ε, φυσικά αυτό σημαίνει ότι μπορεί και η δημοσιοπαλληλοί ε, και γενικά η δημοσιοπαλία να υποφεληθεί όταν προσλαμβάνει κόσμο από τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί, α πούμε, έχουμε πολύ καλά ειδικευμένα άτομα σε τεχνικού τομεί. Θα πρέπει να τονίσω ότι το δικαίωμα στη δουλειά είναι θεμελιώδε. Και οποιασδήποτε οποιοδήποτε περιορισμοί πρέπει να είναι θεμητοί και αναλογικοί. Επίση, σε τεχνικό επίπεδο, η Κομισιόν έχει σημειώσει πρόοδο από τότε που κλείσαμε την πρώτη έρευνα σε αυτόν τον τομέα πριν από αρκετά χρόνια. Όμω, η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάσει αν μπορεί να έχει μια πιο στεναρή προσέγγιση για να αντιμετωπίσει σοβαρέ περιπτώσει σύγκρουση συμφερόντων, ειδικά σε μικρέ περιπτώσει ανωτά των υπαλλήλων που φεύγουν και πάνε στον ιδιωτικό τομέα σε ορισμένε σπάνιε περιπτώσει θα πρέπει να εξετάσει και την απαγόρευση αυτών των ε, κανόνων που προβλέπει ο κανονισμό υπηρεσιακή κατάσταση. Επίση, ζήτησα από την Κομισιόν να δημοσιεύει περισσότερε πληροφορίε και σε πιο τακτικά διαστήματα για τους, το μικρό αριθμό ε, υπαλλήλων που φεύγουν από την Κομισιόν ή από του εκτελεστικού οργανισμού και πάνε σε διάφορε νομικέ εταιρείε, σε λόμπι ή ω σύμβουλοι. Ξέρω, α πούμε, ότι ο πρώτο πρώην Γενικό Γραμματέα Αλεξάνδρου Ταγιάννου, ε, πήγε σε μια νομική εταιρεία όπου με βάση την ιστοσελίδα της νομικής ε, εταιρείας αυτή, δίνει στρατηγικές ε, συμβουλές σε πελάτες για παγκόσμια θέματα που αφορούν τον ανταγωνισμό, διεθνές εμπόριο, ξένες επενδύσεις και ρυθμιστικά θέματα. Είναι σαφές από την ανακοίνωση της εταιρεία για τον ε, διορισμό του πόσο σημασία δίνει στις γνώσεις του ανθρώπου αυτού, ειδικά σε ό,τι αφορά τις συγχωνεύσεις ε, ε αντιμονοπολιακού χαρακτήρα και στις κρατικές ενισχύσεις. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε και να συμφιλιώσουμε ε, το θεμητό δικαίωμα εργασίας με τις υποχρεώσεις που έχει ε, ένας πρώην δημόσιο υπάλληλος, ένας συνταξιούχος δημόσιο υπάλληλος και τις ε, ανάγκες του ιδιωτικού τομέα, ε, για τον, για τον οποίο η δυνατότητα του να αποκτήσει γνώσεις και πρόσβαση σε δίκτυα τους οφούν στο να προσλάβουν υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Δημοσίου Υπαλληλίας. Υπάρχει και μια επιπλέον έρευνα που θα γίνει το 2020 για αυτό το θέμα των κυλιόμενων θυρών για να αξιολογήσουμε κατά πόσο έχει σημειωθεί πρόοδο αυτό το θέμα και στη διαφάνεια. Φυσικά, μερικέ φορέ υπάρχουν διστάμενε απόψει με την Κομισιόν. Ένα παράδειγμα ήταν το πώ ε, χειρίστηκε το διορισμό πέρυσι του σημερινού Γενικού Γραμματέα. Ε, στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα για την απαλλαγή του προπολογισμού, το Κοινοβούλιο επανέλαβε το πόρισμα ότι ίσως φτάσαμε στα όρια του νόμου. Ε, εγώ στηρίζω τις συστάσεις μου ότι η Κομισιόν θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη διαδικασία για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα της, χωρίς ανοιχτή και ανεξάρτητη διαδικασία από το διορισμό άλλων υπαλλήλων. Μετά από δύο ε, διαδοχικά παράπονα από ομάδε αυτού του Κοινοβουλίου, το 2018, περιμέναμε μέχρι να ολοκληρώσει ε, τη δουλειά τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και ξεκίνησαμε μια έρευνα για το πώ διορίστηκε αυτό το άτομο. Ε, εξετάσαμε χιλιάδε σελίδε εγγράφων και στο τέλο έκλεισα την υπόθεση με τέσσερα διαφορετικά απορίσματα κακοδιοίκηση. Η Κομισιόν αρνήθηκε να αναγνωρίσει έστω ότι αυτός ο διορισμός θα μπορούσε να, είχε, να τον είχε αντιμετωπίσει καλύτερα, στο πούμε έτσι, ήπια και να δώσει συνέχεια στην σύστασή μου και να βελτιώσει τα πράγματα στο μέλλον. Επίσης, αγνόησε πάρα πολλά ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, από ό,τι φαίνεται. Η ζημία για την διαδοχή των γεγονότων είναι προβληματική δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και στα πλαίσια μάλιστα των επερχόμενων εκλογών. Επίσης, επέλεξα να θεωρήσω ότι αυτή η υπόθεση είναι ιδιόρυθμη. Είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, δεν αντιπροσωπεύει ε, το τεράστιο αριθμό ε, επαφών που έχει η Κομισιόν με τον διαμεσολαβητή και ήταν εξαιρετικής φύσεως. Και αυτό συνδέεται πάρα πολύ με τον πολύ ε, σημαντικό ρόλο που παίζει ο Γενικός Γραμματέας και με το επίπεδο ορατότητας πολιτικής, ας πούμε, και γενικότερα ασυνήθιστης για ένα δημόσιο υπάλληλο. Φυσικά, ο Γενικό Γραμματέα έχει την εμπιστοσύνη του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Κολέγιου των Επιτρόπων. Συμπρασματικά, η διοίκηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υψηλά πρότυπα και πολύ συχνά υψηλότερα από αυτά που υπάρχουν στα περισσότερα κράτη-μέλη. Και σίγουρα ε, είναι συγκρίσιμα με αυτά των ΗΠΑ και άλλων ε, χωρών του κόσμου. Αλλά υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένες περιπτώσεις που είναι πολύ ε, έντονα στο, στη δημοσιότητα. Και αυτό μπορεί να υποσκάψουν το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Δημοσιοπαλληλία. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε και να το παρεμποδίσουμε να συμβεί στο μέλλον. εγώ συντονίζω το Ευρωπαϊκό ε, δίκτυο ε, διαμεσολαβητών με πάνω από 90 αρμόδιες αρχές. Ε, προεδρεύω σε διάφορες συνεδριάσεις. Φέτος θα γίνει μια συνεδρίαση 8 Απριλίου που θα συζητήσουμε το, την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα είναι πρόεδρος σε αυτή την εκδήλωση και ο κύριος Μπαρνιέ, μάλιστα, ο επίτροπο, θα κάνει και μια βασική ομιλία. Τέλος, για να αναγνωρίσω την πολύ καλή δουλειά που έκαναν πολλοί ε, Ευρωπαίοι δημόσιοι υπάλληλοι, ε, το 2017 ε, ξεκινήσαμε μία εκδήλωση για την απονομή ενό βραβείου για περιπτώσεις καλής διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι μια θαυμάσια μαρτυρία για την σκληρή δουλειά, την αφιέρωση, τη δέσμευση και τη σκληρή δουλειά που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Η τελετή θα γίνει τον Ιούνιο φέτο και είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για το γραφείο μου για να τονίσει τι καλέ διοικητικέ πρακτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση και την καθημερινή σκληρή δουλειά των Ευρωπαίων υπαλλήλων σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο, συνάδελφοι. Όχι. Ερωτήσεις, και απαντήσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη διαδικασία γιατί από ό,τι κατάλαβε η κυρία Ορέλη πρέπει να μας εγκαταλείψει. Ερωτήσεις λοιπόν από μέρους των συναδέλφων. Βιρζινή Ροζιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία της ε, μεσολαβητή σήμερα εδώ. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για μας, ιδιαίτερα για την Επιτροπή μας, η δική σας εργασία και αυτό φαίνεται και από την διοργάνωση της σημερινής μας συζήτησης στα πλαίσια αυτού του εργαστηρίου με θέμα την ακυρεότητα, διαφάνεια και σύγκρουση συμφερόντων. Εμείς, ε, αλλά όχι μόνο εμείς, μόνο η πολιτική μας ομάδα, ε, επιμείναμε να υπάρξει αυτή η συζήτηση εδώ, γιατί κάποια πρόσφατα γεγονότα μας δείχνουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει πραγματικά να παίξει ένα ρόλο ουσιαστικά προβάλλοντας την εργασία σας και πιέζοντας κάποια θεσμικά όργανα να μην κλείνουν τα μάτια και τα αυτιά τους στις πολύ σημαντικές σας ε, προτάσεις. Μιλάμε για διοντολογία, για καλή διαχείριση και διακυβέρνηση, για διαφάνεια. Αξίες τις οποίες προβάλλουμε είναι κοινή μας, ε, ε, κοινός μας αγώνας και σίγουρα θα αναφερθούμε σε θέματα διαφάνειας, καθεστώτος του διαμοσολαβητή, εκθέσεις δραστηριοτήτων πολύ βασικές αξίες της δραστηριότητάς σας που ουσιαστικά στηρίζουν την νομιμότητα όλων των θεσμικών οργάνων. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές και αξίες, τότε όλη η νομιμότητα και η αξιοπιστία μας ε, υπονομεύεται. Μετά από αυτή την πενταετία, ίσως θα πρέπει να ασκήσουμε και κάποια κριτική. Πέντε χρόνια κατά την άποψή μου πολύ γεμάτα με δυσκολίες. Η ορθή διακυβέρνηση που ταλαιπωρήθηκε θα έλεγα ξεκινώντας από τις δραστηριότητες του κυρίου Μπαρόσου σε μια πασίγνωστη τράπεζα, την Goldman Sachs με μια σαφέστατη παραβίαση και του πνεύματος αλλά και του γράμματος των ε, κειμένων των υποχρεώσεων που διέπουν το καθεστώς του κάθε επιτρόπου. Αναφερθήκατε και εσείς σε επαφές με μεγάλους τραπεζίτες. Δεν θα αναφερθώ στην υπόθεση της κυρίας Κρός, Νέλ Κρός. Και βεβαίως το θέμα της τοποθέτησης ε, με τρόπο κάπως αυθαίρετο του κυρίου Σαλμάιερ στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Αμφισβητήσιμο τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Αμφισβητούμενο, συγγνώμη. Και θα αναφερθώ μόνο σε αυτούς, μόνο σε αυτές τις πιο προφανείς περιπτώσεις. Κατά τα άλλα, η θεσμοί μας, οι διαδικασίες μας λειτουργούν με παραδειγματικό τρόπο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπονομευτεί η εξαιρετική τους λειτουργία από τέτοιες υποθέσεις. Πώς μπορεί κάποιος να έχει εμπιστοσύνη στην ουδετερότητα ενός θεσμού που είναι και θεματοφύλακα των συνθήκων εάν αγνοώντας ε, όλους τους κανόνες και αναφερθήκατε ξεκάθαρα σε τέσσερις ε, προφανείς υποθέσεις παραβίασης, με την πολύ συγκεκριμένη παραδείγματο χάρη διαδικασία ε, της τοποθέτησης κάποιου επικεφαλής ο οποίος ανήκει με εμφανή τρόπο σε ένα πολιτικό κόμμα. Καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις, οι διορισμοί και όσον αφορά το τυπικό κομμάτι αλλά και όσον αφορά την προσπάθεια κάλυψης αρχικών σφαλμάτων και ε, ανομαλιών στη διαδικασία. Και πραγματικά σήμερα δεν καλούμαστε να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη αλλά να οικοδομήσουμε μια εμπιστοσύνη που έχει χαθεί και η οποία εμπιστοσύνη έχει πραγματικά υπονομηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα θεσμικά όργανα. Και επειδή κοιτούμε την επόμενη θητεία και τις προοπτικές της, θα ήθελα να ακούσω από εσά τι μπορούμε συγκεκριμένα να κάνουμε, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τους κανόνες. Οι κανόνες υπάρχουν, δεν εφαρμόζονται όμως. Ίσως πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί οι κανόνες γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές τηρείται το γράμμα του νόμου, αλλά όχι το πνεύμα. Αυτό ήθελα να σας πω και πραγματικά το λέω περιμένοντας από σας με απελπισία μια απάντηση. Η εκθέσεις για την επικινδυνότητα της λιφοζάτης ε, θα δημοσιευθούν πολύ πρόσφατα και εκεί θα είχα κάτι να πω και πραγματικά περιμένουμε ε, τις προτάσεις σας ε, για να αποφύγουμε μια παρόμοια κατάσταση με αυτή που ζήσαμε σε αυτή την θητεία. Η κυρία Γκρέσλερ, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε εκ μέρους της Επιτροπής Προπολογισμού. Κυρία Ορέλη, αυτή η υπόθεση με το Γενικό Γραμματέα μας απασχόλησε πάρα πολύ στην δική μας Επιτροπή. Και σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση που υποβάλατε. Έχω τρεις ερωτήσεις. Υπάρχει μια διαδικασία διοικητική και θα θέλαμε να ξέρουμε εάν προσπαθήσουμε να επικαλεστούμε όλες αυτές τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις, πώς μπορείτε να βοηθήσετε, να στηρίξετε έτσι ώστε αυτές οι διαδικασίες να τηρούνται. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερον, ε, διάβασα με μεγάλη προσοχή αυτά που γράψατε για την όλη υπόθεση και τις 1200 ε, σελίδες που δημοσιεύσατε. Δεν ξέρω αν ε, όλα αυτά τα έγγραφα πραγματικά μπορούμε να τα μελετήσουμε. Μιλήσατε πολύ συγκεκριμένα και για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να μας πείτε τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε όσον αφορά τις διαδικασίες, πέραν αυτών που εμπεριέχονται σε αυτές τις 1200 σελίδες. Κοιτάξτε, εμείς πραγματικά τρεις φορές ζητήσαμε την ε, παρέτηση του Γενικού Γραμματέα. Τρεις φορές και πρόκειται πραγματικά για μια πολύ ξεκάθαρη διαδικασία από μέρους μας. Ο διορισμός ε, πολλών γενικών ε, διευθυντών που μας ανακοινώνεται και βλέπουμε ότι ο τρόπος, η διαδικασία επιλογής τους έχει βελτιωθεί. Αυτό είναι για μας μια πολύ σημαντική πρόοδος. Βήματα προς την σωστή κατεύθυνση. Αλλά όσον αφορά το θέμα της ε, πιθανότητας παρέτησης ε, από τη θέση του Γενικού Γραμματέα, μπορείτε να μας πείτε εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει πράγματα τα οποία τελικά δεν υλοποιούνται, δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ η κυρία Ρίβαση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Τιμεσαλαβήτρια. Πάντα με ενδιαφέρουν πολύ οι εκθέσεις σας. Και αυτή τη φορά σκέφτομαι ότι υπάρχει κάτι το οποίο με απασχόλησε πάρα πολύ τα τελευταία πέντε χρόνια και είναι το θέμα της πραγματογνωμοσύνης. Είτε πρόκειται για τους οργανισμούς μας. Υπάρχει ΕΦΣΑ, υπάρχει ΕΜΑ, Σίγουρα έχει γίνει πρόοδος, όμως η πραγματογνωμοσύνη όταν έχουμε σύγκρουση συμφερόντων ε, από τους εμπειρογνώμονες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους εμπειρογνώμονες καταλαβαίνετε ότι τα συμπεράσματά τους είναι για μας προβληματικά. Έτσι λοιπόν, εμείς οι Ευρωβουλευτές, οι πράσινοι που φτάσαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τι δείχνει αυτό, δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Για να έχουμε πρόσβαση στις επιστημονικές μελέτες έπρεπε να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να πούμε ότι όλες οι μελέτες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον πρέπει να είναι ανοιχτέ στο δημόσιο, γιατί είναι θέμα δημοσίου συμφέροντος. Βλέπετε λοιπόν ότι αν εμεί, οι Ευρωβουλευτέ, αναγκαζόμαστε να φτάσουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ε, κάτι δεν λειτουργεί καλά στα θεσμικά μα όργανα και υπάρχει αδιαφάνεια που δεν συνάδει με αυτά που λέμε για διαφάνεια των ε, Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Δύο πράγματα λοιπόν εδώ έχουμε. Το ένα είναι θα έχουμε τις ευρωεκλογέ. Αυτές οι ευρωπαϊκές ε, εκλογές έρχονται και είμαστε υποχρεωμένοι εμείς οι οικολόγοι για την Ευρώπη που θέλουμε να στηρίξουμε να έχουμε εγγύσει. Δεν θα ήταν καλό λοιπόν εσείς πριν από τις εκλογές να δημοσιεύατε μία χάρτα, ε, ένα κώδικα θεντολογίας με κατανομή ρόλων. Τι πρέπει να κάνουν οι επίτροποι, τι οι υπάλληλοι, γιατί και εδώ συχνά πρέπει να τα λέμε. Δεν θέλουμε περιστρεφόμενες θύρες. Πρέπει να υπάρξει άδεια για να μετακινηθεί κανείς από τον ένα τομέα στον άλλον ή για να δεχτεί δώρα πάνω από 300 κτλ. Ο αναφέρθηκε σε ρύθμιση. Μήπως θα μπορούσαμε από σήμερα με όλες τις εκθέσεις να προσπαθούσαμε να φτιάξουμε μια χάρτα δεοντολογίας και να καταλήξουμε σε κανονικότατη ρύθμιση στην επόμενη θητεία και να υπάρχει και μια ανώτατη αρχή για τη διαφάνεια. Γιατί αν ο κάθε οργανισμό, η κάθε υπηρεσία κάνει τα δικά τη. Θα τα δούμε μετά με του ενδοκρινικού διαταράχτες, γιατί ο καθένα έχει το δικό του ορισμό. Αν υπήρχε λοιπόν μια υψηλή αρχή για τη διαφάνεια, θα είχαμε την εγγύηση ότι δεν κάνει ο καθένα τα δικά του. Γιατί όταν ο καθένα έχει τι δικέ του εσωτερικέ ρυθμίσει, ορίζει εντελώ διαφορετικά το ότι είναι σύγκρουση συμφερόντων. Άρα, σαμποτάρεται τελικά ο καλό σκοπό. Θα ήθελα τη γνώμη σα από αυτού. Η για τις περιστρεφόμενες θύρες μιλάνε για πέντε χρόνια. Εμείς έχουμε 18 μήνες. Μήπως θα πρέπει να βάλουμε τρεις μήνες. Όταν πρόκειται για αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν στον ιδιωτικό τομέα, οι επίτροποι, οι υψηλοί υπάλληλοι μας όταν εγκαταλείπουν την υπηρεσία τους εδώ. Γεια, ο τελευταίος. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τις γενικές παρατηρήσεις Νομίζω ότι είναι επίκαιρο το θέμα και βεβαίως οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν ήδη μπει σε ένα πνεύμα προεκλογικό και εννοείται ότι υπάρχουν πολλές σημαντικές ε, αν θέλετε διαδικασίες που θα θέλαμε να είχαν ε, διεκπεριωθεί με άλλο τρόπο και βεβαίως τι θέλουμε να αλλάξουμε, πώς θέλουμε να εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι καλή στιγμή για να συζητήσουμε αυτά εν ώψη των ε, νέων εκλογών και όλες οι καλές ιδέες και οι βέλτιστες πρακτικές δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Βέβαια, έχετε δίκιο ότι πρέπει να συζητήσουμε και τα πράγματα τα οποία δεν πήγανε καλά και για μένα το όριο είναι πάντα η νομιμότητα και θα πρέπει να αναφέρουμε όλες αυτές τις πρακτικές όπου το πνεύμα το γράμμα του νόμου παραβιάζονται. Το θέμα της διαφάνειας, επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένως. Μπορούμε να πούμε ότι πού αρχίζει και πού τελειώνει η διαφάνεια. Γιατί εμένα ως ένα βαθμό με φοβίζουν Αναφερθήκατε στην υπόθεση της ΕΦΣΑ, αλλά υπάρχουν και άλλες, και άλλες περιπτώσεις. Από τη μία λέμε ότι θέλουμε η εμπερογνωμοσύνη μας, οι πραγματογνώμονες να μπορούν να λειτουργήσουν. από την άλλη, αναρωτιόμαστε. Πρέπει να δίνονται με λεπτομέρεια όλες οι πληροφορίες, όλα τα στοιχεία σε βαθμό που αν θέλετε θα δημοσιεύουμε και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και όλες τις ανακαλύψεις. Εδώ μπορεί να είναι προβληματική αυτή η πρακτική. Κάπου λοιπόν θα πρέπει να παραμείνουμε σε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Ναι, διαφάνεια, αλλά θα πρέπει η ζωή μας να μην γίνει δύσκολη. Και εγώ παίρνω σαν παράδειγμα την Εύσα γιατί όσον αφορά παραδείγματο χάρη την περίπτωση των ε, ενδοκρινικών διαταρακτών, ξέρουμε ότι η ίδια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε και εκεί. Τώρα, όσον αφορά τις ε, προσφυγές και όσον αφορά τις ε, περιπτώσεις που επιλύονται στα δικαστήρια. Κοιτάξτε, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα αυτό δεν είναι κάτι το αρνητικό και νομίζω ότι μεταξύ της διαφάνειας που ζητούμε σε περιπτώσεις που αφορούν συγκεκριμένα άτομα, φυσικά πρόσωπα και τις διαδικασίες, νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση και βεβαίως κάθε φορά όταν υπάρχουν παράπονα, διαμαρτυρίες, προσφυγές, ισχυρισμοί και απαιτήσεις, διεκδικήσεις να μπορούμε κατά περίπτωση επαναλαμβάνω να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ της διαφάνειας και των ε, πραγματικών γεγονότων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς τώρα για να απαντήσετε στις ερωτήσεις οποίες μπορείτε να απαντήσετε και στις άλλες που δεν είσαστε σε θέση να απαντήσετε τώρα αμέσω αν νομίζετε έτσι, μπορείτε να επανέλθετε αργότερα. Ε, κύριε Ρέλη, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις της κυρίας Ποζιέ. Αντιλαμβάνομαι την απογοητευσή σας που την εκφράσατε σε σχέση με τις συστάσεις που δεν γίνονται, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο θα αλλάξει την κατάσταση είναι καλή ηγεσία. Είναι καλή θεσμική ηγεσία, είτε πολιτική είτε διοικητική. Και ελπίζω στην περίοδο αυτή στην οποία αναφέρεται ο κύριος Γιάρ να υπάρξει προβληματισμός για το τι έγινε τα θέματα τα οποία είτε εγώ ανέφερα είτε εδώ στο κοινοβούλιο εσείς αναφέρετε. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος είναι ακριβώς να ενώσετε στελίτσες για αυτά τα θέματα που συμβαίνουν, τα επίμαχα, ε, τον ευρωσκεπτικισμό και την εχθρότητα απέναντι στην Ευρώπη. Να τα συνδέσετε αυτά τα δύο, γιατί το ότι ανεβαίνει ο ευρωσκεπτικισμός, ο λαϊκισμός και η εχθρότητα απέναντι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι κάτι που μερικές φορές οφείλεται σε αυτά. Ή χρησιμοποιούν υποθέσεις που οδηγούν στο να εκμεταλλεύονται κάποιοι καταστάσεις και να δημιουργούν ε, εικόνες καρικατούρας σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το είδα. Αυτά που είπατε, με ποιο τρόπο εμφανίστηκαν ε, στα μέσα ενημέρωσης πολύ ε, διαφορετικά από την πραγματικότητα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ombudsman. Και αν δείτε την περίπτωση Μπαρόσο, και εκεί εγώ διερεύνησα να δω πώς το χειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπήρξε ε, κάτι, ή αναφερόταν κάτι στον κώδικα δοντολογίας, ίσως όχι αρκετά έντονα όπως θα ήθελα, αλλά αναγνωρίστηκε το πρόβλημα εκεί. Κάτι το οποίο δεν έγινε στις άλλες υποθέσεις. Κάτι άλλο στο οποίο αναφέρθηκα και στην αρχή για τους επένους όσον αφορά την καλή διακυβέρνηση. Το έκανα ακριβώ για να πω ότι πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Να μην αφήνουμε πάντα την κακή εικόνα να υπερισχύει, κακή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οφείλεται και σε αυτές τις πρακτικές στις οποίες αναφερθήκαμε εδώ, αλλά και στο Brexit και σε οτιδήποτε άλλο. Εγώ προσπαθώ να υπογραμμίσω την καλή δουλειά που γίνεται επίση. Αλλά πάνω από όλα αυτό που χρειάζεται είναι προβληματισμός από την πολιτική και διοικητική ηγεσία, προβληματισμός για το τι συμβαίνει, πού οδηγεί και τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτό στο μέλλον για τις ερωτήσεις της κυρίας Γκράσλε και τις διοικητικές διαδικασίες. Ξέρετε ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και είναι και αυτό ένα από τα θέματα που χρειάζονται πρωταθλητές. Και εσείς το λέτε ότι ίσως θα πρέπει να έχουμε πιο συγκεκριμένους κανόνες για το τι μπορεί κανείς να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει ώστε να μην γλιστράει ανάμεσα στις γραμμές κανείς και αποποιείται τις ευθύνες του. Να μην υπάρχει κάτι αφηρημένο, να ξέρουμε τι είναι το δημόσιο συμφέρον, την ακαιρεότητα, πολύ συγκεκριμένα. Ναι, με μια νομοθεσία αναγκαστικά θα τα πούμε πολύ συγκεκριμένα. Και εντάξει, υπάρχει αξία σε αυτό που λέτε, ναι. Από την άλλη όμως, έχω ακούσει ότι σε μια πραγματικά καλή διοίκηση, μια πραγματικά καλή διοίκηση, χαρακτηρίζεται από τι, από λίγους κανόνες και ρυθμίσεις, όσο γίνεται λιγότερου. Γιατί βλέπετε υπάρχει μια νοοτροπία η οποία ισχύει και η οποία επιτρέπει να συμπεριφέρονται οι υπάλληλοι καλά, ε, χωρίς να χρειάζεται να του το επιβάλλει κανείς με τον νόμο. Χωρίς να χρειάζεται ένα πρωτόκολλο, μια νομοθεσία. Αλλά εντάξει, αυτό είναι κάτι που ε, πρέπει να μας προβληματίσει ίσως σε αυτή την περίπτωση να είναι χρήσιμη μια νομοθεσία για να βελτιωθούν και οι διοικητικές πρακτικές γενικότερα. Όσον αφορά τώρα την διερεύνηση που κάναμε και τα χιλιάδες πρακτικά που εξέτασαν οι συνεργάτες μου, πολλά από αυτά ήταν ε, κάποια σχέδια. Κοιτάξτε, είδα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει αρκετά. Η δικιά μου δουλειά είναι συμπληρωματική. Σκέφτηκα πώς θα μπορούσε να βοηθήσει το γραφείο μου. Και κατάφερα να βρω διάφορα έγγραφα και ελπίζω να κατέγραψα τα γεγονότα χρονολογικά, ώστε όποιος διαβάζει την έκθεσή μου να μπορεί πολύ εύκολα να δει τι έγινε πότε και να καταλήξει σε συμπεράσματα. Ίσως να υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαν ε, να, να επιπλέον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά έτσι όπως έχει έκθεση σήμερα, εγώ πιστεύω ότι έχουμε καταγράψει την υπόθεση βάσει των εγγράφων στο οποίο μπορέσαμε να φτάσουμε. Τώρα για το 1049 για το περιβάλλον, ότι χρειάστηκε να προσφύγετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και εδώ, ό,τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το 1049, όντως κράτησε πάρα πολύ και μια ιστορία που έχει αρχίσει πολύ πριν εμφανιστώ εγώ εδώ, είναι πολιτικά ζητήματα. Ε, ο κόσμος αλλάζει, έχει αλλάξει πάρα πολύ από το 1049 και μετά. Υπάρχει ένα θέμα και καταλαβαίνω την απογοητευσή σας και είναι ότι έχουμε την αίσθηση πως είναι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που ελέγχουν την πληροφορία. Αυτό είναι που σας ενοχλεί, το καταλαβαίνω. Για να το παρακάμψουμε αυτό, εσείς αναγκαστήκατε να πάτε στο δικαστήριο. Αν είχατε έρθει στο δικό μου το γραφείο, θα ήθελα να το είχατε κάνει. Εγώ δεν είμαι δικαστήριο για να, κάνω, να καταλήξω σε δεσμευτικές αποφάσεις, αλλά θα μπορούσε ίσως να είχα βοηθήσει με τις διαδικασίες και πάλι για το 1049 αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη στιγμή οι πολιτικοί και διοικητικοί πρωταθλητές, όπως είπαμε και νωρίτερα, που θα αναλάβουν. Κύριε Γιάρο, όσον αφορά τη διαφάνεια, ε, την είχαμε αυτή την ε, συνομιλία πολλές φορές ξανά. Δεν είναι δυνατόν να δώσει κανείς ξεκάθαρα απαντήσεις ασπρομαύρο Η διαφάνεια για μένα δεν είναι αυτός σκοπός, είναι ένα εργαλείο για να λογοδοτεί κανείς. Ό,τι ίσχυε πριν από 10 χρόνια ε, δεν φτάνει σήμερα. Οπότε και εδώ καταλαβαίνω τη δικιά σας απογοήτευση για το πώς θα φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα για τα όρια της διαφάνειας, όπως λέτε. Πάντως, σε διάφορες υπηρεσίες έχει λειτουργήσει καλά η διαφάνεια. Και θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια, πριν γίνω διαμεσολαβήτρια, ο κύριος Διαμαντούρος πριν από μένα είχε κάνει πάρα πολλή δουλειά για τη διαφάνεια στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμούς και είχε κάνει διάφορες ε, δοκιμές. Δεν υπήρχε τίποτα για εμπορικές ε, απόρριτες πληροφορίες. Το θέμα δεν είναι να ξέρουμε από τι είναι φτιαγμένα τα φάρμακα. Πάντως για πολύ καιρό με τη δουλειά που έκαναν οι υπηρεσίε μου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άλλαξε η νοοτροπία για τη διαφάνεια. Σίγουρα υπήρξαν περιπτώσεις ε, όπου φτάσαμε στα δικαστήρια με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πάντως έγιναν αλλαγές που μπορεί να μην είναι ικανοποιητικέ απόλυτα ούτε για τη μία ούτε για την άλλη πλευρά, αλλά είμαστε σε, ένα, σε μια λογική κατάσταση και από εκεί και πέρα παίρνουμε και μαθήματα από το παρελθόν. Πάντως συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και το είπα και πριν. Με ρωτάνε αν θέλω 100% διαφάνεια. Κοιτάξτε, η διαφάνεια είναι καλή όταν είναι για το δημόσιο συμφέρον. Μερικές φορές όμως είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος να μην αποκαλυφθούν κάποια έγγραφα κάθε ρύθμιση δεν αποκαλύπτει απαραίτητα όλα τα στοιχεία πριν ε, γίνει νόμος. Μερικές φορές το δημόσιο συμφέρον είναι να αποκαλυφθούν, μερικές φορές όχι. Η διαφάνεια στις περισσότερες περιπτώσεις δεν κάνει κακό. Αν όμως κάνει, Πάντως ευχαρίστω να δώσω συνέχεια σε όλα αυτά που άκουσα εδώ σήμερα. Πρόεδρος, βεβαίω, Και αυτό που κάναμε εμεί στην τελευταία συνάντηση συντονιστών είναι ότι επεκτείναμε την επίσκεψη, την πρόσκληση μάλλον πιο σωστά, και στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Και χαίρομαι που η πρόεδρος της Επιτροπής αυτή η κυρία Γκρέσλερ, δέχτηκε την πρόσκλησή μα και ήρθε σήμερα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σα εδώ σήμερα και Περιμένω να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. And Ωραία, και τώρα συνεχίζουμε. Και εδώ χαίρομαι πολύ που θα δώσω το λόγο στον κύριο Κρίστιαν Ροκ από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τη Δημοσιολαβήτρια. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω και να σα εξηγήσω τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την αντιμετώπιση τη σύγκρουση συμφερόντων. Είναι ένα θέμα που προέρχεται από διάφορα στοιχεία, είτε από αυτού που κατέχουν κάποιο δημόσιο αξίωμα, τις οικογένειές τους ή προσωπικά συμφέροντα, ή άλλα συμφέροντα όπως λέει και το κείμενο, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιος δέχεται δώρα ή φιλοξενία. Κάτι επίσης που είπε η κυρία Βασιλοβήτρια ή περιστρεφόμενες θύρες. Λοιπόν, έχουμε εμεί κανόνες και είμαστε τυχεροί γι' αυτό, είτε το δημοσιονομικό κανονισμό, είτε το καταστατικό του προσωπικού, που ειπε και η διαβασολαβήτρια η περιστρεφομενες στήρες. λοιπον εχουμε εμει κανονες και ειμαστε τυχεροι γι αυτο ειτε το δημοσιονομικο κανονισμο ειτε το καταστικό του προσωπικου που εξηγει πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την σύγκρουση συμφερόντων. Θα ήθελα λοιπόν να σας εξηγήσω ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες. Αλλά να πω επίσης ότι η τήρηση κατά γράμμα του τι σημαίνει και ποιος είναι ο ορισμός της σύγκρουσης συμφερόντων είναι στοιχείο κλειδί για να μπορούμε να ε, σεβαστούμε και τα δικαιώματα που προσφέρουν τα ίδια αυτά κείμενα στους υπαλλήλους. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάλεξε την διαφάνεια, λαμβάνοντας υπόψη το όσα είπε η Διαμεσολαβήτρια πριν από λίγο, διαφάνεια, γιατί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύουμε ότι ο δημόσιος έλεγχος ενισχύει την ευαισθητοποίηση και τον ε, ρόλο που αποκτά ο καθένας από εμά σε περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων. Θα σας εξηγήσω ποιοι είναι οι κανόνες μας. Και θα τους διαιρέσω τους κανόνες αυτούς, σε αυτούς που εσείς εγκρίνατε και σε αυτούς που έχουμε στο εσωτερικό και στο καταστατικό του προσωπικού. Όταν λοιπόν δούμε πώς εφαρμόζονται οι κανόνες, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το χρονοδιάγραμμα. Τι γίνεται πριν την θητεία κάποιου, κατά τη διάρκεια της θητείας του και μετά. Τόσο ισχύει αυτό για τους επιτρόπους, τους πολιτικούς, όσο και για το προσωπικό. Λοιπόν, για τους επιτρόπους υπάρχουν κανόνες που αναφέρονται στη συνθήκη, είναι το άρθρο 245 και 247, αλλά υπάρχει και ο κώδικας δεοντολογίας ο νέος, γιατί υπήρχε και πριν ένα από το 2018 έχουμε το νέο. Και αυτός ο νέος κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται σε συγκεκριμένους κανόνες για να καταπολεμάμε τη σύγκρουση συμφερόντων. Πριν αναλάβει κανείς, ο Επίτροπος πρέπει να κάνει μια δήλωση συμφερόντων. Τι επενδύσει έχει, θέσεις, ε, χρήματα πάνω από 10.000 ευρώ, όλα πρέπει να αναφέρονται. Και επίση οτιδήποτε άλλο προκύψει πρέπει να αναφέρεται. Συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα, σε συνδικάτα, επαγγελματικέ δραστηριότητες, επίσης ζύγου ή συντρόφων. Κατά τη διάρκεια τώρα τη θητεία, πρέπει κάθε χρόνο να δηλώνουν την 1η κάθε χρόνο επίσης όλα αυτά τα στοιχεία. Και βέβαια αν υπάρξει αλλαγή όποτε αυτή προκύψει. Κατά τη διάρκεια επίση τη θητεία, θα πρέπει να ενημερώνουν αν υπάρξει οποιαδήποτε ανάκριση ή βρίσκονται κοντά σε τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, όταν κάποιος δέχεται ένα δώρο ή μια φιλοξενία πάνω από 150 ευρώ δώρα πρέπει να τα δηλώνουν και να τα δέχονται μόνο βέβαια αν πρόκειται για διπλωματικούς λόγους ή για λόγους πρωτοκόλου και για την φιλοξενία δεν πρέπει κανείς να την δέχεται τα δώρα, αν είναι παραπάνω, πρέπει να φτάνουν να καταλήγουν στο πρωτόκολλο. Ή αν κάποιος κερδίσει χρήματα από κάποιο μάθημα που διδάσκει, ε, τις απολαβές του πρέπει να τις δορίζει σε κάποιον ανθρωπιστικό σκοπό. σε πολύ συγκεκριμένε περιπτώσεις μόνο μπορούν να τα δεχτούν. Συμμετοχή τώρα στην πολιτική ζωή. Εδώ υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Είμαστε σε μια πολιτική επιτροπή υγιών ο ο πρόεδρός μας το καυτό. Λοιπόν, αν συμμετέχετε ως επίτροπος σε τοπικές περιφερειακές ε, εκλογές, είσαστε υποχρεωμένος να πάρετε άδεια εκλογική άνευ αποδοχών. Άλλο αν είσαστε υποψήφιοι σε ευρωεκλογέ. Γιατί τότε, ναι, μένα δεν έχετε πια τις απολαβές σας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά δεν χρειάζεται να πάρετε εκλογική άδεια. Τώρα, μετά την θητεία σας, και αυτή είναι μια καλή εξέλιξη, για δύο-τρία χρόνια για τον πρόεδρο, δύο χρόνια για του επιτρόπους, πρέπει να κοινοποιήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα να λαμβάνουν που μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων. Και υπάρχει και μια ανεξάρτητη ηθική επιτροπή η οποία εξετάζει όλε αυτέ τι υποθέσει και μπορεί να εκφράσει συστάσει προ το σώμα των επιτρόπων και επίση προβλέπονται και κυρώσει. Είτε πρόκειται για επίπληξη, είτε πρόκειται για παραπληκτικό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για το προσωπικό υπάρχουν δύο στοιχεία, δύο πυλώνες. Υπάρχουν και εδώ και εσωτερικοί κανόνες και κώδικας διοντολογίας. Το προσωπικό έτσι καλλιώς αναλαμβάνει να συμπληρώσει ένα έντυπο και είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί για προσωπικούς λόγους να σταματήσει να δουλεύει για κάποιους μήνες κάποιος από το προσωπικό. Όταν επιστρέψει όμως πρέπει να συμπληρώσει επίσης ένα έντυπο για να εκφράζει εκεί οποιαδήποτε υποψία μπορεί να υπάρχει για σύγκρουση συμφερόντων. Έπειτα, ό,τι ισχύει και για του επιτρόπου, ισχύει και εδώ για την φιλοξενία κτλ. Απασχόληση. Είναι πολύ περιορισμένη. Κανονικά απαγορεύεται. Έχετε πάντα τη δυνατότητα να αναλάβετε κάποιες δραστηριότητες, όχι βέβαια τις ώρες εργασίας και πολύ περιορισμένες απολαβές. Και αυτό για να μπορεί να διατηρεί τη σχέση του με το σώμα ο υπάλληλο. Τώρα, δύο χρόνια αφού φύγει από την υπηρεσία, αν ε, η δραστηριότητα που αναλαμβάνει έχει να κάνει με τις αρμοδιότητές του τα τελευταία τρία χρόνια της θητείας του, πρέπει να στήσει άδεια από τη δίκηση. Δεν δίνεται αυτή αυτόματα. Μερικές φορές τώρα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μπορεί να απαγορευτεί ή εν πάση περιπτώσει περιορίζεται πάρα πολύ η άδεια. Τώρα υψηλά σταμενοί αξιωματούχοι. Επίσης έχουν την υποχρέωση να μην προβούν σε κανένα είδου λόμπινγκ 12 μήνες αφού εγκαταλείψουν τις υπηρεσίες τους. Και κάτι πολύ σημαντικό, η διαφάνεια. Δημοσιεύονται όλες οι απαγορεύσεις που επιβάλλονται στο προσωπικό. Έπειτα, δημοσιονομικός κανόνας. Εδώ αναφέρεται ρητά τι είναι η σύγκρουση συμφερόντων για να περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις και με ποιο τρόπο πρέπει να ενημερώσει κανείς αμέσως τον διατάχτη για οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος ώστε αν υπάρχει τέτοια σύγκρουση συμφέροντος να απομακρυνθεί από το συγκεκριμένο αντικείμενο ο υπάλληλο και να αναλάβει κάποιο άλλο. Οι κανόνες έχουν ενισχυθεί και όσον αφορά τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες. Και το προσωπικό εκεί συμπεριλαμβάνεται στους ίδιους περιορισμούς. Η διαμεσολαβήτρια έχει εγκρίνει τους κανόνες αυτούς, τα ακούσαμε. Είναι και τα συμπεράσματα της μελέτης που έγινε για τις ε, περιστρεφόμενες θύρες. Μία ήταν η σύσταση και αυτή είναι ότι όταν κάποιος φεύγει από την υπηρεσία να μην μπορεί να αναλάβει κάποια άλλη θέση τα πρώτα χρόνια. Έχει πάρει αποφάσεις δικαστικές και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το δικαίωμα ε, ανάληψης ε, απασχόλησης αφού εγκαταλείψει την υπηρεσία. Εμείς να ξέρετε ότι φτάνουμε πάντα ε, στα όρια των όσων επιτρέπονται. Τώρα, για τον ορισμό της σύγκρουσης συμφερόντων, τι σημαίνει. Πρέπει να υπάρχει συμφέρον. Πρέπει να υπάρχει συμφέρον. Δεύτερον, πρέπει να είναι τέτοιο που να εμποδίζει την αμεροληψία του υπαλλήλου. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό πρέπει να γίνεται για κάποιον τρίτον. σημαίνει ότι κάποιο τρίτο πρέπει να κοιτάξει όλα τα στοιχεία, αλλά πρέπει να κοιτάξει επίση κατά πόσο θεωρείται λογικό να θεωρήσει αυτή η τρίτη πλευρά ότι μπορεί να μην είναι αμερόληπτος πια υπάλληλο. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό, γιατί άμα θέλουμε μια καλή διακυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος. Δεν μπορεί να είσαι, ας πούμε, στην ε, Κριτική Επιτροπή για έναν ε, συνάδελφο όταν αυτός έχει δουλέψει για σένα πριν από μερικά χρόνια. Εκτός αν είναι σαφές για όλους ότι τον ήξερε αυτόν τον υπάλληλο και θεωρούν επίσης ότι μπορεί να τον κρίνεις χωρίς να μεροληπτήσεις. Διαφάνεια τώρα και συνειδητοποίηση. Αυτά είναι τα βασικά για μας, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρουμε ότι έχει αναλάβει πάρα πολλές πρωτοβουλίες για την διαφάνεια, να υπάρχει ένα μητρό διαφάνειας για τις σχέσεις που έχουμε με τρίτες πλευρές, όπως επίσης για τα έξοδα αποστολής για τους επιτρόπους, για τις σχέσεις τους με lobbyists. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο Μητρό. Και συνειδητοποίηση. Και εδώ θέλω να σας πω δύο λόγια για τη συνειδητοποίηση. Συνειδητοποίηση των υπαλλήλων μας. Για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να αποφεύγεται σύγκρουση φερόντων από τα άτομα τα οποία έχουν καταλήψει την υπηρεσία. Υπάρχουν κανόνες ηθικής. Κάνουμε training, ε, μαθήματα, σεμινάρια, ελέγχους, όλο το χρόνο, διασκέψεις για την ηθική και όταν είναι κάποιος υπάλληλο, αλλά και όταν εγκαταλείψει την υπηρεσία. Και αυτό πολύ σημαντικό για την καταπολέμηση της σύγκρουσης συμφερόντων. Όλα αυτά ευθυγραμμίζονται απόλυτα από τον Πρόεδρό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και προσβλέπω σε παρατέρω συνεργασία μου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Χοκ. Τώρα, θα σας υποβάλουμε ερωτήσεις αφού ακούσουμε όλες τις παρεμβάσεις, αν σας πειράζει. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Έλεν Φως καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Μάστριχτ. Συγγνώμη, έλεγε λάθος ε, η ημερήσια διάταξη. Η Νατάσα Θανασιάδου, λέ, επίκουρος καθηγητής στην ε, νομική σχολή ε, του Πανεπιστημίου του Μάστρετ που αντικαθιστά την κυρία Φως. Ευχαριστούμε την επίκουρο καθηγητή, την κυρία Αναστασιάδου. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Πρόεδρε, δεξιότιμοι βουλευτέ. Ε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε τα πρώτα πορίσματα της μελέτης μας για τη σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις ε, ενωσιακέ υπηρεσίες και οργανισμούς ε, υπό την αιγίδα της Erlen Foss και μια ομάδα ακαδημαϊκών που έκαναν αυτή την έρευνα ε, κατόπιν ετήσεω του Policy Department του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα πολιτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την τον Οτάβιο Ματζότη για τη θαυμάσια συνεργασία. Ήταν ο υπάλληλο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το Policy Department. Θα σα παρουσιάσω το, τη δομή τη έρευνας, τη μεθοδολογία και θα σας παρουσιάσω τις έννοιες της ανεξαρτησίας και της σύγκρουσης συμφερόντων και συνεχεία θα εστιάσω ε, στις περιπτώσει συγκρούσεων συμφερόντων επιλεγμένων ευρωπαϊκών οργανισμών και μετά θα μιλήσω για το ερωτηματολόγιο που θα μοιραστεί στο δίκτυο ε, ευρωπαϊκών οργανισμών ούτω ώστε να συλλέξουμε εμπειρικά στοιχεία και πληροφορίες και θα καταλήξω με κάποια προκαταρτικά πορίσματα γιατί όπως σας είπαμε αυτή η μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί. Λοιπόν, ποιο είναι ο στόχο αυτή τη μελέτη. Ο στόχο είναι να αξιολογήσει του κανόνε και τι πολιτικέ για τη σύγκρουση συμφερόντων στου οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση με αίσθηση στι αποκεντρωμένε υπηρεσίε και να εξετάσουμε ε, εάν ε, ο έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλο ιδιαίτερο μπορεί να βελτιωθεί και αν υπάρχει ανάγκη να απλουστεύσουμε και να ενισχύσουμε την συνέπεια των διαφόρων και συνοχή των διαφόρων κανόνων που υπάρχουν. Ε, θέλουμε να έχουμε ένα πλαίσιο για την εξαρτησία και την σύγκρουση συμφερόντων και να συστηματοποιήσουμε τους κανόνες που είναι ποικίλοι και διαφορετικοί. Εξετάσαμε λοιπόν τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον ε, κανονισμό υπηρεσιακή κατάσταση τη Ένωση, τι ιδρυτικέ πράξει όλων των ε, εκτελεστικών οργανισμών και του εσωτερικού κανονισμού επιλεγμένων οργανισμών. Αξιολογήσαμε επίση και θα αξιολογήσουμε περαιτέρω τι συστάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στα πλαίσια της διαδικασίας απαναγής και της πιο τελευταίας διαδικασίας επαναλλαγή, ε, το, τα όσα λέει ο ΣΑ, η ΜΚΟ, ε, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, το Ελεκτικό Συνέδριο κτλ. Και μέσω της συνεργασίας με την Επιτροπή Κοντ και ΠΕΤΗ θα συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες και το δίκτυο των ενωσιακών οργανισμών. Έχουμε ένα δικό χάρτη, θα σας και ένα ερωτηματολόγιο αργότερα, και τα τελικά πορίσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν ε, μέχρι 1η Ιουλίου του 2019. Θα ξεκινήσω με την έννοια της ανεξαρτησίας. Γιατί μόνο όταν ορίζουμε από ποιον κάποιον πρέπει να είναι ανεξάρτητος, μπορούμε να αποφανθούμε τι σημαίνει ε, σύγκρουση συμφερόντων για αυτό το άτομο και τι μπορεί να τον δεσμεύει. Με βάση τις συνθήκες της Ένωσης, προβλέπεται ποια είναι η ανεξαρτησία, θα έπρεπε να είναι η ανεξαρτησία τη Κομισιόν από τα κράτη-μέλη, από άλλου ε, θεσμικού οργανισμού και από ιδιωτικά συμφέροντα. Σε ό,τι αφορά τι ε, όμω ενωσιακέ υπηρεσίε και οργανισμού, οι συνθήκε λένε ότι η Ευρωπαϊκή Επαλληλία πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Αλλά από ποιον πρέπει να είναι ανεξάρτητοι αυτοί οι οργανισμοί. Δεν είναι σαφέ. Επίση, οι ιδρυτικοί κανονισμοί έχουν συγκεκριμένε διατάξει για την ανεξαρτησία. Είτε για το σύνολο του οργανισμού, ή για συγκεκριμένους φορείς, παραδείγματο χάρη ο εκτελεστικό διευθυντή ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά επειδή υπάρχει υβριδική φύση των οργανισμών αυτών, είναι σαφές ε, από ποιον υπάρχει εξαρτησία, από την Κομισιόν, από την Κεντρική Διοίκηση, από τα κράτη-μέλη, από ποιον. Τα κράτη-μέλη εξάλλου συχνά συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο των Οργανισμών. Ή μήπω σημαίνει εξαρτησία μόνο από τα ιδιωτικά συμφέροντα η θεσμική δομή των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ξέρουμε, είναι πολύ περίπλοκη. οι οργανισμοί και ειδικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπλέκεται στον σχεδιασμό των οργανισμών και στη λειτουργία των οργανισμών αυτών, καθώς και τα κράτη-μέλη εμπλέκονται επίσης ε, στην ε, διοίκηση, στη διαχείριση καθώς και η σχέση με τους stakeholders. Δεν είναι τόσο εύκολο να ξεκαθαριστεί και να απομονώσουμε τους οργανισμούς από τις ομάδες συμφερόντων οι οργανισμοί χρειάζονται αυτή την πραγματογνωμοσύνη και χρειάζονται και εξειδικευμένο προσωπικό που έχει εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα και χρειάζονται συχνά εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού κλάδου. Είναι δύσκολο λοιπόν να βρούμε τη σωστή ισορροπία και να ε, έχουμε μια πραγματική καλή πολιτική για τη σύγκρουση συμφερόνων που θα λαμβάνει υπόψη και την ανάγκη όμως για εμπειρογνωμοσύνη που έχουν οι οργανισμοί της Ένωσης. Ποιος είναι ο ορισμός ε, της σύγκρουσης συμφερόντων. Ε, βασίζεται αναγκαστικά στην έννοια της ανεξαρτησίας αυτός ο ορισμός. Η σύγκρουση συμφερόντων, ο ορισμός σύγκρουσης συμφερόντων υπάρχει σε, διάφορες, σε διάφορα νομοθετικά κείμενα. Με διαφορές όμως. Εδώ τις μελετάμε τις διαφορές στη μελέτη. Φυσικά από τη μία έχουμε το δημόσιο συμφέρον και από την άλλη έχουμε το προσωπικό συμφέρον. Αλλά αυτά πώς ε, ορίζονται. Το δημόσιο συμφέρον είναι το συμφέρον της Ένωσης σε το συνόλο της ή είναι απλώς το συμφέρον μια συγκεκριμένης θέσης. Το συμφέρον της Ένωσης μπορεί να είναι κάτι πολύ γενικόλογο. Αν κοιτάξουμε όμως τη συγκεκριμένη θέση θα πρέπει να δούμε τα συμφέροντα που παίζουν σε σχέση με τη θέση και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει το άτομο αυτό που καταλαμβάνει τη θέση. Από την άλλη, το προσωπικό συμφέρον μπορεί να συμπεριλαμβάνει και το εθνικό συμφέρον, ε, που είναι ασύμβατο με, το, με τα συμφέροντα της θέσης ή με πολιτικά συμφέροντα, τα οποία μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση επίσης με τα συμφέροντα που εκπροσωπεί η θέση. Και η σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να λάβει διαφορετικές μορφές. Ε, μπορεί να είναι πραγματική, μπορεί να είναι δυνητική ή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ο Christian Rock είπε ότι η νομολογία κοιτάει την πραγματική σύγκρουση συμφερόντων και οι συστάσει του ΩΣΑ το ίδιο. Αλλά οι κανόνε ε, κανόνες του κανονισμού υπηρεσιακή κατάσταση ε, συμπεριλαμβάνουν και πιθανέ περιπτώσει σύγκρουση συμφερόντων. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι κανόνε είναι πολύ αυστηροί. Και αν κοιτάξουμε και του εσωτερικού κανόνε και τι κατευθυντήριε γραμμέ των οργανισμών γενικά, βλέπουμε κανόνε για πιθανολογούμενη σύγκρουση συμφερόντων. Ε, δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκρουση συμφερόντων. Δυνητικά δεν υπάρχει, αλλά μπορεί να θεωρηθεί από κάποιον ο σύγκρουση συμφερόντων. Βλέπετε λοιπόν την ευαισθησία. Και η ευαισθησία αυτή λαμβάνει υπόψη στου εσωτερικού κανόνε, ούτω ώστε να αντιμετωπιστεί και αυτή η λεπτή σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί απλώ να θεωρηθεί ότι υπάρχει από κάποιο. Στην αντίληψη κάποιου δηλαδή. Για να σα δώσω μια γεύση για τι τρέχουσε πρακτικέ, λοιπόν, θα εστιάσουμε σε λίγους ε, επιλεγμένους οργανισμούς Ένωσης που έρχονται σε επαφή με εξωτερικές ομάδες ε, συμφερόντων, με εξωτερικούς stakeholders και έχουν μεγάλο συμφέρον και εστίαση στη σύγκρουση συμφερόντων λόγω της θέσης τους. Ε, θα κοιτάξουμε λοιπόν ε, τον ΕΟΦ, ε, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Προϊόντων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο και το Γραφείο Διανοτική Διοκτησία. Ποιο είναι το πρόβλημα. Οι δηλώσει συχνά έχουν διαφορετική μορφή, είναι διαφορετικά τα έντυπα. Βλέπουμε, α πούμε, ότι οι οργανισμοί ε, ακολουθούν όλο και περισσότερο τι συστάσει που κάνει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φύγουμε από την αρνητική δήλωση, όπως λέμε, συμφερόντων. Εγώ, δηλαδή, δηλώνω προσωπικά ότι δεν έχω, δεν υπάρχει για μένα σύγκρουση συμφερόντων, ε, να το δηλώνουμε πιο θετικά. Να λέμε, δηλαδή, τι συμφέροντα έχω ως άτομο και συνεχεία να γίνεται μια αξιολόγηση για το αν υπάρχει σύγκρουση ή όχι συμφερόντων από την ιεραρχία, ας πούμε, από το, τα διορισμένα για αυτό το σκοπό άτομα. Μια άλλη διαφορά είναι το πεδίο της δήλωσης Παράδειγμα, έτσι. Το EMA, ο EOF, ε, απαιτεί δηλώσει ε, ε, για τα συμφέροντα που μπορεί να έχει κανεί απέναντι στην φαρμακοβιομηχανία. Ενώ ο ΕΚΑ ζητάει σύγκρουση δήλωση συμφερόντων στον νομοθετικό κλάδο τη δραστηριότητά του, στο ρυθμιστικό κλάδο τη δραστηριότητά του. Και η ΕΦΣΑ, πρέπει να, για την ΕΦΣΑ πρέπει να δηλώσει όλα τα συμφέροντα που που έχεις για το, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που καλύπτει η ΕΦΣΑ. Ακόμα ευρύτερο δηλαδή. Επίσης, ε, υπάρχει και διαφορά σε ό,τι αφορά το χρονικό διάστημα για τα συμφέροντα. Δύο έως πέντε χρόνια. Στις δηλώσεις ετήσια, τις κάνουμε ετήσια, μία άπαξ του έτους δηλαδή, ή ε, με αφορμή κάποια συνεδρίαση. Αυτό είναι γενικό. Υπάρχουν κάποιε διαφορές για τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονε. Ε, θα δείτε τι λεπτομέρειε στη μελέτη μα για του εξωτερικού εμπειρογνώμονε. Ό,τι αφορά του ε, συμβουλευτικού φορεί, μία από τι συστάσει ε, για αυτού έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ υπάρχουν διαφορέ και σε ό,τι αφορά την εντολή αυτών των φορέων και σε ό,τι αφορά τη σύνθεσή του. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφή στάση ενίσχυση των ε, φορέων αυτών, των συμβουλευτικών φορέων, ειδικά σε οργανισμού όπου έχουν την διακριτική ευχέρεια ε, να ασχοληθούν και με σύγκρουση συμφερόντων. Στη διαδικασία ελέγχου. Ποιο ελέγχει τη δήλωση αυτή για τη σύγκρουση συμφερόντων. Έχουμε και εκεί δει διαφορέ και έχουμε κατηγοριοποιήσει του οργανισμού ανάλογα με διάφορα μοντέλα. Αν έχουμε δηλαδή μια κεντρική διαδικασία ελέγχου ή αποκεντρωμένη διαδικασία ελέγχου και υπάρχουν και οργανισμοί που έχουν ένα μεικτό σύστημα, υβριδικό σύστημα. Τώρα, παρατηρήσαμε διαφορές ό,τι αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ε, για να μετριαστεί η σύγκρουση συμφερόντων όταν προκύψει. Βλέπουμε διαφορές. Μερικές φορές υπάρχει διακριτική ευχέρεια ε, να λάβει κάποια μέτρα ο οργανισμός όταν εντοπιστεί η σύγκρουση συμφερόντων. Άλλες, άλλοι οργανισμοί δεν έχουν αυτή την διακριτική ευχέρεια όταν βρεθεί σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνε εκ των προτέρων έτσι, και δεν μπορούν να αποκλίνουν από αυτού. Συνοψίζω. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να, έχουμε, να περισσότερο εμπειρικό υλικό και να εντοπίσουμε αυτές τις διαφορές μέσω ενός ερωτηματολογίου με τη βοήθεια του δικτύου ε, ευρωπαϊκών οργανισμών ε, και τα προκαταπτικά μας πορίσματα είναι τα εξή. Βλέπουμε διαφορά στις, ε, στα έντυπα των δηλώσεων, στις μορφές και υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη συγκρισιμότητα στις διάφορες δηλώσεις, στα διάφορα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τη δήλωση σύγκρουση συμφερόντων. Υπάρχει μια τάση ε, προς την εξωτερική ανάθεση σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση. Ποιο κάνει την αξιολόγηση, εξωτερικοί δηλαδή ε, άνθρωποι, εμπειρογνώμονες. Ε, και πώς θα μετριάσουμε τη σύγκρουση, μερικές φορές προβλέπεται αυτό από του εσωτερικού κανόνε, από τα κείμενα και άρα δεν έχει αρκετή διακριτική ευχαίρεια η διορισμένη αρχή να λάβει αυτά τα μέτρα για να μειωθεί η σύγκρουση συμφερόντων. Όπω είπε και η Πρόεδρο σήμερα το πρωί, η αντιμετώπιση τη σύγκρουση συμφερόντων ε, δεν είναι κάτι που τελειώνει, δεν γίνεται ad hoc, είναι κάτι που γίνεται συνεχώ και ελπίζουμε εμεί με την ε, μελέτη μα να συνεισφέρουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σχεδόν ε, τέλεια όσον αφορά την τήρηση του χρόνου ομιλία 11 λεπτά. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον τελευταίο μας ομιλήτη, τον κύριο Ντέτκεν, επικεφαλή τη Νομική Υπηρεσία της ΕΦΣΑ. Συγγνώμη, και θα μιλήσει εξ ονόματος ε, του δικτύου των ε, οργανισμών και ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα θα μιλήσω για την ανεξαρτησία σαν εκπρόσωπος των ε, οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανεξαρτησία είναι μια καθοριστική έννοια, η νομική, η οικονομική ανεξαρτησία, ανεξαρτησία από τις ρυθμιστικές αρχές. Και πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι περισσότερες από τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. Πάνω από 40 έχουν μια εντελώς ανεξάρτητη διοίκηση και διακυβέρνηση. Αλλά τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για ανεξαρτησία. Ανεξαρτησία από το νομικό πλαίσιο και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την περίπτωση της ΕΦΣΑ και βέβαια δεν είναι όλες οι διοικήσεις ακριβώς ίδιες τους διάφορους οργανισμούς. Έχουμε από το 2013 κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως ε, οι τρόποι εφαρμογής, τα συστήματα εφαρμογής, οι εφαρμοστικές διατάξεις διαφέρουν από τον ένα οργανισμό στον άλλο. Η ΕΕΦΣΑ, η Ευρωπαϊκή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων ανήκει στο δίκτυο και ακριβώς επειδή η διατροφή, τα τρόφιμα είναι κάτι το εξαιρετικά ευαίσθητο και εξαρτάται από τις ε, παραδόσεις των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Από την αρχή λοιπόν της λειτουργίας της ΕΦΣΑ η έννοια της εμπιστοσύνης ήταν καθοριστική και η αίσθηση ότι έπρεπε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας των τροφίμων ήταν πάντα κάτι που μας ε, απασχολούσε. Γι' αυτό ακριβώς για το 2017 το θέμα της απαλλαγής ήταν κάτι που μας χαροποίησε ιδιαίτερα αυτό κατά κάποιο τρόπο ενισχύει και την έννοια της ανεξάρτητης διακυβέρνησης για αυτόν τον οργανισμό. Σήμερα έχουμε την τρίτη γενιά κανόνων ανεξαρτησίας για την ΕΨΑ. Έχουν αλλάξει τρεις φορές και οι αλλαγές αυτές έχουν ε, βεβαίως άμεση σχέση και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα σχόλια που έγιναν στην ΕΦΣΑ μέσω της διαδικασίας της απαλλαγής έπαιξαν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά αυτές τις αλλαγές. Σε μεγάλο ποσοστό, 95% των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων ήταν αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας απαλλαγής και των σχολείων. Μπορούμε να πούμε ότι μάθαμε από την παρελθούσα εμπειρία μας, από τα σφάλματά μας και επαναλαμβάνω ότι οι συστάσεις είναι κάτι το καθοριστικό, κάτι στο οποίο βασιζόμαστε για να προοδεύσουμε. Επίσης, <clears throat> δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από το 2017 και πέρα βασιστήκαμε σε όλα τα σχόλια, στις συζητήσεις μέσω της δημόσιας διαβούλευσης και προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά για την εξέλιξή μας. Θα σας αναφέρω κάποια από τα χαρακτηριστικά της πολιτικής ανεξαρτησίας της ΕΦΣΑ. Και εμείς ε, έχουμε ενσωματώσει τη νέα διατύπωση, το νέο ορισμό, αν θέλετε, της σύγκρουσης ε, συμφερόντων. Η σύγκρουση συμφερόντων είναι μία κατάσταση, δεν είναι μία αξιόπινη πράξη, είναι κάτι στο οποίο μπορεί να βρεθεί κάποιος. Απλώς θα πρέπει να εντοπιστεί, όπως είπε και η προηγούμενη ε, ομιλήτρια, είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και ακριβώς γι' αυτό έχουμε προβλέψει μια περίοδο διετίας ε, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα πρέπει ο εν λόγω υπάλληλο, παραδείγματο χάρη, να ενσωματωθεί σε έναν άλλο ιδιωτικό οργανισμό από τη στιγμή που υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Λαμβάνουμε υπόψη μα επίση το γεγονό ότι η ΕΦΣΑ είναι ένα επιστημονικό φορέα, ένας φορέας επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης. Έχουμε λοιπόν ειδικού κανόνες που ισχύουν για όλους αυτούς που μετακινούνται από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα και αυτό σε ευρωπαϊκό ή σε εθνικό επίπεδο. Το θέμα της χρηματοδότησης επίσης και εδώ θα πρέπει να ισχύουν ειδικοί κανόνες έτσι ώστε αυτός ο επιστημονικός φορέας, αυτός ο επιστημονικός θύλακας που είναι η ΕΦΣΑ να διασφαλίσει την ανεξαρτησία του. Το θέμα των κυρώσεων, της διαφάνειας, εδώ είναι ένας πολύ λεπτός τομέας αυτός. Όπως ξέρετε, οι εμπειρογνώμονες που εργάζονται στην ΕΦΣΑ δεν είναι υπάλληλοι. Έχουν συμβατική σχέση με τον οργανισμό. Γι' αυτό και η διακοπή, η απόλυση είναι κάτι που θα πρέπει να συμμορφώνεται και να συνάδει με τους κανόνες μας. Πιστεύω επίσης ότι το θέμα της απαλλαγής είναι κάτι που μας οδήγησε σε νέους κανόνες, νέες πρακτικές, ιδιαίτερα στα πλαίσια της εμπειρογνωμοσύνης και της λειτουργίας του οργανισμού μας, της ΕΦΣΑ. Το θέμα των χορηγεών, της συμβατικής σχέσης ε, με κάποιους εξωτερικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες, αλλά και το γεγονός ότι κάποιοι από τους εμπειρογνώμονες που εργάζονται στην ΕΦΣΑ μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν κάπου αλλού. Ακριβώς γι' αυτό και εξετάζουμε τις αποδοχές με πολύ προσεκτικό τρόπο των εμπειρογνώμονων που εργάζονται στην ΕΦΣΑ. Και βεβαίως όλα αυτά βασίζονται σε εκ των προτέρων ελέγχους, εξάντε έλεγχοι, και βεβαίως η ενημέρωση και επικαιροποίηση σε προσωπικό επίπεδο των εμπειρογνωμόνων μας για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνονται ε, αυτές οι δημοσιεύσεις έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να ελέγξει βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που είναι δημόσια και γνωστά σε όλους. Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει, παραδείγματο χάρη, κάποιες αποφάσεις που λαμβάνει η ΕΦΣΑ. Λαμβάνουμε επίσης υπόψη μας και τις ε, συμφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και εκτός των επιστημονικών μονάδων και εμπειρογνωμόνων συγκεντρώνονται όλα αυτά τα στοιχεία στην νομική υπηρεσία. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν οι εξάντε έλεγχοι αλλά και οι ex post εκ των υστέρων, όταν ολοκληρωθεί δηλαδή η σύμβαση ενός εμπειρογνώμονα. Όσον αφορά την υλοποίηση για το 2018, για το 2018 έχουμε ήδη δημοσιεύσει στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσής μας τουλάχιστον 7.000 ελέγχους. Αυτό είναι περίπου και ο ετήσιος αριθμός ε, δημοσιεύσεων. Ο έλεγχος γίνεται και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από κοινού με κάποιους ε, ε, δημόσιους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τη στιγμή δηλαδή που ελέγχονται κάποιες από τις ε, αποστολές και μετά από ενδεχόμενες συστάσεις ή παρατηρήσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Και αυτό ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2019, αυτή η νέα πρακτική δημοσίευση στοιχείων. Εδώ βλέπετε, είναι και η τελευταία μου διαφάνεια, τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που ακριβώς έχουν εντοπιστεί τέτοιες περιπτώσεις στα πλαίσια της δικής μας δραστηριότητας ελέγχου, της ΕΦΣΑ, μπορείτε να σημειώσετε ότι δεν είναι ε, αυτές οι περιπτώσεις τις περισσότερες φορές εκεί που θα φανταζόταν κανείς. Σημειώνουμε επίσης ότι με αυτούς τους αριθμούς βλέπουμε ότι πολλοί εμπειρογνώμονες ακριβώς επειδή γνωρίζουν τους κανόνες δεν μπόρεσαν να υποβάλουν υποψηφιότητα καν για συνεργασία με τον οργανισμό μας, με την ΕΦΣΑ. Ολοκληρώνω. Σήμερα θα έλεγα ότι οι κανόνες της ΕΦΣΑ είναι κατά κάποιο τρόπο σημείο αναφοράς για πολλούς άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και το θέμα του ελέγχου, του δημόσιου ελέγχου αυτών των κανόνων και αυτών των διαδικασιών είναι για μας ε, εξαιρετικά σημαντικό. Η ποιότητα, η επιστημονική ποιότητα, αν θέλετε, των ε, αποστολών μας δεν αμφισβητείται από κανέναν, το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων λοιπόν πολλές φορές προκύπτει ακριβώς από αυτήν την εμπειρογνωμοσύνη. Τα στοιχεία όμως του 2017 προκύπτουν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Πιστεύουμε όμως ότι σήμερα το σύστημα που χρησιμοποιούμε είναι αποτελεσματικό, είναι βιώσιμο και θα μπορέσει να μας επιτρέψει και να εξελιχθούμε αλλά και να συνεχίσουμε να λειτουργούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στις ερωτήσεις, τα σχόλια. Έχετε το λόγο. Κυρία Ριβασί, εσείς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, χαίρομαι που μιλάμε για τη σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί εδώ και καιρό οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, κάποιοι ευρωβουλευτές είχαμε πρόβλημα σε αυτό με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμούς. Θέλω να ρωτήσω κυρίως αυτόν που εκφράστηκε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αλήθεια είναι, και πριν και η κυρία Ροζιά αναφέρθηκε στον κύριο Μπαρόσο, αλλά εγώ θυμόμαι τον κύριο Λενγκρέν, το θυμόσαστε, που ήταν ο διευθυντής της ΕΜΑ. Ο κύριος Λενγκρέν, όταν σταμάτησε τη σταδιοδρομία του εδώ, πήγε σε μια ιδιωτική εταιρεία και έφτιαξε ε, φαρμακευτική εταιρεία και εργαστήρια. Και μάλιστα όταν ακόμα δούλευε είχε ξεκινήσει αυτή τη δραστηριότητα. Ε, μιλήσατε για κυρώσεις. Στον κύριο Λεγκρέν δεν επιβλήθηκε καμία κύρωση, ήταν μόνο name and shame. Οπότε εγώ θέλω να ξέρω. Εντάξει να υπάρχουν οι κανόνες, αλλά αν δεν υπάρχουν κυρώσει, τι να τα κάνουμε αυτά. Ο κύριο Λεγκρέν τι έκανε, πήγε λοιπόν έφτιαξε το δικό του φαρμακευτικό εργαστήριο, πήγε και σύμβουλο σε ένα σωρό άλλα. Λοιπόν, κυρώσει είπατε. Μπορείτε να μου δώσετε κάποια παραδείγματα κυρώσεων που επιβλήθηκαν. Έπειτα. Για την ανεξαρτησία, εσείς κυρία μου υπονοείται ότι το πρόβλημα των εμπειρογνωμόνων είναι περίεργο γιατί αν θέλουμε καλούς εμπειρογνώμονες θα πρέπει να είναι εμπειρογνώμονες που να έχουν δουλέψει για τη βιομηχανία. Μα εγώ έχω την κυρία Μπουζάκ που είναι υπουργό στη Γαλλία και η οποία λέει ότι οι καλοί εμπειρογνώμονες είναι αυτοί που έχουν δουλέψει σε φαρμακευτικά εργαστήρια. Μα αν αυτό υπονοείται, τότε όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, είτε το Mediator, είτε άλλα σκάνδαλα, σκάνδαλα που ξέσπασαν στη Γαλλία έχουν να κάνουν ανθρώπους που δεν είχαν καμιά σχέση. Το Mediator, για παράδειγμα, ήταν η Ρεν Φνασόν, που ήταν πνευμονολόγος. Οπότε υπάρχουν πανεπιστημιακοί εμπειρογνώμονες που είναι ικανότατοι. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η γνώμη σας. Τι άκουσα και την έψα, έχω και για εσάς ερωτήσεις. Ποια είναι η ανώτερη αρχή για τη διαφάνεια που καλύπτει τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φροντίζει να υπάρχει ένας οριζόντιος ορισμός για τη σύγκρουση συμφερόντων και που να είναι ίδιος αυτός ορισμός για όλους και να κοιτάει κατά πόσο τηρείται από τους διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Γιατί εγώ δεν πιστεύω στον αυτό έλεγχο θα θελήσουμε να προστατεύσουμε τον έναν ή τον άλλον που είναι πιο σημαντικός ή που είναι πιο γνωστός διεθνώς. Οπότε γι' αυτό θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Οι, οι οικολόγοι αυτό θέλουν, μια νότατη αρχή για την διαφάνεια και υπό την αιγίδα του οποίου να βρίσκονται όλοι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και ανισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους. Θέλω επίσης να σας διηγηθώ και κάτι. Είμαι 10 χρόνια εδώ ευρωβουλευτής και έχω δει πολλά. Για τη διακριτική ευχέρεια των εμπειρογνωμόνων. Εγώ ασχολούμαι με τα πυρηνικά, κατά των πυρηνικών βέβαια. Έχουμε την συνθήκη Ευρατόμ. Είμαι συγγήτρια για τη ραδιενέργεια. Θέλω να δω τους εμπειρογνώμονες της ε, Eurotom και μου λένε δεν μπορούμε να σας δώσουμε τα ονόματά τους, γιατί αν σας τα δώσουμε μπορεί να υποστούν συνέπειες. Ε, αυτό είναι καινούριο. Νέο φρούτο. Απαράδεκτο. Στον Οργανισμό Υγείας, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όταν υπήρξε το σκάνδαλο εκεί, οι διάφοροι υπεύθυνοι μου είπαν δεν μπορούμε να σας δώσουμε το όνομα των εμπειρογνωμόνων γιατί κινδυνεύουν να γίνουν θύματα επιθέσεων. Οπότε... Πώς είναι δυνατόν οι πυρογνώμονες αυτοί που ήταν πυρογνώμονες γιατί τη γρήπη δεν μπορούν να έρθουν εδώ να μας τα πούν από πρώτο χέρι. Και τώρα για την Εύσα. Όταν λέτε και το καταλαβαίνω πολύ καλά. Μιλάτε για τη σύγκρουση φερόντων. Ωραία, δεν πιστεύετε ότι εμείς οι ευρωβουλευτές θα μπορούσαμε να σας δώσουμε παραπάνω πόρους αν έχουμε καλούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι να είναι μισθωτοί στην ΕΦΣΑ για μία περίοδο 5-6 ετών. Οπότε πραγματικά αυτό που κάνουν να είναι πραγματογνωμοσύνη. Γιατί τελικά τι έγινε και με τη γλυφοσάτη. Δεν είδατε το copy-paste της γερμανικής υπηρεσίας. Λοιπόν, δεν είδατε τίποτα ή δεν καταλάβατε τίποτα ή δεν θελήσατε να δείτε. Ε, καταλαβαίνετε ότι το θέμα των εμπειρογνωμόνων στην ΕΦΣΑ είναι κάπως περίεργο. Οπότε, ίσως θα ήταν καλύτερα να έχουμε μια υπηρεσία με πραγματικούς εμπειρογνώμονες που πληρώνουμε εμείς, παρά να φωνάζουμε εμπειρογνώμονες απ' έξω για το ένα και για το άλλο. Και η πραγματογνωμοσύνη που θα παρουσιάζεται να είναι πραγματική, αυθεκτική, είτε πρόκειται για χημικούς παράγοντες, είτε πρόκειται για φάρμακα, είτε πρόκειται για οτιδήποτε να πληρώνονται αυτοί οι εμπειρογνώμονες, βεβαίως, από την Ευρώπη, από εμά και όχι να είναι εξωτερικοί που δεν ξέρουμε από πού μας έρχονται και τι πρεσβεύουν. Είναι από τις χώρες μέλη, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν ε, συγκρούσεις συμφερόντων. Και τέλος, όταν πήγα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Έρευνα για τον Καρκίνο, είδα ότι ήταν πολύ καλό όταν ε, δηλώνανε και εμφανιζόντουσαν στο διαδίκτυο οι δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Γιατί καμιά φορά μπορεί κάποιος εμπειρογνώμονας να μην το δήλωνε, ναι, αλλά ο κόσμος τα έβλεπε αυτά τις δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και κάτι δεν πήγαινε καλά, το έλεγε. Καλό θα ήταν λοιπόν αυτές οι δηλώσεις ε, συμφερόντων να αναφέρονται και να ανεβάζονται στο διαδίκτυο. Αυτό ήθελα να πω. Η κυρία Γκρέσλε τώρα. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και χαίρομαι που μπορώ να πάρω το λόγο. Εμείς ε, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού πραγματικά έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτούς τους ε, φορείς και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργούν. Δεν ε, λειτουργήσαν πάντα τόσο καλά. Όταν υπάρχουν ανομαλίες και προβλήματα επεμβαίνει και το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, υπάρχουν ε, φορείς, υπάρχουν οργανισμοί και υπηρεσίες που δεν έχουν πολλά χρόνια ύπαρξης. Και βεβαίως δεν υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα, αλλά σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε υπηρεσίες όπου ο έλεγχος ε, η σύγκρουση, για τη σύγκρουση συμφερόντων γίνεται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο βάση κάποιων ενιαίων διαδικασιών. Από την άλλη, μην ξεχνάτε ότι οι οργανισμοί αυτοί δεν έχουν ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργίας, δεν είναι ομοιογενείς και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργεί ο κάθε οργανισμός για να καταλάβουμε ακριβώς πώς ε, μπορεί να μιλήσει κανείς για σύγκρουση συμφερόντων. Παράδειγμα, το, το θέμα των ε, αποσπασμένων εμπειρογνωμόνων, αυτών που εργάζονται εκτός της, ε, σε μια άλλη χώρα, οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται και βεβαίως Καταλαβαίνετε ότι οι εμπειρογνώμονες και η εργασία τους δεν μπορεί να περικλείεται από μια γενικευμένη δυσπιστία. Και θα πρέπει κάθε φορά να είναι σαφείς οι κανόνες, δημοσίοι κανόνες και να τηρούνται κάποιες διαδικασίες και κάποια μέθοδος εργασίας. Νομίζω ότι αν διαβάσετε προσεκτικά τα έγγραφα τους κανονισμούς όλων, που πολλές φορές ε, φτιάχνονται, προετοιμάζονται και μετά κλείνονται σε ένα ντουλάπ και κανείς πια δεν τις κοιτάει, θα καταλάβετε ότι ο έλεγχος υπάρχει. Τουλάχιστον η δική μου εμπειρία, η εμπειρία της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού, δείχνει ξεκάθαρα ότι το σύστημα λειτουργεί σε γενικές γραμμές για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εμπειρογνώμονες αυτοί, οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να δουλέψουν χωρίς να τους υποψιάζονται όλοι ότι πραγματικά να δείξουμε ότι υπάρχει και κάποια εμπιστοσύνη έτσι ώστε αυτή η περίοδος παραδείγματο χάρη που έχει προβλεφθεί η διετία μετά το τέλος της σύμβασής τους κατά την οποία δεν πρέπει να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων να μπορεί να ε, λειτουργήσει χωρίς να υπάρχει μια γενικευμένη δυσπιστία πριν και μετά από αυτό. Ο κύριος Γιάρ, αλλά γρήγορα παρακαλώ, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Ναι, μια φράση. Εγώ ήθελα να κάνω την ίδια παρατήρηση και την ίδια ερώτηση με τη συνάδελφο Γκρέσλε. Η εμπειρογνωμοσύνη που αφορά την ΕΦΣΑ με ξάφνιασε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, πραγματικά, για να προσλάβει η ΕΦΣΑ έναν εμπειρογνώμονα τα έγγραφα, τα δικαιολογητικά, η έρευνα που πρέπει να γίνει πραγματικά είναι πάρα πολύ βαριά. Ναι για τη διαφάνεια, αλλά η ερώτησή μου είναι υπάρχουν πραγματικά ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Δεν ξέρω, για πείτε μου. α είμαστε προσεκτικοί με τον ορισμό των ενιών. Τι ακριβώς εννοούμε ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων, παραδείγματος χάρη. Όχι, δεν θα μιλήσει κανένα άλλο. Καμία άλλη ερώτηση. Αν έχετε κάτι να πείτε, σύντομα να το ακούσουμε. Θα ξεκινήσω με το ερώτημα που άκουσα για την αίμα, για τον Οργανισμό Οργανισμό Φαρμάκων. Είναι ένας οργανισμός με νέο καταστατικό. Ε, σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία ε, υπάρχει αυτό το νέο ε, καταστατικό. Ε, ένας διευθυντής είναι ένας έκτατος υπάλληλο, έτσι. Ε, και όταν μιλούσα για συστήματα ε, κυρώσεων, ε, αυτά, αυτά ισχύουν και για τους επιτρόπους και για τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου και για τους διευθυντές κτλ. Τώρα για το προσωπικό, ε, τον έκτατο διευθυντή, προσωρινό διευθυντή όπως ο διευθυντής της ΕΟΦ, του ΕΟΦ, εδώ είχαμε μια βελτίωση του καταστατικού. Ε, ένας ε, διευθυντής δεν μπορεί για ένα χρόνο να ασκήσει, να κάνει λόμπι ή να συμμετέχει σε ομάδα υπεράσπιση φερόντων. Και οι κυρώσει ε, μπορεί να είναι μέχρι και πειθαρχικέ και θα μπορούσαν δηλαδή να του καταργήσουν, να του μειώσουν πάρα πολύ τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Ε, μπορούμε να πάμε ακόμα πιο μακριά. Γιατί οποιοδήποτε υπάλληλο ή πρώην υπάλληλο έχει κάποιες ευθύνε απέναντι στην, στον οργανισμό του. Υπάρχουν κυρώσει λοιπόν και σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία βελτιώσαμε πάρα πολύ τον έλεγχο. Ευχαριστώ. Για τη σύγκρουση συμφερόντων για τους συμπειρογνώμονες είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή και αυτό που εννοούσα είναι ε, να υπενθύμισε αυτό που ακούσαμε από την Ευρωπαία Δημεσολαβήτρια, η οποία είπε ότι χρειάζεται να, έχει να υπάρχει προσωπικό που έχει δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να κάνει μια κατηγοροποίηση. Κάποιο ο οποίο απασχολείται πλήρω, που είναι υπάλληλο και έχει δουλέψει στο παρελθόν στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι ένα πράγμα. Και ένα άλλο πράγμα, ένα εμπειρογνώμονα που δεν είναι υπάλληλο όμω, απλώ έχει κάνει μια δουλειά ad hoc, α πούμε, ε, και δίνει συμβουλές στον οργανισμό. Αυτός ο εμπειρογνώμονα μπορεί να έχει δουλέψει στο παρελθόν στον ιδιωτικό τομέα. Και για την ΕΦΣΑ ε, υπάρχουν ε, κανόνες για μια περίοδο που δεν μπορεί να κάνει να δουλέψει πούμε, για την ΕΦΣΑ ο εμπειρογνώμονα. Αν έχει δουλέψει πούμε, για τον ιδιωτικό τομέα, για μια ΜΚΟ, επί δύο χρόνια δεν μπορεί να δώσει συμβουλές, δεν μπορεί να δουλέψει ω εμπειρογνώμονα στην ΕΦΣΑ. Cooling off period λέγεται αυτό. Και Εάν, ας πούμε, ε, υπάρχουν και ιδιωτικές μελέτες ε, ε, οι οποίες υποβάλλονται μέσα σε ένα ντοσχέ από το, την ιδιωτική εταιρεία στον οργανισμό, εδώ έχουμε ένα λεπτό σημείο. Ποιος χρηματοδοτεί αυτές τις μελέτες. Όταν, ας πούμε, ο κλάδος, μια ιδιωτική εταιρεία ζητάει μια άδεια, ας πούμε, και υποβάλλει αυτό το ντοσχέ. Υπάρχει ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα για να ενισχύσει ε, την δημόσια χρηματοδότηση τέτοιων μελετών. Επίσης αναγνωρίζεται ότι δεν είναι δυνατό να έχουμε χρηματοδότηση 100% με δημόσιο χρήμα, γιατί ας πούμε και τα πανεπιστήμια από μόνα τους. Δεν μπορούν να κάνουν όλες τις απαραίτητες μελέτες που χρειαζόμαστε. Έχουμε ένα σύστημα, δηλαδή, όπως συχνά ε, οι εταιρείε πληρώνουν τα πανεπιστήμια για μία μελέτη και εκεί υπάρχει τότε σύγκρουση συμφερόντων. Συμφωνώ μαζί σας ότι ιδανικά θα έπρεπε να έχουμε ε, δημόσιο έλεγχο των ε, μελετών. Εγώ το λέω σαν ακαδημαϊκό αυτό. Είναι προσωπική γνώμη. Αλλά γιατί το γεγονό ότι υπάρχουν και δημοσιονομικοί περιορισμοί, αυτό το καθιστά αδύνατο. Υπάρχει και μια πρόταση Κομισιόν αυτή τη στιγμή για να ενισχύσουμε τον έλεγχο των μελετών για το πώς δηλαδή, σχεδιάζονται οι μελέτες, να ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα από τον κλάδο ε, που θα πρέπει να βάζει στη μελέτη για να υπάρχει μεγαλύτερο έλεγχο των μελετών, να υπάρχει και δημόσια διαβούλευση και αξιολόγηση από μότιμους ε, των μελετών. Και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός να εξετάζει όλες τις μελέτες, όχι μόνο τη μελέτη που παρήγγειλε, ας πούμε, ε, που ετοίμασε η βιομηχανία για το συγκεκριμένο θέμα. Όλε τι σχετικέ μελέτε είναι υποχρεωμένο ο οργανισμό να τι μελετάει. Είναι δύσκολο να υπάρξει μια καλή ισορροπία του δημοσίου με το ιδιωτικό συμφέρον. Χρειαζόμαστε περισσότερο έλεγχο επί των μελετών, σίγουρα. Αυτό θα δούμε πώς θα το καταφέρουμε χάρη στη τελευταία πρόταση Κομισιόν. Θα ήθελα πριν να πριν απαντήσει ξανά ο κάποιος ομιλητή να ξαναπάρει το λόγο η κυρία Χωζιέ. Έχω μια ερώτηση που αφορά όλους σας και όλα τα θέματα που σχολιάσατε και που αφορά πολλούς οργανισμούς. Συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο με βάση μιας, μια πρόταση της Κομισιόν για την προστασία των καταγγελόντων, των whistleblowers. Όλες οι ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες θα πρέπει να θετήσουν αυτούς τους προστατευτικούς κανόνες για αυτούς τους καταγγέλλοντες. Αλλά που δεν ισχύουν για τον κανονισμό υπηρεσιακή κατάσταση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Έχουμε ξεχωριστή διαδικασία εδώ. Η ευρωπαϊκή δημοσια... δημοσια... υπαλληλία με βάση αυτόν τον κανονισμό, εκτός και αν αλλάξει ε, τα επόμενα δύο χρόνια, ε, αυτό τόσο ο κανονισμός λοιπόν θα προστατεύει λιγότερο τους πιθανούς καταγγέλλοντες. Όταν έχουμε σύγκρουση συμφερόντων, συχνά ε, έχουμε πληροφορίες εκ των ένδο που μας αποκαλύπτουν διάφορα πράγματα. Θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας άποψη μια και ξέρετε περισσότερα, μήπως χρειαζόμαστε περισσότερη προστασία ε, για αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ στα, στα νοσιακά όργανα, για να μπορούν να καταγγέλουν, να φύγουν τα κακοσκήμενα, ας πούμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την επιπλέον προστασία για, τους, ε, για την ευρωπαϊκή δημοσιοπαλληλία. Μήπως χρειάζεται ενδεχομένω να προσφύγουμε σε εξωτερική αρχή. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι χρειαζόμαστε περισσότερη προστασία. Ποια είναι η γνώμη σας. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν προβλέπονται με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν, όπως σας είπα, τα επόμενα δύο χρόνια. Κύριε Ντέτκεν, θέλετε να αντιδράσετε σε κάποια ερώτηση σε αυτή ή σε κάποια άλλη. Να απαντήσω στην κυρία Γιβαζή. για το θέμα της ανεξαρτησίας. Η ΕΦΣΑ ως τεχνική υπηρεσία πρέπει να εφαρμόσει τους κανόνες που την αφορούν. Και έχουμε συγκεκριμένους κανόνες τους οποίους σεβόμαστε. Ε, υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για τους δικούς μας εμπειρογνώμονες από τους άλλους α, οργανισμούς. Ε, αυτό το θέμα ενδεχομένως πρέπει να το ξαναδεί ο νομοθέτης, οι νομοθετικές αρχές. Πάντως, εμείς σεβόμαστε τους κανόνες που μας αφορούν. Τώρα, από πού βρίσκουμε εμπειρογνώμονε. Ε, το σύστημα είναι συγκεκριμένο για την ΕΦΣΑ. Εμεί πιστεύουμε ότι τα πάει καλά για μα, αλλά αν το σύστημα ε, για τι απολαυέ του θα πρέπει να αλλάξει, αυτό θα πρέπει να γίνει με πρωτοβουλία του νομοθέτη. Δεν θα αλλάξουμε εμεί του κάνονες που μα αφορούν. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, θέλω να επαναλάβω ότι η δήλωση συμφερόντων τη ΕΦΣΑ ε, είναι δημόσια έγγραφα, οι δηλώσει όλε είναι δημόσια έγγραφα και τα κριτήρια ελέγχου επίσης είναι δημόσια. Ε, εμείς ε, αυτές τις δηλώσεις τις βάζουμε στην ιστοσελίδα μας. Δεν τη βάζουμε σε διάφορα κινητά κτλ. Για τους εμπειρογνώμονες και τα προβλήματα που είπατε. Το 2017 ε, υπήρξαν νέοι κανόνες, ούτω ώστε η ΕΦΣΑ να ελέγχουν τους εθνικούς εμπειρογνώμονες ε, για το, την περίπτωση της αναθεώρησης του μηχανισμού των φυτοφαρμάκων. Για τους καταγγέλλοντες, ας απαντήσει ο συνάδελφος από την Κομισιόν. Για την ε, υπηρεσία, το δικό μου οργανισμό, θέλω να σας πω ότι έχουμε κανόνες εναρμονισμένους για όλους τους οργανισμούς για το πώς θα προστατεύσουμε τους καταγγέλλοντες, ε, τα δικαιώματα που έχουν οι καταγγέλλοντες και τους τελευταίους 12 μήνες η ΕΦΣΑ ε, υιοθέτησε αυτούς τους κανόνες και το έκαναν και οι άλλοι οργανισμοί. Αυτή τη στιγμή ε, δημοσιεύτηκαν από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Επομένως, εμείς εφαρμόζουμε αυτά τα στοιχεία του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Αυτά. Άλλα σχόλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί βλέπετε ότι η υπηρεσιακή κατάσταση είναι κάτι βελτιωμένο και προβλέπει ήδη μεγάλη προστασία για τους καταγγέλλοντες συναδέρφους και είναι κάτι που πριν το νέο καταστατικό είχαμε προβλέψει προστασία για τους καταγγέλλοντες. Για να σας πω δηλαδή ότι έχουμε ήδη ένα σχέδιο. Δεν απαντήσατε στην ερώτησή μου όμως, λέει κύριε Ριβαζή. Αν θεωρείτε λογικό να μην μαθαίνουμε τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων. Την Επιτροπή ρώτησα γι' αυτό. Γιατί. Γιατί δεν μπορέσαμε να μάθουμε τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων της ε, Euratom, για παράδειγμα, ή άλλων. Ξέρετε γιατί. Δεν μπορώ να απαντήσω σε πράγματα που ξεπερνάνε τις αρμοδιότητές μου. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η προστασία δεδομένων, δηλαδή ότι υπάρχει κάποια ισορροπία ανάμεσα στη διαφάνεια και την προστασία δεδομένων. Και υπάρχει και απόφαση στη, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση Bayer Lager που ακριβώς προσπαθεί να πετύχει αυτή την ισορροπία. Και ακόμα κι αν ε, έβαλε σε δοκιμασία αυτή την ισορροπία, πάντα έλεγε ότι η προστασία του ατόμου είναι πολύ σημαντικό και το λαμβάνει υπόψη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και λέει ότι αυτά τα δικαιώματα υπερέχουν. Λυπάμαι να πρέπει να κλείσουμε αυτό το εργαστήριο τώρα, λέει ο Προεδρεύων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τι σκέψεις σας που μοιραστήκατε μαζί μας για ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα και που σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα μας απασχολήσει για μήνες και για χρόνια ακόμα. Ευχαριστώ τους ομιλητές και όλους όσοι πήραν το λόγο που μας βοήθησαν. Η Επιτροπή ελέγχου προπολογισμού και νομική επιτροπή στις 15 Απριλίου επίση θα συζητήσουν το θέμα των διαδικασιών ορισμού στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. 15 Απριλίου. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Και αυτούς που είναι ικανοποιημένοι πλήρως από τα συμπεράσματα και αυτούς που δεν είναι ικανοποιημένοι πλήρως από τα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πολύ η πρόεδρος. Ωραία. Don't worry, be happy. Αυτά ουσιαστικά μας είπε ο Προεδρεύων. Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ όλοι, Πρόεδρος, για τη συμμετοχή σας εδώ. Ελπίζω να διαφωτιστήκαμε λιγάκι, ακόμα και αν μπήκαν πολλά ερωτηματικά. Θα είμαστε σε επαφή. Και σίγουρα είναι ένα θέμα που θα επανέλθει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και στην επόμενη θητεία. Συνεχίζουμε και πάμε τώρα στην επόμενη αναφορά μας αναφορά T28 με 12 υπογραφές για την έκθεση ε, εργαζομένων στη Γεωργία σε παρασιτοκτόνα. Ο κύριος Σέρζ Λεκεό είναι ο αναφέρον και ο κύριος Λοραντουριού που είναι εδώ θα πάρουν το λόγο. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εν ονόματι όλων των μελών της ομάδας μας, ε, σας ευχαριστώ για την ε, στήριξη στα θύματα ε, των φυτοπαρμάκων της εταιρείας Τρισκαλία και σας ευχαριστώ που μας προσκάλεσατε σήμερα. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που ήρθαν τον περασμένο Ιούνιο στην Βρετάνη και που τα συναντήσαμε. Αυτή η έκθεση είναι ένα βαρύ κατηγορό. Λέει όχι μόνο ότι η χώρα μας, η Γαλλία, δεν μειώνει τη χρήση των φυτοφαρμάκων, αλλά λέει επίσης ότι, κάτι που είναι πολύ σοβαρό, ότι το Υπουργείο Γεωργίας γνωρίζει ότι το σχέδιο μείωσης των φυτοφαρμάκων καθορίζει στόχους που δεν θα μπορέσει να εκτοπίσει. Ποιο κοροϊδεύει ποιον. Από την άλλη, η έκθεση ε, διατρανώνει το 70% των επιθεωρήσεων που γίνονται στου λιανέμπορου και διανομή ε, φυτοφαρμάκων τη Βρετάνη δείχνουν ότι τα επικίνδυνα προϊόντα δεν αποθηκεύονται μακριά από τα άλλα προϊόντα σε συγκεκριμένε αποθήκε στην περιοχή τη Βρετάνη. Οι μισθωτοί λοιπόν, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να γνωρίζουν τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται. Ακριβώ γι' αυτό ε, έγιναν σοβαρές, ε, υπήρξαν σοβαρέ δηλητηριάσει στου εργαζόμενου του Τρισκαλιά που δεν έχουν καμία προστασία. Τι θα κάνει η Γαλλία απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Ζητούμε από την Επίτροπο Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων, την κυρία Τίσεν, να κάνει μια ε, αποστολή ελέγχου στη Βρετάνη. Ο συνάδελφός μου θα συνεχίσει την παρουσίαση. Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, βουλευτές, ζητούμε από την Επιτροπή Αναφορών να αποστείλει μια επίσημη προειδοποίηση προς τη Γαλλία για να σεβαστεί τους κανονισμούς για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Γνωρίζουμε και έχουμε συνέστηση ότι η έκθεση ελέγχου ε, αφορούσε μόνο ένα τμήμα του προβλήματος που ε, θέτει η αναφορά μας. Σημειώσαμε ότι η Επίτροπος, ο Επίτροπος Υγείας, ο κ. Ανδριουκάητης, θέλει να δώσει συνέχεια μετά τις πληροφορίες που του διαβιβάσαμε το Σεπτέμβριο του 2018. Θα θέλαμε να μάθουμε πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η έκθεση. Επίσης, εκφράζουμε την ε, θλίψη μας που η Γαλλία μέχρι στιγμής ε, παρέμεινε σιωπηλή απέναντι στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι απαράδεκτο τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πέφτουν σε κοφεύοντα ότα στη Γαλλία. Είμαστε θύματα και αντιμετωπίζουμε και εμείς την ίδια σιωπή από τις αρχές. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί όμως. Σήμερα η ομάδα μας ε, έχει, που έχει δημιουργηθεί και εδώ και τρία χρόνια έχει 300 μέλη και λαμβάνει δύο νέες κλήσεις από θύματα τη βδομάδα από την τελευταία επίσκεψη στην Επιτροπή Αναφορών, την επίσκεψή μας, τρία από τα μέλη μας πέθαναν λόγω της αρρώστιας τους. Θα θέλαμε επιτέλους, κυρία Πρόεδρε, να μας ε, διασφαλίσετε ότι η αναφορά μας δεν θα εξαφανιστεί όταν αναλάβει τα καθήκοντά της η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσεχώς. Σας ευχαριστώ. Εγώ. σα ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Θα επανέλθω σε κάποια από αυτά τα σημεία και επανέρχομαι στην κατάσταση πριν την δημοσίευση της έκθεσης για τη Γαλλία, το σχέδιο δράσης, τις συστάσεις μας, καθώς και τις ερωτήσεις και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας. Υπάρχουν ε, συστάσεις, αξιολογήσαμε σειρά δράσεων που έχουν ε, προταθεί και μέτρα τα οποία έχουν αξιολογηθεί σαν μη ικανοποιητικά. Ζητήσαμε περισσότερες πληροφορίες. Το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι δεν καλύπτεται το φάσμα των μέτρων από την μέχρι τώρα πολιτική δράση και ότι θα πρέπει να υπάρξει και νέα αξιολόγηση. Οι δικές μας συστάσεις ουσιαστικά παρακολουθούνται από τους εμπειρογνώμονες ε, των ε, δικών μας γραφείων και περιμένουν τις ε, απαραίτητες απαντήσεις. Βεβαίως η έκθεση αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί και να υπάρξει παρακολούθηση και περαιτέρω επεξεργασία. Το Υπουργείο Εργασίας της Γαλλίας θα πρέπει να δώσει διευκρινήσεις και απαντήσεις σε αναπάντητα ερωτήματα. Όσον αφορά τα φυτοφάρμακα, τα εντομοκτώνα και τη χρήση τους, έχουμε μια συγκεκριμένη ποσότητα στοιχείων πληροφοριών. Κάποια από τα ερωτήματα, επαναλαμβάνω, παραμένουν αναπάντητα. Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας είναι ότι περιμένουμε διευκρινήσεις, περιττέρω διευκρινήσεις από μέρους των γαλλικών αρχών. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Συνάδελφοι, θέλετε να πάρετε το λόγο. Κυρία, κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν θέλω να χαιρετήσω τους αναφέροντες που εκπροσωπούν δύο συλλογικά όργανα που πραγματικά εδώ και χρόνια μάχονται για να γνωριστεί η ευθύνη του εργοδότη. Και επειδή δεν έχει ακόμα επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αναφέρονται σήμερα στις αρχές αυτές που θα έπρεπε να διασφαλίσουν την ε, αναγνώριση της ευθύνης του συγκεκριμένου εργοδότη. Δυστυχώς δεν είναι η μόνη αναφορά, η μόνη υπόθεση που ουσιαστικά περιγράφει αυτές τις τραγικές προσωπικές υποθέσεις. Άτομα που προσπαθούν ε, να βρουν το δίκιο τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εγγυημένα από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ε, δικαιώματα. Πρόκειται για διαδικασίες επίπονες, χρονοβόρες, ε, κάτι που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Πρόκειται για μια δικαστική διαδικασία μέσω των ε, μέσων ζητούν αποζημίωση μια τόσο χρονοβόρα διαδικασία που πολλές φορές τα θύματα δεν είναι πλέον στη ζωή για να λάβουν τις αποζημιώσεις τους. Και σίγουρα θα πρέπει να αλλάξει και η διαδικασία εφαρμογής ε, της ε, εν λόγω νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ για όλα όσα έχετε κάνει και ελπίζω ότι θα υπάρξει μια συλλογική απάντηση και αντιμετώπιση αυτής της ε, υπόθεσης. Η συγκεκριμένη περίπτωση ενδεχομένως είναι εμπεριστατωμένη περισσότερο από άλλες και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μία πάρα πολύ ε, εμπεριστατωμένη έκθεση που αφορά την έλλειψη ελέγχων όσον αφορά τη χρήση των ε, φυτοπαρμάκων νέοι έλεγχοι, νέα στοιχεία, μας ανέφερε η Επιτροπή. Εγώ είχα την εντύπωση ότι αν ένα κράτο μέλος δεν τηρεί συγκεκριμένες οδηγίες, ξεκινάει η διαδικασία επί παραβάς. Και εδώ βλέπουμε ότι παρόλο που δεν με χαροποιεί το γεγονός ότι η ίδια μου η χώρα παραβιάζει την οδηγία αυτή, περίμενα να έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Μπορείτε λοιπόν να μου πείτε και απευθύνομαι προς την Επιτροπή ε, πώς μπορεί να γίνει συγκεκριμένη αξιολόγηση και πώς γίνεται να παραβιάζεται συγκεκριμένη οδηγία και να μην ξεκινάει διαδικασία προσφυγής που να καταλήξει σε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Κάτι που θα είχε μια συγκεκριμένη επίπτωση για την εν λόγω διαδικασία αναφοράς ε, στην περίπτωση που θα υπήρχε καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα ήταν πολύ πιο εύκολο να αναγνωριστεί η ευθύνη του εργοδότη από μέρους των εταιριών όπως τη συγκεκριμένη εταιρεία στη Γαλλία, της Τρισκάγια. Η κινητοποίηση των ε, συγκεκριμένων ε, Γάλλων πολιτών βασίζεται σε μια διαδικασία τόσο χρονοβόρα που δεν μπορούμε πια να περιμένουμε κι άλλο. Είναι μια παράδεκτη κατάσταση και τα πλήγματα είναι εξαιρετικά σοβαρά. Η κατάσταση από υγειονομικής απόψεως είναι πάρα πολύ σοβαρή, απαράδεκτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ε, πραγματικά κάνει ένα πολύ ενθαρρυντικό βήμα με αυτόν τον έλεγχο, αλλά πραγματικά θα πρέπει να εμποδίζουμε αυτές τις ε, καταστάσεις και εμείς συγκεκριμένα να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε χημικές ουσίες όπως τα φυτοφάρμακα, τα εντομοκτώνα, την αρχή της πρόληψης, μια έννοια που μας απασχόλησε πολλές φορές εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά συγκεκριμένα για αυτήν εδώ την αναφορά δεδομένων των νέων στοιχείων πραγματικά θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και να στηρίξουμε τους αναφέροντες έτσι ώστε να μπορέσει να αναγνωριστεί ε, η παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι όντως παράδεκτη αυτή η κατάσταση και δικαιολογείται πλήρως η στήριξη που θα πρέπει να δώσουμε. Θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει όλοι να εμφαρίνουμε την ε, Επιτροπή. Εγώ σαν πολύ ευαισθητοποιημένο σε θέματα γεωργικά, ε, σαν Γερμανός, πιστεύω ότι όλες αυτές οι ουσίες, η χρήση τους, η αρνητικές επιπτώσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με εξαιρετική σοβαρότητα και αυστηρότητα. Νομίζω λοιπόν πολύ συγκεκριμένα ότι η Γαλλία εδώ θα πρέπει πραγματικά να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό όπως και πολλές άλλες χώρες του δυτικού ανεπτυγμένου κόσμου και ζητώ από την Επιτροπή και γι' αυτό αλλά και για άλλα κρατημέλη να εφαρμόσει τις διαδικασίες. Και όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, πρόκειται για επικίνδυνες ουσίες, πρόκειται για χημικές ουσίες, τα εντομοκτώνα, τα φυτοφάρμακα, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με πολύ μεγάλη προσοχή. Και τα κράτη-μέλη νομίζω ότι προσπαθούν να παρεκκλίνουν και εμείς ε, εδώ στις Βρυξέλλες δεν καταδικάζουμε, δεν κρίνουμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και αυστηροί. Ευχαριστώ. Η κυρία Ριβασί. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω να σας πω ευτυχώς που υπάρχει αυτή η Επιτροπή Αναφορών, γιατί επιτρέπει να έρχονται εδώ οι άνθρωποι αυτοί, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι καταγγέλνουν μια δυσλειτουργία που υπάρχει στη Γαλλία, θα μπορούσε να ήταν και αλλού. Θέλω να επενθυμίσω μερικά πράγματα για τη Τρασκαλία, που είναι ένας μεγάλος γεωργικός συνεταιρισμός, ο πιο μεγάλος στην Βρετάνη, με 4.800 υπαλλήλους και 6.000 αγρότες. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια μικρή επιχείρηση, πρόκειται για μια τεράστια επιχείρηση, η οποία δηλητηρίασε μισθωτούς, αλλά και αγρότες που χρησιμοποιούν τα φυτοφάρμακα αυτά. Πήγε λοιπόν η Επιτροπή, είδε την κατάσταση επιτόπου και η έκθεσή σας τι λέει. Δίνει πληροφορίες που δείχνουν ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και προς τους ε, υπαλλήλους και προς τους ε, συνεργαζόμενους ότι δεν υπάρχει αρκετός έλεγχος και εποπτεία με αποτέλεσμα τη δηλητηρίαση των υπαλλήλων. Και ποια είναι η απάντηση τρισκαλιά? Ε, όταν αρρωσταίνουν τους απολύει. Και τη μόνη λύση που βρήκαν τώρα είναι ή να πεθάνουν ή να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να αποζημιωθούν. Η κατάσταση είναι τραγική λοιπόν πιστεύω. Μία ερώτηση έχω στην Γενική Διεύθυνση υγεία. Λέτε ότι περιμένουμε τις απαντήσεις τη Γαλλία. Μάλιστα. Αλλά κοιτάξτε, να έρχονται οι ευρωεκλογέ στις 26 Μαΐου. Επίγει να έχουμε τη δεύτερη έκθεσή σα ακριβώ για να πάμε στη Γαλλία και να πούμε «Κοιτάξτε, αν δεν απαντάτε, ε, πρέπει να του βάλουμε ένα όριο. Θα σα ε, προειδοποιήσουμε». Παραβιάστε την οδηγία και είναι σημαντικό για όλους τους εργαζόμενους για όλους τους συνδικαλιστές. Γιατί αν εσείς προειδοποιείτε τη Γαλλία και πείτε ότι παραβιάζει κάποιους νόμους η Γαλλία, τότε θα αναγκαστεί η επιχείρηση να προβαίνει στην ενημέρωση που πρέπει προς εργαζόμενους κτλ. Γιατί εδώ αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, αυτό. Έπειτα, στην έκθεση λέτε επίσης ότι όλο το θέμα υγείας των εργαζομένων έχει, είναι αρμοδιότητα της Επιτρόπου Τίσεν. Εσείς κύριε Πρόεδρε μπορείτε να ζητήσετε από την Επίτροπο να έρθει εδώ σε ακρόαση ώστε να συζητήσουμε μαζί της όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία στην εργασία και να υπάρξει και έλεγχος επιτόπου. Οι υπεύθυνοι δηλαδή της Επιτροπής μας να πάνε επιτόπου και να ελέγξουν την κατάσταση και να κάνουν τις ερωτήσεις που θέλουν γιατί το θέμα δεν είναι μόνο η χρήση των φυτοφαρμάκων αυτών, είναι και η αποθήκευση αυτών των υλικών στην επιχείρηση. Να λοιπόν, διάφορες λύσεις και πραγματικά μόνο η δικιά μας Επιτροπή μπορεί να καταγγείλει τέτοιες δυσλειτουργίες στις χώρες μέλη. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ωραία. Θα δώσω το λόγο και πάλι στους αναφέροντες. Τον κύριο Λεκεό πρώτα για λίγα λεπτά παρακαλώ. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Γιατί και εμείς έχουμε περιορισμό στο χρόνο. Ε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, πράγματι η έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας έχει να κάνει με την 128 του 2009 οδηγία. Και πράγματι η ΣΕ 1 αναφέρεται ειδικά στην προστασία των ε, μισθωτών που χειρίζονται ε, φυτοφάρμακα. Ευχαριστούμε πολύ για τις παρεμβάσεις των ε, Ευρωβουλευτών μελών της Επιτροπής αυτής αναφορών που ζητούν η Γαλλία να δεχτεί επίσημη προειδοποίηση ότι θα υπάρξει προσφυγή στο δικαστήριο. Δεν υπάρχει καμία δικαστική απόφαση στο ποινικό. Δύο φορές στο Σαμπριέ το δικαστήριο εξέτασε την υπόθεση. 40 μάρτυρες πήγαν στη δίκη. Δεν υπήρξε εξέταση. Οπότε η οι υπάλληλοι είναι πολύ απογοητευμένοι, γιατί όπως λέει η κυρία Ριβαζή, δηλητηριαστήκαμε σε μεγάλο βαθμό. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους. Οι αποζημιώσεις ήταν πάρα πολύ αδύναμες και πιστεύουμε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι αν δεν υπάρξει ποινική κύρωση, το θέμα μας δεν είναι να πάει κάποιος ε, στη φυλακή, το θέμα μας είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένα σημαντικό μήνυμα που θα βγει προς τα έξω. Γι' αυτό ζητάμε την ποινική καταδίκη, ώστε να φανεί ότι πράγματι φταίνε. Πρόεδρος, ωραία. Να συνοψίσω και τι θα κάνουμε στο μέλλον με την αναφορά αυτή. Πιστεύω και εγώ ότι είναι τρομακτικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε την έκθεσή της για τον έλεγχο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ αλλά δυστυχώς μία μόνο πρόταση αφορά την αναφορά μέσα στην εκθεσή σας αυτή και τους ελέγχους στους οποίους προβήκατε. Θα έπρεπε να υπάρχει μια χωριστή αξιολόγηση και μια χωριστή έκθεση, πιστεύουμε, για το θέμα της αναφοράς. Τι να κάνουμε λοιπόν, να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή, να ζητήσουμε γραπτή ενημέρωση με χωριστή αξιολόγηση του ελέγχου όσον αφορά την αναφορά και να στείλουμε ε, μια επιστολή στους Επιτρόπους Αντροκαΐτης και Μαρία Τάισεν και να τους ζητήσουμε να λάβουν υπόψη τους όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην αναφορά και που πιστεύω ότι δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη στην δικιά σας έκθεση. Και να στείλουμε επιστολή και στις γαλλικές αρχές μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας τους στις Βεξέλλες ενημερώνοντάς τους για το τι έγινε στην σημερινή συνάντηση και να τους ρωτήσουμε τι έκαναν και ιδιαίτερα τι δεν έκαναν για την ασφαλή χρήση των φυτοφαρμάκων. Επίσης θέλω να υπογραμμίσω ότι η αποζημίωση όποια και αν είναι, δεν φέρνει πίσω ανθρώπινες ζωές. Όσοι υπέφεραν όμως πρέπει να έχουν τη δυνατότητα κάποιας αποζημίωσης εξαιτίας της ζημιάς που τους έγινε, της βλάβης τους. Εντάξει, συμφωνείτε? Καλώς, ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους πάρα πολύ για όλα αυτά. Τώρα ερχόμαστε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Είμαστε στην παρουσίαση της μελέτης όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράχτες και τη ζημιά που κάνουν στην ανθρώπινη υγεία. Έχουμε εδώ πέρα διάφορους εμπειρογνώμονες. Την Μπάρμπαρα Ντεμινιέ πρώτα απ' όλα και την Ρέμι Σλάμα. Και σας παρακαλώ, έχετε το λόγο. Από εδώ αν συμφωνείτε με την ε, συνάδελφο Σάλμα αντιμετωπίσαμε τα επιστημονικά στοιχεία για τις επιπτώσεις των ενδοκρινικών διαταρακτών στην ανθρώπινη υγεία. Καταρχάς, σύγκρουση συμφερόντων. Δεν έχουμε οικονομική σύγκρουση συμφερόντων, να δηλώσουμε. Εγώ είμαι συνειδήτρια του Watch Frog, είναι μια εταιρεία η οποία εμπλέκεται στην ανάπτυξη τεστ για να εντοπίσει τους ενδοκρινικούς διαταράχτες και δεν πληρώνομαι για οποιαδήποτε δραστηριότητα που κάνω στα πλαίσια της εταιρεία αυτής. Λοιπόν, γιατί θα μιλήσουμε. Θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή στο ορμονικό ενδοκρινικό σύστημα, γιατί είναι τόσο ευαίσθητο στις ε, διαταραχές από τα χημικά θα μιλήσω για τις παρενέργειες στην υγεία που έχουν τεκμηριωθεί λόγω της συνεχούς ε, έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράχτες. Θα μιλήσω για το κόστος που έχουν ε, οι ενδοκρινικοί διαταράχτες, τα χημικά αυτά και ο κύριος Σάλμα θα ασχοληθεί με τον κανονισμό για τους ανδοκρινικούς διαταράχτες στην Ευρώπη και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη υγεία στην Ευρώπη. Ποια είναι τα επιστημονικά στοιχεία και γιατί οι ενδοκρινικοί διαταράχτες είναι τέτοιο μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Οι ορμόνες λειτουργούν, ε, δουλεύουν με πολύ μικρές ε, δόσεις, Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Το ενδοκρινικό ή ορμονικό σύστημα, ε, η στρογόνα, τεστοστερόνη, πάγκρεας, παγκρεας ε, δημιουργούν μια φυσιολογία σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του ανθρώπου, από τη σύλληψη μέχρι την, τα γυρατιά. Οι ορμόνες λειτουργούν σε πολύ χαμηλές δόσεις, νανομόρια είναι η συγκέντρωσή τους Και ο καλύτερος τρόπος για να σας το δείξω είναι να σας δώσω την εικόνα ότι αν πετάξουμε μία σταγόνα νερού σε μία ε, πισίνα ε, Ολυμπιακών διαστάσεων θα μας δώσει αυτή την ε, νανομοριακή συγκέντρωση. Αυτή είναι η συγκέντρωση των ορμονών στον ανθρώπινο οργανισμό. Μία ορμόνη η οποία λειτουργεί σε πολύ χαμηλές δόσεις είναι η ορμόνη του θηροειδού. Αυτή παράγεται από την, τον αδένα του θηροειδού, στη βάση του κλεμού, η θυροξίνη, αυτή η ορμόνη, έχει διαφορετικέ ε, λειτουργίε ανάλογα με την ηλικία του ατόμου. Στου ενήλικε θα ελέγξει τη θερμοκρασία του σώματο και το μεταβολισμό. Αλλά ελέγχει την δραστηριότητα του εγκεφάλου, την ε, διάθεσή μα, τη μνήμη μα, ε, το στρες, το πόσο συγκεντρωνόμαστε σε ένα θέμα. Στην φάση ανάπτυξη του εμβρίου είναι ακόμα πιο σημαντική η θηροξένη είναι ουσιαστική για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και την ανάπτυξη. Αν δεν υπάρχει θυροξίνη, θα επηρεαστεί η εξυπνάδα του αγέντου παιδιού και θα αυξηθεί ο κίνδυνος να έχει νευρολογικές ε, διαταραχές όπως ο αυτισμό. Ένα σαφές παράδειγμα είναι το πόσο παχής είναι ο φλοιός του εγκεφάλου του εμβρίου ε, έχουμε κάνει πειράματα σε 8 χρόνια παιδιά. Και αυτό συνδέεται με την συγκέντρωση της ηροξίνης ε, στην έγκυο μητέρα, στις αρχές μάλιστα της εγκυμοσύνης. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η, το πάχος επηρεάζεται από τη χαμηλή συγκέντρωση της ορμόνης ή την ψηλή συγκέντρωση. Ε, και η δεύτερη ιδέα είναι μία μη μονοτονική, μη γραμμική δηλαδή απόκριση στην ορμόνη. Δηλαδή δεν υπάρχει σχέση τόση δόση αυτή η απόκριση. Δεν είναι έτσι γραμμικά τα πράγματα δηλαδή. Το δεύτερο πράγμα το οποίο θα πρέπει να αναφέρω είναι Δεν βρίσκω αυτό που θέλω να σας πω. Πρέπει να αναφέρω ότι οι έγκυες γυναίκες ε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ. Ε, είναι μία ευαίσθητη περίοδος στην έκθεση και κάτι την ε, εγκυμοσύνη. Η έκθεση ενδοκρινικούς διαταράχτες μπορεί να επηρεάσει τρεις γενιές μετά. Προφανώς τη μητέρα την ίδια, το παιδί και την ανάπτυξη, το παιδί που αναπτύσσεται στη μήτρα, αλλά όχι μόνο και τα κύτταρα του παιδιού τα οποία αναπτύσσονται και που είναι αποφασιστικά για την παραγωγή σπέρματος και ο οαρίων και άρα επηρεάζουν τις μελλοντικές γενιές. Ένας ενδοκρινικός διαταράχτης ορίζεται λοιπόν ως μία εξωγενής ανθρωπογενής ουσία ή ένα μείγμα το οποίο αλλοιώνει τη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος, του ορμονικού συστήματος και επηρεάζει αρνητικά την υγεία στον οργανισμό. Τον ίδιο τον οργανισμό, στους απογόνους και στους μελλοντικού απογόνους. Ο ενδοκρινικός διαταράχτης λειτουργεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για την ανάπτυξη πολλών ασθενειών. Π.χ. μπορεί να τροποποιήσει την παραγωγή ορμονών, τη μεταφορά των ορμονών, να επηρεάσει τους ο, υποδοχής στους ιστούς. Αυτό είναι σημαντικό και αφορά και όλες τις μεγάλες ορμόνες. Δηλαδή, οι ενδοκρινικοί διαταράξεις επηρεάζουν όλες τις σημαντικές ορμόνες. Κατά συνέπεια, Η έκθεση στους διαταράχτες αυτούς ε, μέσω επιδημιολογικών μελετών και μέσω πειραμάτων ε, έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με αρρώστιες η έκθεση αυτή. Ε, επηρεάζει τους μεταβολικούς υποδοχείς που ελέγχουν το μεταβολισμό και άρα έχουν μεταβολικές ασθένειες, παχυσαρκία, ακόμα και διαβήτη τύπου 2 επηρεάζει την ορμόνη του θηροειδούς και δημιουργούνται νευρολογικές ε, αρρώστιες και χαμηλό IQ. Ε, αν επηρεάσει τις ε, στεροειδείς ορμόνες υπάρχει ε, υπογονιμότητα. επίσης μπορεί να δημιουργήσει καρκίνους σε ευαίσθητα, ευαίσθητους ιστούς όπως το στήθος, το μπροστάτι και στους όρχες. Η περίπτωση του καρκίνου του στήθους είναι πολύ σημαντικό παράδειγμα εδώ. Όπως και για άλλε μη μολυσματικέ αρρώστιες, ξέρουμε ότι ε, αποκτά κάνει καρκίνο του στήθους λόγω πολλών ας πούμε, παραγόντων. Ε, λόγω της, ε, του ιστορικού της γυ, γυναίκας, του αναπαραγωγικού ιστορικού της, κατά πόσον έχει θυλάσει, όλα αυτά συνδέονται με την έκθεση σε ιστρογόνα. όταν τα ιστρογόνα περιλαμβάνονται σε φάρμακα μπορεί να αυξήσουν αυτό το κίνδυνο και οι ενδοκρινικοί διαταράχτες εδώ, ε, όπως ας πούμε είναι η διεθυλστιλβιστρόλη, μπορεί να επηρεάσει ακριβώς ε, το, το, το στήθος και να δημιουργηθεί καρκίνος. Jesus λέει η ομιλήτρια. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι τα συνθετικά ιστρογόνα επίσης αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του στήθους, όπως το DDT, στην αρχή τη ζωή κάποιου, ή το βυσφενόλι, ή βισφενολι σε οποιαδήποτε φάση τη ανάπτυξη του οργανισμού. Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα πιθανολογούμενης ή σίγουρης παρενέργειας των ενδοκρινικών διαταραχών. Φυσικά δεν περιοριζόμαστε εδώ στον καρκίνο, έτσι. Αυτό προέρχεται από τον πίνακα 2 της εκθεσής μας, αυτό που βλέπετε. Και έχουμε έξι από αυτές τις ενώσεις. Έχουμε όργανοφωσφάτες, ε, φυτοφάρμακα, ε, προϊόντα προστασίας των φυτών που επηρεάζουν την ομοιόσταση, ομοιόσταση των, του θυροειδούς. Ε, μόλι, παραδείγματος χάρη που μπορεί να πάρει κανείς μια έγκυος αρχές εγκυμοσύνης της και που αλλάζει την ε, ορχική λειτουργία, τη λειτουργία των όρχεων, από ό,τι έχει αποδειχθεί. Μία άλλη ερώτηση ανησυχητική είναι η έκθεσή μας σε μείγματα. Συχνά ε, εδώ έχουμε συσσωρευτικές επιπτώσεις. Ε, εκτιθέμαθα σε ενώσει και σε μείγματα. Ε, Συχνά, ας πούμε, ε, υπάρχει πολλαπλασιαστική απάντηση στην έκθεση αυτή. Ε, Παραδείγματος χάρη στη βυσφινολένη, που χαμηλώνει τα επίπεδα τεστοστερόνης κατά 50%. Αν η BPA ανακατευτεί με άλλες ενώσεις, μάλιστα 8 ενώσεις ας πούμε, η δόση για να χαμηλώσει την τεστοτερόνη διαιρείται δια 10. Δηλαδή 10 φορές χαμηλότερη ε, δόση μπορεί να μειώσει εξίσου την τεστοστερόνη. Επίσης αυτή η έκθεση είναι, στην δυσφενόλη είναι πανταχού, παρόσα, πανταχού παρούσα στην, ε, στον ευρωπαϊκό πληθυσμό. παιδιά από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες τα εξετάσαμε για να δούμε τι ενδοκρινικούς διατάραχτες έχουν στο αίμα και στο, στα ουρά. Ε, 33 από τα 45, από τους 45 ενδοκρινικούς τα βρήκαμε σε πάνω από 90 παιδιά που ελέγξαμε. Επομένως δεν έχουμε απλώς καθολική έκθεση, αλλά μια και πολλές από αυτές τις ενώσεις ε, σε αυτές τις ενώσεις εκτιθέμεθα συνεχώς, συχνά. Για ορισμένους από αυτούς τους ενδοκρινικούς διαταράχτες, όταν έχουμε στοιχεία έκθεσης, να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το κόστος υγείας. Το κόστος είναι εξωφρενικό, δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οι περισσότερες, ε, τα περισσότερα προβλήματα έχουν να κάνουν με την απώλεια IQ και την, το, τα προβλήματα στον εγκέφαλο. Γιατί έχουμε τεράστιες νευρολογικές αρρώστιες. Ε, γιατί τα προβλήματα ε, διαγνώνονται ε, νωρί στη ζωή του παιδιού. Ενώ για τι μεταβολικέ αρρώστιε, α πούμε, τα καταλαβαίνουμε πολύ αργότερα και είναι πολύ πιο δύσκολο ας πούμε, να τα συνδέσουμε με κάποιε αρρώστιε. Επίση, για τι νευρολογικές νευρολογικέ αρρώστιε, θα ήθελα να σα πω ότι συνδέονται πολύ περισσότερο από άλλε με φυτοφάρμακα. Τώρα θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μου. Ε, ε, Ευχαριστώ. Τώρα θα συζητήσουμε για την συνέπεια των επιστημονικών δεδομένων που ακούσαμε με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προστασία και τι νομοθεσία έχει εγκριθεί μέχρι τώρα. Σε τι βαθμό λοιπόν υπάρχει συνέπεια ανάμεσα στην επιστήμη και τους ευρωπαϊκούς στόχους και τη ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πάνω από 20.000 χημικά έχουν επισημανθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει εντοπιστεί η βλάβη που μπορούν, μπορεί να προκαλέσουν Και έχουμε τον κανονισμό, ο οποίος διέπει όλα αυτά τα χημικά και τα ταξινομεί. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές. Μία βασική αρχή είναι ότι κατηγορίες που απειλούν πολύ σημαντικά την ανθρώπινη υγεία έχουν εντοπιστεί και ταξινομηθεί. Υπάρχουν λοιπόν τα χημικά που ανήκουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες και απαιτούν κάποια σημαντική και ιδιαίτερη διαχείριση. Πρόκειται για τα καρκινογόνα, τα μεταλλοξιογόνα, ε, ουσίες ε, μεταξύ άλλων και ενδοκρινικοί διαταραχτές. Οι διάφορες κατηγορίες ορίζονται στον κανονισμό REACH με συγκεκριμένε κατηγορίε. Υπάρχει επίση και οδηγία CLP, η οποία δεν αναφέρεται σε όλε τι βλάβε ούτε περιλαμβάνει κάποιον ορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών. Υπάρχουν διάφορα κείμενα επίση, όπω είναι το 7ο πρόγραμμα δράση για το περιβάλλον, που λέει ότι στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 2020 τα χημικά να παράγονται και να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Και λέει επίσης ότι το 2020 διάφορε ουσίε, μεταξύ άλλων αυτές που, έχουν, που προκαλούν διαταραχές ενδοκρινικές, θα πρέπει να έχουν περιοριστεί. Το 2008 στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα πλαίσιο για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες αναφέρεται στην αρχή της πρόληψης και την ελεγχιστοποίηση της έκθεσης των ανθρώπων σε τέτοιες ουσίες. Μπορεί κανείς να εντοπίσει και πέντε προσθήκες που θα πέτρεπαν όντως την ελεγχιστοποίηση της έκθεσης στους ενδοκρινικού διαταράκτε. Πρώτα απ' όλα, ένα σαφή ορισμός βάσει των επιστημονικών δεδομένων. Δεύτερον, ένα έγγραφο καθοδηγητικό που να εντοπίσει τις διάφορες ουσίες που εμπίπτουν στον ορισμό. Με κάποιες προϋποθέσεις, αλγορίθμους κτλ. Τρίτον, δοκιμές που θα πρέπει να υποστεί μια ουσία για να δούμε αν ανταποκρίνεται ή όχι στον ορισμό. Να κρυθεί κατά πόσο η ουσία ε, διαταράσει την ορμονική λειτουργία του οργανισμού ή τι βλάβες προκαλεί στον οργανισμό ή σε ένα πληθυσμό. Τέσσερα. Δεν φτάνει να υπάρχουν αυτές οι δοκιμές. Πρέπει να ε, ζητηθεί από μια επιχείρηση να γίνουν αυτές οι δοκιμές σε μια ουσία που χρησιμοποιεί. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και η λογική της διαχείρισης κινδύνου, δηλαδή ποια είναι η ελάχιστη έκθεση η οποία πρέπει να επιτρέπεται. Αν αυτές οι πέντε προϋποθέσεις υπάρχουν, τότε όντως θα πετύχουμε την ελάχιστη έκθεση των ανθρώπων σε ενδοκρινικούς διαταράκτες. Τώρα στην αξιολόγηση που κάναμε διαπιστώσαμε ότι το τομέα όπου μπορεί να πετύχουμε περισσότερο αυτή την ελάχιστη έκθεση είναι εκείνος των βιοκτώνων. Προϊόντα για το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο. Όσον αφορά την φυτοπροστασία, από το 2018 υπάρχει ο ορισμός επιστημονικών κριτηρίων για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Υπάρχουν δηλαδή οργανισμοί όπως ε, η ΕΦΣΑ που έχουν ε, ετοιμάσει, εκπονήσει έγγραφα τα οποία βασίζονται σε αυτούς τους ορισμούς. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα προϊόντα φυτοπροστασίας μπορούν να αναγνωριστούν ως δοκρινικοί διαταράκτες και τότε δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε αυτά οι άνθρωποι, εκτός αν πρόκειται για πραγματικά μια πυρολάχιστη έκθεση. Ο στόχος αυτός όμως για να εφαρμοστεί πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δοκιμές για να παίρνουν την άδεια τα προϊόντα αυτά πριν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν φυτοφάρμακα. Κάτι το οποίο όμως δεν συμβαίνει από ό,τι είδαμε εμείς. Δεν συμβαίνει κυρίως για τα βιοκτώνα. Γιατί οι δοκιμές δεν γίνονται πάντοτε, καλύπτουν όλες τις μορφές ενδοκρινικής διαταραχής. Επίσης, οι αιτήσει δεν ξέρω αν φτάνουν για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα αν ένα βιοκτόνο είναι βλαβερό ή όχι. Και πρέπει να δούμε και αυτός ο οποίος αποφασίζει πώς θα αντιμετωπίσει την αξιολόγηση ενός νέου βιοκτόνου. Αν τώρα περάσουμε σε έναν, άλλο, σε έναν άλλο τομέα ανθρώπινη έκθεση που είναι τα χημικά περιλαμβάνοντα τον στον κανονισμό REACH, εδώ η κατάσταση είναι διαφορετική και λιγότερο αποτελεσματική. Η Γαλλική Υπηρεσία έχει κάνει την αξιολόγηση και προσπάθησε να δει κατά πόσο τα συστατικά περιλαμβάνοντα στο REACH καλύπτονται από κανονισμό ή όχι δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμπεράσματα γιατί οι πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της, που συνοδεύουν δηλαδή το προϊόν, δεν ήταν αρκετές. Έπειτα, οι απαιτήσει για τις δοκιμές δεν έχουν έναν νομικά αξιόπιστο ορισμό και η λογική, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι τόσο σαφής όπως η παρουσία των ενδοκρινικών διαταρακτών στα φυτοφάρμακα. Κάποιες ουσίες δεν φαίνεται αν έχουν απευθείας συνέπειες ή όχι εφόσον χρησιμοποιούνται. Έχουμε τώρα 13 ενδοκρινικούς διαταράχτες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Και παρόλο που ο κανονισμό REACH δεν μας βοηθάει σε αυτό αρκετά, παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να εντοπίσει 13 χημικά που θεωρούνται ότι έχουν επικίνδυνη δράση ενδοκρινικής διαταραχής αλλά δεν πρόκειται μόνο βέβαια για 13, υπάρχουν πολύ περισσότερα και αυτό το βλέπω από τις διάφορες επιστημονικές μελέτες. Θα έπρεπε να μπουν όλα σε αυτές οι ουσίες το 2020 στον κατάλογο REACH. <clears throat> τα, καλλιντι... τα καλλιντικά τώρα. Οι γυναίκες βέβαια κυρίως εκτίθενται σε αυτά. Υπάρχουν διάφορες οικογένειες τέτοιων προϊόντων που έχουν εγκαταλειφθεί επειδή φαίνεται ότι είναι καρκινογόνα. Όμως, όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράχτες, μερικοί που δεν επιτρέπονται στα φυτοφάρμακα, δεν απαγορεύονται εδώ στα καλλιντικά. Γιατί εδώ ε, κρίνονται κατά περίπτωση. Σε άλλους, σε άλλες ε, συμφωνίες που πρόκειται για την ε, προστασία των εργαζομένων. Επίσης η αντιμετώπιση είναι συνολική. Τώρα, εκεί που υπάρχει συνένεση, νομίζω από όλες τις πλευρές, είναι όσον αφορά τον επιστημονικό ορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών και τις επιπτώσεις τους, τη βλάβη τους στην υγεία. Δεν μπορούμε να πούμε πόσοι είναι ακριβώς αυτοί οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, πόσοι κυκλοφορούν. Αλλά αυτό ισχύει και για τα καρκινογόνα, για παράδειγμα τις καρκινογόνες ουσίες. Το ίδιο ούτε εδώ ξέρουμε πώς ακριβώς είναι τα καρκινογενή προϊόντα, οι ουσίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Όμως ρυθμίζονται και υπάρχει νομικός ορισμός και βρίσκονται και σε τρεις κατηγορίες. Εξελίσσεται η γνώση μας όσον αφορά τις βλάβες που δημιουργούν οι διάφορες αυτές ουσίες, οπότε καλό θα ήταν να έχουμε οριζόντιο κανονισμό για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και να τους βάλουμε σε κατηγορίες. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελεγχιστοποίηση της έκθεσης των ανθρώπων και του περιβάλλοντος είναι κάτι που επιστημονικά δικαιολογείται απόλυτα. Ζούμε σε μια περιοχή του κόσμου όπου τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τα θέματα της υγείας ε, ρυθμίζονται με κανονισμούς. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης συνήθως. Η φυτοπροστασία, τα βιοκτώνα, είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να ρυθμιστούν για να περιοριστεί η έκθεση. Η κατάσταση μπορεί να μην είναι τέλεια, γιατί είπαμε ότι οι απαιτήσει για τις δοκιμές για τα τεστ είναι περιορισμένες, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με τα χημικά REACH που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές, εκεί υπάρχουν απαιτήσει για ε, δοκιμές ώστε τελικά να μην έχουμε εγγυήσει για ελαχιστοποίηση της έκθεσης για όλους τους ενδοκρινικούς διαταράκτες που γνωρίζουμε. Το 2020 θα θέλαμε να συμπεριληφθούν όλες αυτές οι ουσίες στο REACH. Εμείς στην έκθεσή μας κάνουμε προτάσεις για τον οριζόντιο ορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών που να ισχύει για όλους τους τομείς, τους τομείς και πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης στους ενδοκριτικούς διαταράκτες ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτος, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε που μας ε, τα εξηγήσατε όλα αυτά. Σε εμά που δεν είμαστε ειδικοί στα χημικά και πραγματικά είναι μια δύσκολη υπόθεση και δύσκολο να τα χωνέψουμε όλα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάντως. Και τώρα θα ήθελα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την έκθεση αυτή που αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Να συμπληρώσω την παρουσίασή σας με κάτι που ουσιαστικά αναφέρεται στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της ανακοίνωσης του Νοεμβρίου 2018. Μία ανακοίνωση που ουσιαστικά ακολουθεί τη δέσμευση της Επιτροπής από κοινού κράτη-μέλη για την ανάπτυξη κριτηρίων για την αντιμετώπιση των ενδοκρινικών διαταρακτών στα φυτοφάρματα κτλ. Προβλέπονται πολλές διαφορετικές δράσεις. Το ξεκίνημα όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας της νομοθεσίας σε όλα τα κράτη-μέλη αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ελέγξουμε αν καταρχήν η ευρωπαϊκή νομοθεσία καλύπτει τον βασικό στόχο προστασίας, αν υπάρχουν αδυναμίες, κενά που πρέπει να καλυφθούν όσον αφορά τη βελτίωση της συνοχής αυτής της νομοθεσίας που αφορά τους ενδοκρινικούς διακταράκτες και αυτό σε όλους τους τομείς, τομείς και όσον αφορά τους ελέγχους πώς ορίζονται οι έλεγχοι, ποια είναι τα μέτρα για την διαχείριση του κινδυνού που απορρέει από την χρήση των ενδοκρινικών διαταρακτών. Μία σειρά μέτρων που έχουν ενσωματωθεί σε ένα νοδικό χάρτη που έχει γνωστοποιηθεί σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να μπορέσουν να αντιδράσουν. Επίσης, μία διαβούλευση έχει οργανωθεί Πολλές φορές συνεχίζουμε να παρατηρούμε έλλειψη ενημέρωσης και ελέγχων. Έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση στα πλαίσια του Οριζοντά 2020 καθώς και κονδύλια για την έρευνα που αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει επίσης την οργάνωση ενός ετήσιου φόρουμ με σκοπό τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών, επιστημονική φορείς, δημόσιες αρχές, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό να υπάρξει μια ευρεία συζήτηση για την ε, ευρύτερη αντιμετώπιση των ενδοκρινικών διαταρακτών. Τέλος, μια ιστοσελίδα με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες και που υπάρχουν σήμερα σε πολλούς διαφορετικούς ε, ιστότοπους ε, της ΕΦΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις Χημικές Ουσίες κτλ. Αυτές είναι οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και Πρόεδρος. Συνάδελφοι, Ξέρετε ότι πρόκειται για την παρακολούθηση των αναφορών που έχουμε λάβει. 19 συνολικά που αφορούν το θέμα αυτό. 13 παραμένουν ανοιχτές, θα παραμείνουν εξάλλου ανοιχτές μέχρι να υπάρξουν απαντήσεις από τις εθνικές αρχές είτε έως ότου να καλύψει το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις συγκεκριμένες αυτές αναφορές έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει η ε, νεότερη αξιολόγηση. Παραμένουν λοιπόν οι 13 αυτές αναφορές ανοιχτές και συνεχίζουμε την παρακολούθηση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σημειώσαμε όλα αυτά που μας παρουσιάσατε και εσείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από μέρους των εμπειρογνωμόνων. Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι. Συμφωνείτε όλοι. Η κυρία Ριβαζή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, ερευνητές μας και να πω ότι κάτι με εκπλήσει όταν κοιτάω τον ε, κατάλογο δράσεών σας. Εξηγήσατε τα θέματα που αφορούν ε, τα φυτοφάρμακα. Υπάρχει ορισμός, υπάρχουν δοκιμές, αξιολόγηση κινδύνου κτλ. Η ερώτηση μου είναι εξή. Πώς είναι δυνατόν ό,τι έχει σχέση με τα καλλιντικά, με τις ε, ουσίες ε, και τα πρόσθετα στα τρόφιμα που μας αφορούν άμεσα. Πρόκειται για το νερό, για τα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις και μπορείτε να μας πείτε παραδείγματο χάρη γιατί δεν υπάρχει οριζόντιος ορισμός και γιατί δεν υπάρχουν ε, τεστ, δοκιμές υποχρεωτικά. Εάν ε, δεν ξέρουμε αν η συγκεκριμένη ενεργή ουσία, δραστική ουσία είναι ενδοκρινικός διαταράκτης ή όχι, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε κατώτατα όρια από τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, που δεν ξέρουμε αν ένας ενδοκρινικός διαταράκτης μπορεί ακόμα και σε πάρα πολύ μικρές ποσότητες να προκαλέσει συγκεκριμένες βλάβες. Αν δεν ξέρουμε, παραδείγματο χάρη, ποια είναι η κατώτατη περιεκτικότητα. Επίσης, κοιτώ εδώ τη μέθοδο αξιολόγησης της ΕΦΣΑ για τη λεγόμενη δράση στα μείγματα. Και αναρωτιέμαι αν, ενώ έχουμε τον κατάλογο τουλάχιστον 50 ουσιών που χαρακτηρίζονται ως ενδοκρινικοί διαταγράκτες, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την δράση όλων αυτών. Μας μιλήσατε για τις επιπτώσεις στην υγεία, τους καρκίνους παραδείγματο χάρη, ναι, ε, επί της ε, γονιμότητας. Σήμερα υπάρχει επιδημία, αύξηση του αριθμού των ε, περιπτώσεων καρκίνων και όσον αφορά τη γονιμότητα, όσον αφορά την ε, ευφυΐα. Μα τελικά τι μας λέτε. Δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα-βήμα και με προσοχή. Εδώ υπάρχει επίγουσα κατάσταση. Είναι όπως με το κλίμα. Όλα αυτά που λέτε αφορούν το κληροδότημά μας στην επόμενη θητεία, στο επόμενο κοινοβούλιο περιμένουμε να μας απαντήσετε. Όλα αυτά μας φοβίζουν, μας ανησυχούν και σας ευχαριστώ πολύ για την δράση σας. Υπάρχει η έκθεση αυτή και βεβαίως μας αφορά το θέμα αυτό όχι μόνο εμάς αλλά και πολλές άλλες επιτροπές. Περνάμε στην 879 αναφορά που αφορά τον ε, άνθρακα και την μόλυνση πηγών. Όχι, δεν είναι εδώ ο αναφέρον, αλλά ο εκπρόσωπός του. Έχετε πέντε λεπτά. Dobrý deň prajem a ďakujem za možnosť vystúpenia na tomto výbore v súvislosti s petíciou, ktorá pojednáva práve o spore kúpeľov a banskej spoločnosti ťažiacej uhlie. Mám iba 5 minút, prejdem preto priamo k veci. Obe tieto spoločnosti, ktoré vidíte... Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο και μπορούμε να πάρουμε το λόγο για την μόλυνση αυτών των πηγών. Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στην εταιρεία αυτή που βρίσκεται στην περιοχή της Πριέβιτσα. Πρόκειται για μια με κόκκινο χρώμα περιοχή στο χάρτη και βεβαίως θα αναφερθούμε εδώ στους εργαζόμενους αυτής της ιδιωτικής επιχείρησης. Το γεγονό ότι αυτή η επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει τι δραστηριότητέ μέχρι το 2023 διαπιστώνουμε ότι τα ιαματικά ε, ύδατα ε, ε, επηρεάζονται από εξορυκτικές δραστηριότητες του λιγνίτη. Και βεβαίως διαπιστώνουμε την ίδια ώρα ότι με κίτρινο χρώμα βλέπετε τις υπόλοιπες εξορρυκτικές δραστηριότητες. Είναι σημαντικό ότι η εταιρεία αυτή που έχει δραστηριότητες και σε, πολλές άλλες, σε πολλά άλλα ορυχεία έχει μολύνει συγκεκριμένες πηγές ιαματικών ε, λουτρών και μάλιστα είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι το μισό ορυχείο ουσιαστικά προστατεύεται. Στην πράξη όμως βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να διαχωρίσει κανείς την προστατευόμενη περιοχή των ιαματικών λουτρών από την άλλη περιοχή η οποία μολύνεται. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να αναφερθώ σε τρία σημεία θα πρέπει να σταματήσει άμεσα αυτή η εξορρυκτική δραστηριότητα του άνθρακα. Και με τον τρόπο αυτό βλέπουμε ότι η περιεκτικότητα σε εχνοστοιχεία αυτών των ιαματικών ε, υδάτων και λουτρών μειώνεται και πλέον η ποιότητά τους δεν είναι αυτή η οποία αναφέρεται. Είναι επίσης σημαντικό ότι 12 περίπου χιλιόμετρα συγγνώμη, 3 χιλιόμετρα διορθώνει ο μιλητής από το επίκεντρο αυτής της μόλυνσης παρατηρείται η μείωση της ποιότητας, η επιδείνωση της ποιότητας όλων αυτών των πηγών των ιαματικών λουτρών. Μπορούμε επίσης να αναφερθούμε επίσης και στην θερμοκρασία αυτών των πηγών. Και θα σας δώσω και κάποια στοιχεία. Βλέπετε σε αυτό το πίνακα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν την ποιότητα των ε, υδάτων, ένας μέσος όρος τη δεκαετία του 60, του 70 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε λοιπόν και αυτό είναι ένας πολύ συγκεκριμένος πίνακας με παραδείγματα για την ε, μόλυνση των υδάτων αυτών αλλά και για την ροή τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισκεφτεί την ε, περιοχή, έχει ζητήσει την εξέταση αυτής της υπόθεσης θα πρέπει να σταματήσουν αυτές οι δραστηριότητες και αυτό για την περιοχή είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες αυτής της συγκεκριμένης περιφέρειας. Έχουμε κάνει μία μελέτη όσον αφορά τα ιαματικά αυτά λουτρά και την ποιότητα των ε, υδάτων. Και γι' αυτό και προετοιμάσαμε αυτή τη συγκεκριμένη αναφορά. Ελπίζουμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα ασχοληθούν με την υπόθεση αυτή ότι θα υπάρξει μια ουδέτερη αξιολόγηση και όχι η αξιολόγηση η εντελώς μεροληπτική που έγινε από μέρους της ε, επιχείρησης. Προσβλέπουμε, αν θέλετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνομιλήσει κατευθείαν με το Υπουργείο Υγείας της ε, Σλοβακίας έτσι ώστε στο μέλλον να σταματήσει αυτή η δραστηριότητα. Τέλος, θα ήθελα να κάνω μια έκκληση προς ε, όλους σας. Χρειάζεται πολύ αυστηρή προειδοποίηση προς τις ε, αρχές της χώρας μας, προς την κυβέρνηση, έτσι ώστε πραγματικά να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν και πριν είναι πολύ αργά η κατάσταση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος ή εκπρόσωπος της Επιτροπής είναι εδώ. Μαρκέτα Μπένου βαλεύομαι, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Θέλω να ευχαριστήσω τον αναφέροντα για την αναφορά του. για την επέκταση, παράταση μάλλον της διάρκειας αυτού του εργοστασίου εξόριξης λιγνίτη, το οποίο είναι επίμαχο η μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου ε, είναι κάτι που θα κάνουν οι σλοβακικές αρχές. Δεν υπάρχει ενωσιακή νομοθεσία ειδική για την προστασία των ιαματικών πηγών. αλλά η οδηγία πλαίσιο για το νερό απαιτεί από τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν όλα τα project και να αρνηθούν την αδειοδότηση για μεμονωμένα project εάν το project μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση των υπόγειων υδάτων ή να επιδεινώσει την κατάσταση των υπογείων υδάτων ή ε, υδάτων του εδάφους. Οι σλοβακικές αρχές θα πρέπει να αποφασίσουν τι επίπτωση θα έχει το project με βάση την οδηγία και να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με την ενωσιακή οδηγία για το νερό, για τις επιδοτήσεις που δίνονται. Η Κομισιόν είναι σε επαφή με τη Σλοβακική Δημοκρατία για το εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας του Νοβάκη, το οποίο το αξιολογούμε για να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα με τους ενωσιακούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Δεν ξέρουμε να έχουν δοθεί δημόσιες επιχορηγήσεις στους υπαλλήλους που δουλεύουν στο εργοστάσιο Λιγνίτη. Ε, η περιοχή του Μπρέβιτσα είναι μία από τις περιοχές που επέλεξε η περιοχή ε, για, και τις θεωρεί περιοχές σε μετάβαση ε, είναι μια πρωτοβουλία που βάσει τη οποία η Κομισιόν δίνει τεχνική βοήθεια στην Σλοβακία για να αναπτύξει μια στρατηγική μετάβαση και ένα σχέδιο δράση. Ε, η στρατηγική και το σχέδιο δράση ε, θα είναι έτοιμο μέσα στο πρώτο μισό του 19 και ελπίζω και η στρατηγική και το σχέδιο δράση θα λαμβάνουν υπόψη τα προβλήματα που ανέφερα αναφέροντας. Η ανάπτυξη διαφόρων ιαματικών πηγών και λουτρών, σπα, θα είναι προφανώς εποφελής για το μέλλον μιας περιοχής που βασιζόταν στην εξόριξη, στα ορυχεία δηλαδή. Η παράταση της διάρκειας της λειτουργίας του ορυχείου δεν έχει αδειοδοτηθεί ακόμα, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Ε, και με βάση τη Σλοβακική νομοθεσία πρέπει να γίνουν μια σειρά από μελέτε. Δεν είναι αρμοδιότητα τη Κομισιόν να παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία. Επομένω, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει παράβαση τη ενωσιακή νομοθεσία σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε πολλού ευρωβουλευτέ σήμερα, αλλά όσοι είναι, μιλάνε πολύ. Ο Κρίστιαν Πρέντα. Ε, ευτυχώ που είμαι εδώ λοιπόν, αφού είμαι τόσο δραστήριο. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση της αναφορά αυτής. Μας ε, ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό. Άκουσα την εκπρόσωπο της Κομισιόν να λέει ότι δεν υπάρχει παράβαση. οι συνάδελφοι της Επιτροπής Περιβάλλοντος, τι άποψη έχουν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ενημερώθηκαν για αυτό το θέμα οι συνάδελφοι της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Νομίζω πως ναι. Τι είπαν αυτοί. Κατά αυτούς η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σωστή, είναι αποδεκτή. Εμείς το ΕΛΚΑ θα θέλαμε να διευκρινιστούν όλα αυτά τα θέματα η περιβαλλοντική σκοπιά του θέματος. Η κυρία Βαλέρα νομίζω είναι η αρμόδια για αυτά τα θέματα. Σωστό δεν είναι αυτό που λέω. Και επειδή θα επανεκλεγεί, κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει το έργο της. Είναι σημαντικό λοιπόν το δούμε αυτό το θέμα, γιατί έχουμε και άλλες παρόμοιες αναφορές. Αυτά ευχαριστώ. Κυρία Τρεμπέσιους, ευχαριστώ. Επίτροπε, είπε η ομιλήτρια. Ε, ευχαριστώ την κυρία Βίξτρομ, Ευχαριστώ την Κομισιόν. Εκ μέρους του ECR θα ήθελα να υποστηρίξω στεναρά την αναφορά. Πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Αυτό λέει η ομάδα μου. Η Επιτροπή ΠΕΤΗ θα πρέπει να ξεκινήσει μια γραπτή διαδικασία ε, με τα συνυπεύθυνα σλοβακικά υπουργεία για να διευκρινιστούν τα θέματα τα οποία αναφέρει η αναφορά. Επίσης, προτείνουμε να παραπέμψουμε αυτή την αναφορά στην Επιτροπή περιβάλλοντο, όπω είπατε και εσεί, κύριε Πρέντα, για να γνωμοδοτήσει και αυτή η Επιτροπή. Και η Κομισιόν θα θέλαμε, να τη πούμε, να συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την κατάσταση. Το συστήνουμε θερμά. Πολύ ωραία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Ε, κυρία Χάουτα, ε, συγγνώμη. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Έχουμε, είναι τεράστια η καταστροφή και για το κλίμα και για το περιβάλλον από τα ορυχεία, από την εξωτερική βιομηχανία. Την απάντηση παίρνουμε πάντως από την ε, Επιτροπή. Ε, και απλώς εμείς κάνουμε μια διαμαρτυρία post-mortem, μετά θανάτιο. Καλό θα ήταν να έχουμε κάπου την αίσθηση ότι υπάρχει επικοινωνία με τις αρχές, όχι για να κάνουμε μόνο νεκροψία, αλλά για να προλάβουμε και το κακό. Έτσι, και προφανώς, προφανέστατα πρέπει να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, αλίμονο. Εννοείται, λέει η Πρόεδρος. Επομένως, πρώτον, στείλαμε αυτό το θέμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ενημερωτικά, για να ενημερωθούν για το πρόβλημα, για το τι συμβαίνει. Θέλω να ζητήσω μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, να δούμε ποια είναι η άποψή της. Επομένως, το σημειώνουμε αυτό και θα το κάνουμε. Επίσης, θα πρέπει να ετοιμάσουμε μια επιστολή προς τις Σλοβακικές Αρχές, να τις ενημερώσουμε για τις ανησυχίες μας και για το τι διεμήφθη εδώ στην Επιτροπή μας και επίσης ξέρουμε ότι η αδειοδότηση είναι καθοδόν, έτσι. Επομένως είμαστε στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Παράλληλα θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γραπτή επικαιροποίηση, γραπτή ενημέρωση. Γιατί πρέπει να μπει αυτή στο φάκελο του θέματος αυτού. Πέρα από την προφορική ενημέρωση θέλουμε και μία γραπτή, έτσι. Και ενημερωτικά Θέλω να σας πω ότι το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος ε, Νοβάκη θα κλείσει το 2021 και είναι υπεύθυνο για το 7% όλων των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στη χώρα. Μιλάμε τώρα για τεράστια νούμερα, έτσι. Από ένα εργοστάσιο μόνο. Επομένως, ε, είναι σοβαρή ιστορία αυτή, έτσι, σοβαρό θέμα. Ευχαριστώ. Εμίλια, θες ξανά το λόγο? Όχι you Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ που μα το θέσατε αυτό το θέμα υπόψη, που ταξιδέψατε από τη χώρα σα. Ε, κάποια μέρα θα σας θεωρήσουν ήρωα της Ευρώπη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Περνάμε... τις απόψεις αυτές που εκφράστηκαν και άκουσα εδώ. Περνάμε στην επόμενη αναφορά. Πρόκειται για την Δανέζικη εταιρεία για την προστασία της ε, φύσης που εναντιώνεται στην κατασκευή ενός φράχτη κατά μήκος των συνόρων Δανίας-Γερμανίας ε, για την παρεμπόδιση της μετανάστευσης των αγριόχειρων. Δεν είναι εδώ να φέρω. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως ναι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που δίνετε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγώ δουλεύω στο τμήμα που ασχολείται με τις ε, ζωονόσους στη Γενική Διάθεση ΣΑΝΤΕ. Η αναφορά αφορά ε, ένα επίμεχο θέμα, ε, ένα φράχτη που θέλει να χτίσει η δανέζικη κυβέρνηση στα σύνορα με τη Γερμανία για να προβλέψει τη μετατόπιση των αγριόχειρων και την διείσδυση μιας αρρώστιας που είναι η αφρικανική πανόλη των χείρων που είναι αρκετά σοβαρή και που μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότατες βλάβες ε, εντός της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τα μέτρα, αυτά, αυτό το μέτρο του δηλαδή φράχτη, ε, με γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ, της Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Και δεν έχει καταλήξει ότι αυτού του είδους τα, οι φράχτες είναι αποτελεσματικοί πραγματικά δεν, δεν έχουμε καταλήξει σε κάτι τέτοιο. Η διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχειρων, εξ, η σωστή διαχείριση, ε, ε, απαιτεί ένα σύνολο μέτρων. Έχουμε εμπειρία και από το Βέλγιο και από την Τσεχία όταν, εμφανίστηκαν, ε, όταν εμφανίστηκε αυτή η αρρώστια στους αγριόχειρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ποτέ δεν στήριξε τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες στηρίζει περισσότερο μέτρα περιορισμού του πληθυσμού, πολύ στοχευμένα όμως. Καταλήγοντας, η Κομισιόν οργάνωσε μια υπουργική ε, συνεδρίαση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, ακριβώς για να δούμε τα όρια αρμοδιοτήτων ε, και τις σχέσεις ε, στον τομέα αυτό. Μια στρατηγική μακροπρόθεσμη συμφωνήθηκε υπάρχουν συστάσεις που τονίζουν ότι οποιοδήποτε μέτρο που θα ληφθεί για τον περιορισμό της Αφρικανικής Παντολής των Χείρων και του πληθυσμού των αγριόχειρων θα πρέπει να είναι συμβατό και με την περιβαλλοντική νομοθεσία και με την κτηνιατρική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά θα πρέπει να επαληθεύσουμε και επιστημονικά αυτά τα μέτρα και τεχνικά σε ό,τι αφορά την επίπτωση και στην πανίδα αλλά και στο περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, ε, κυρία Οκέν. Θα μιλήσω δανέζικα. Μια που το θέμα αυτό το παρακολουθούμε στη Δανία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντησή της που ήταν ξεκάθαρη. Όλοι στη Δανία γνωρίζουμε ότι αυτός ο φράχτης που εμποδίζει την μετακίνηση των αγριόχειρων δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Είπαν όλοι των χείρων φυσικά και είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σωστά. Για παράδειγμα, η μεταφορείς αγριόχειρων είναι και αυτοί υπεύθυνοι. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται η ασθένεια αυτή με τη μεταφορά κρέατος γίνεται ή από τραυματισμένα ζώα. Οπότε αυτός ο φράχτης δεν πρόκειται να μας προστατέψει. Ε, το άλλο που πιστεύω είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση της Δανίας πρέπει να παρέμβουν. Γιατί το φράχτη αυτό τον βλέπουμε, μπορούμε να τον δούμε από τη θάλασσα. Φτάνει μέχρι τη θάλασσα εξάλλου και εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία ανάμεσα στη Δανία και τη Γερμανία. Θα λέγαμε δηλαδή ότι ξαφνικά θέλουμε να γίνουμε σύνορα ανάμεσα στη Δανία και τη Γερμανία. Οπότε πρόκειται για ένα φράχτη που έχει φτιαχτεί και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, σε δάση για παράδειγμα, ενώ πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον. Οπότε ναι, σας ευχαριστώ πολύ που υπογραμμίσετε ότι η Δανία δεν έχει τηρήσει την περιβαλλοντική νομοθεσία. Είναι το ελάχιστο. Όταν έχουμε περιοχές Natura 2000 πρέπει να προστατεύουμε αυτές τις περιοχές. Και αν δεν έγινε μελέτη στη Δανία είναι ότι ακριβώς δεν αναφέρθηκε ότι ο φράχτης αυτός μπορεί να βλάπτει το περιβάλλον, ενώ το κάνει, είναι προφανές. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια εγγύηση να πούμε ότι η Δανία δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της και να δούμε τι γίνεται με την προστασία του περιβάλλοντος εκεί. Και έπειτα είναι και μια πρόκληση κατά των Γερμανών συναδέρφων, γιατί στις διασυνοριακέ περιοχές ο κόσμος ανησυχεί τόσο από την πλευρά της Δανία, όσο και από τη ε, Γερμανίας για τη δημιουργία αυτού του φράχτη ανάμεσα στις δύο χώρες. Ενώ πρόκειται για ζώνες ε, προστασίας διασυνοριακές, για τη συνεργασία, μετανάστευση κτλ. Θα πρέπει να βρεθεί Μάλλον οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν άλλο τρόπο τελικά για να περάσουν από τη μία χώρα στην άλλη, εκεί που υπάρχει αυτός ο φράχτης, ενώ τα αγριογούρουνα κυκλοφορούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω απέναντι στη Δανία, να επιμείνει να έχει μια απάντηση ή ακόμα και να ξεκινήσει μια δικαστική διαδικασία επί παραβάση τη στιγμή που υπάρχει μια τόσο κατάφορη παράβαση από πλευράς της Δανίας των περιοχών Natura 2000. Δεν έχει κανένα νόημα αλλιώ να υπάρχουν τέτοιες περιοχές Natura 2000. Έπειτα σπαταλώνται 4 εκατομμύρια κορώνες που όμως βλάπτουν την φύση και το περιβάλλον. Ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει λοιπόν στην κυβέρνηση της Δανίας και να ζητήσει να σταματήσει η οικοδόμηση αυτού του τείχους και μια για πάντα να δούμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικό ένα τέτοιο μέτρο, αλλά και κυρίω τι επιπτώσει έχει στο περιβάλλον. Γιατί τι νόημα έχει να έχουμε νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντο, αν ξεφεύγουμε κάθε φορά με τέτοιο τρόπο. Ναι, νομίζω ότι θα ήθελα να γραφτεί στα πρακτικά ότι στηρίζω την δήλωση της ε, κυρία Σόκεν και πιστεύω ότι οι αριθμοί που έχουμε ενδεχομένως δεν είναι και η τελική. Έχουμε κάποια στοιχεία που αφορούν την πανόλη των χείρων και θα πρέπει να δούμε και όλες οι άλλες ε, ουσίες και όλες οι άλλες πηγές, ε, αν θέλετε, πώς αξιολογούνται. Δεν υπάρχει σήμερα πάντως προστασία, όχι μόνο κατά αυτής της ασθένειας, αλλά και άλλων. Και η εξάπλωσή της ε, είναι ανησυχητική. Ο τρόπος πάντως αντιμετώπισης και τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν είναι καλά ούτε για το περιβάλλον, αλλά ούτε και για την προστασία της ανθρώπινης ε, υγείας, ούτε και βεβαίως της υγείας των ζώων. Κάπως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξαναδεί λίγο την στρατηγική της. Είμαστε, αν θέλετε, περήφανοι στην Ευρώπη γιατί μπορούμε ενδεχομένως να βάλουμε σύνορα όταν πρέπει, αλλά εδώ δεν βλέπω να είμαστε αποτελεσματικοί καθόλου. Ναι, πρόκειται. Αυτή είναι η ιστορική στιγμή όταν ο κύριος Γιάρ και η κυρία Όκεν συμφωνούν πραγματικά ιστορική στιγμή. Μπράβο. Ξέρετε, εγώ κάθομαι εδώ Συνήθω γράφω και τώρα αυτή τη φορά σταμάτησα και κοιτάω. Είναι πραγματικά μια συμβολική στιγμή αυτή. Αν συμφωνούν, σίγουρα θα κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή. Και τώρα κάτι πιο σοβαρό, αλλά βέβαια είναι και αυτό συμβολικό, γιατί στην Ευρώπη ε, δεν ε, έχουμε έρθει εδώ για να φτιάχνουμε φράχτες και τείχους, γέφυρες να φτιάχνουμε. Οπότε είναι και πολύ πιο συμβολική η αξία από ό,τι φανταζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό πολιτικά να πούμε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να φτιάχνουμε φράχτες, να παίρνουμε τέτοια μέτρα στην Ευρώπη. Να υπογραμμίσω επίσης κάτι που κάνουμε πάντα. Να μετράμε την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα. Υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση. Ο Πίτερ Γιάρ το είπε πάρα πολύ καλά ότι τελικά ο φράχτης δεν εμποδίζει τους αγριόχειρους να περάσουν και αν πρόκειται να έχουμε μια πανδημία με, από την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων δεν θα τη σταματήσει κανένας φράχτης γιατί δυστυχώς πάνε πιο γρήγορα. Οπότε κρατάμε ανοιχτή την αναφορά αυτή και ζητάμε από την κυβέρνηση της Δανίας να σταματήσει τον φράχτη αυτό, να μην συνεχίσει και θα πούμε, θα υπογραμμίσουμε και θα τονίσουμε για άλλη μια φορά αυτά που λέμε για την αναγκαιότητα και την αναλλαγικότητα, αλλά θα αναφερθούμε επίσης και στην συμβολική αξία. Και δεν πρόκειται εδώ πέρα μόνο για τη Δανία και τη Γερμανία, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Συμφωνείτε? Καλώς. Και συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι η αναφορά 513 για την μη αναγνώριση οικογενειών ΛΟΑΔΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται επίσης και για την οδηγία 1081 που δεν επιτρέπουν χωρίς θεώρηση πρόσβαση στην ε, Πολωνία συζύγου Πολωνού. Λοιπόν, για την πρώτη υπόθεση δεν είναι εδώ η αναφέρουσα, ούτε και για τη δεύτερη, ούτε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως είναι εδώ. Οπότε παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα αρχίσω με την πρώτη αναφορά του 2016, την 513. Θέτει διάφορα ζητήματα. Αλλά θα ασχοληθώ πιο πολύ με την μη αναγνώριση του ονόματος του παιδιού της αναφέρουσας και η συνάδελφος θα αναφερθεί στα άλλα θέματα. Ένα λοιπόν από τα ζητήματα που θέτει η είναι το γεγονό ότι οι ελληνικές αρχέ αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν το όνομα, το διπλό όνομα του παιδιού, το οποίο γεννήθηκε ε, από ένα ζευγάρι ή δύο φίλου. Αγγλίδας και Ελληνίδας. Οι Ισπανικέ αρχέ δέχτηκαν ε, το διπλό όνομα, χρησιμοποίησαν και τα ονόματα για των δύο γονιών, ενώ οι ελληνικέ αρχέ δεν αναγνωρίζουν το διπλό όνομα. και δέχονται το όνομα ενός από τους δύο γονείς. Η Επιτροπή εξήγησε την προηγούμενη φορά, τον Ιούλιο του 2018, ποιο είναι το νομικό καθεστώς, αλλά θα ε, συνοψίσω ότι βάσει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εάν το όνομα έχει καθοριστεί νομικά σε μια άλλη χώρα μέλος, τότε η χώρα μέλος υπηκότητας δεν μπορεί να αρνηθεί την αναγνώριση αυτού του ονόματος γιατί εμποδίζει την άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάστασης νοσηπικού. Διακόπτη η πρόεδρος. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να σας ενοχλούν οι συνάδελφοι, οπότε Ζητάω από τους προηγούμενους αναφέροντες που έχουν να κάνουν την προηγούμενη αναφορά να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους εκτός αιθούσης παρακαλώ. Ορίστε, σας ακούμε. Μάλιστα έλεγα λοιπόν ότι ένα τέτοιο εμπόδιο στην άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας μπορεί να αιτιολογηθεί αλλά κάτω από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Μπορεί να δικαιολογηθεί αν υπάρχουν αντικειμενικές, αντικειμενικοί λόγοι ή αντιτίθεται σε εθνικές διατάξεις ή αν κάτι που έχει να κάνει με τη ε, δημόσια πολιτική πρέπει να γίνεται αποδεκτό και από τις δύο χώρες και όχι μόνο μερός. Οι αντιρρήσεις σχετικά με την πολιτική αυτή θα μπορούσε να είναι μόνο απειλή για την κοινωνία μέτρα επίσης που περιορίζουν αυτή την ελευθερία ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής δικαιολογούνται μόνο με στόχους χωρών ε, μελών εφόσον τα, οι στόχοι των χωρών μελών δεν μπορούν να υλοποιηθούν με άλλα μέτρα λιγότερο δραστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως σας είπαμε τον Ιούλιο, έγραψα σε ελληνικές αρχές και οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν έτοιμα στο, στην ενωτάτη αρχή όσον την υπεύθυνη για τα ονόματα των παιδιών και το έτοιμα αυτό εκρεμεί ακόμα οπότε δεν μπορούμε να απαντήσουμε τις αναφέρουσης. Επίσης, ενημερωθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα από τις ελληνικές αρχές ότι το Συμβούλιο Επικρατείας τελικά ε, ενέκρινε τη γνωμοδότηση 201 το 2018 και έδωσαν και πληροφορίες ελληνικές αρχές για τα βήματα τα οποία σκοπεύουν να αναλάβουν μετά από την άρνηση αναγνώρισης του ονόματος. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τώρα την απάντηση των ελληνικών αρχών αλλά η προκαταρτική ανάλυση που κάναμε δείχνει ότι οι ελληνικές αρχές είναι διατεθειμένες να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα και να διορθώσουν την άρνηση αποδοχής του ονόματος. Και θα δώσω το λόγο τώρα στη συνάδελφο που θα απαντήσει στα άλλα θέματα που θέτει η αναφέρουσα. Ευχαριστώ Ρούτ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να προσθέσω μόνο ότι ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αναφέρουσα ε, να φροντίσουν και για την αναγνώριση των εγγράφων του παιδιού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε διαδικασία προβληματισμού και θεωρεί ότι ο Εθνικός Νόμος για την Αναγνώριση της υπηκότητας είναι αρμοδιότητα της κάθε χώρας ε, μέλους και βέβαια πρέπει να συνάδει και με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και έχουν υπάρξει διάφορες δικαστικές αποφάσεις για ονόματα. όταν πρόκειται για γάμο ας πούμε, που έχει λάβει χώρα σε μια άλλη χώρα πρέπει να αναγνωρίζεται βάσει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των συνθήκων. Ένα από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες ΛΟΑΔΕ για να αναγνωριστεί το παιδί τους όσο τέτοιο έχει να κάνει, όπως είπαμε, με την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται καμία άλλη νομοθετική δράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα έχει αναλύσει κατά πόσο προτάσεις για νομοθεσία έχουν πιθανότητα να καταλήξουν σε κάτι. Σε αυτό το στάδιο βλέπουμε ότι ούτε στο Σεβούλιο ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υπάρξει πλειοψηφία για μια τέτοια νομοθετική δράση. Εξού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει για την αναγνώριση να υπάρξει νομοθετική πρόταση. Όπως έλεγε και η συνάδελφος, υπάρχει η Εθνική Νομοθεσία που αναγνωρίζει τα δικαιώματα του πολίτη και υπάρχει και η νομολογία βέβαια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Κανείς δεν βλέπω να θέλει το λόγο. Α, η κυρία Βόρντο. Συγγνώμη, δεν σας είχα δει πριν. Mm. Παρακαλώ, κύριε Ward. Ναι, δεν είμαι τακτικό μέλος της Επιτροπής Αναφορών, αλλά πάντα όταν είμαι παρούσα χαίρομαι ιδιαίτερα για τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτής της αναφοράς και σαν Βρετανίδα Και όπως ξέρετε, επειδή δεν συνέβη το Brexit ε, την προηγούμενη εβδομάδα, μπορεί να μην συμβεί και ποτέ, υπάρχει βρετανικό ενδιαφέρον για αυτήν την ε, αναφορά. Η διαδικασία του Brexit έχει περιπλέξει πάρα πολύ τα πράγματα σε περιπτώσεις σαν αυτήν. Ξέρω ότι η αναφορά αυτή αφορά ένα ζευγάρι η Ελληνίδα που έχει υποβάλει την αναφορά αναφέρεται στις ελληνικές αρχές, την αναγνώριση από μέρους των ελληνικών αρχών και την ίδια ώρα θεωρώ ότι θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να αναβαθμίσουν το επίπεδο των απαιτήσεών τους και να μπορέσουν να είναι εξίσου απαιτητικά σε σχέση με τέτοιες ε, υποθέσεις και ελπίζω αυτή η αναφορά να παραμείνει ε, μία αναφορά που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Και θεωρώ, λέει η Πρόεδρος, ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι για όλα όσα κάναμε μέχρι τώρα. Το 2016 ήδη, αλλά και το 2018, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό, ζητήσαμε γνωμοδότηση, Συζητήσαμε το 2018 τον Ιούλιο το θέμα εδώ στην Επιτροπή. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Κατά την άποψή μου, αυτή η αναφορά, αυτές οι αναφορές πρέπει να κλείσουν. Ξέρετε γιατί. Γιατί εμείς ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το έχουμε κάνει. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να συνηγορήσει υπέρ του να παραμείνουν ανοιχτέ, είναι η διαδικασία του Brexit. Ας τις αφήσουμε λοιπόν ανοιχτές μέχρι την επόμενη ε, συνεδρίαση της επόμενης Επιτραπής ε, Αναφορών στο επόμενο Κοινοβούλιο για το λόγο αυτό. Επαναλαμβάνω ε, διαδικαστικά, αν κοιτάξει κανείς τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητές μας, έχουμε εξαντλήσει κάθε δυνατότητα. Παρ' όλα αυτά, Ας την αφήσουμε ανοιχτή. Έχουν νομίζω σταλεί όλες οι πληροφορίες. Μάλιστα πήραμε πολύ εμπεριστατωμένη ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές. Υπήρχε και το θέμα του ονόματος, αν δηλαδή κάποιος που έχει παντρευτεί μπορεί να κρατήσει το όνομά του και έχουμε σήμερα αναλύσει όλες αυτές τις διαφορετικές περιπτώσεις και διατάξεις. Περιμένουμε και την γραπτή αναφορά. Μπορούμε να στείλουμε μια επιστολή στην Επιτροπή ζητώντας περισσότερες διευκρινήσεις και πιστεύω ότι καλό θα ήταν να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βοηθούν πολύ στην καταπολέμηση αυτών των απαράδεκτων ε, συμπεριφορών. Και εμείς σαν θεσμικά όργανα θα πρέπει να έχουμε παραδειγματική συμπεριφορά. Ιδιαίτερα όταν ε, πρόκειται για περιπτώσεις παιδιών. Πιστεύω λοιπόν να σταλεί, ότι θα πρέπει να σταλεί μία επιστολή. Και αυτό πολύ γρήγορα τις επόμενες ημέρες. Συμφωνείτε όλοι? Εντάξει. Νομίζω λοιπόν ότι μας αξίζει ένα ωραίο βραδινό δείπνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.